Uh, um, Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο δεύτερο τμήμα των τριών ακροάσεων που έχουμε όσον αφορά την Cambridge Analytica και την προστασία των δεδομένων και τις συνέπειες που είχαμε μέχρι τώρα. Είναι η δεύτερη ακροασή μας λοιπόν αυτή η οποία λαμβάνει η χώρα εκ μέρους της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αλλά επίσης και εκ μέρους των Επιτροπών Ήτρε, ΑΦΚΟ και Γιούρι. Όλες οι επιτροπές αυτές εκπροσωπούνται εδώ. Οι άλλοι πρόεδροι των άλλων επιτροπών θα έρθουν αργότερα, δεν ξέρω ακριβώς ποιοι θα έρθουν. Ο αντιπρόεδρος της Τζούρι, η κυρία Μάντι Ντελβός της ναι, σε ξέρω Μάντι ότι είσαι εδώ, για τους άλλους λέω ότι δεν ξέρω αν είναι εδώ. Αύκο, η κυρία Χούμπνερ κανονικά, θα έρθει φαντάζομαι, και η κυρία Ήτρε από τον κύριο Ρούμπικ είναι σημαντικό όλες οι επιτροπές να συμμετέχουν στην ακρόαση αυτή. Και θα έχουμε μαζί μας, νομίζω, και την Αντιπρόεδρο της ΙΜΚΟ και την Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού. Κάλτ, σωστά. Αυτέ είναι οι δυνατότητε τέλο πάντων που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, 4 Ιουνίου είχαμε την πρώτη μα ακρόαση. Και επιτρέψτε μου να σα διαβάσω εδώ πέρα κάποια εισαγωγικά σχόλια πριν μπούμε στην ουσία της ακρόασής μας. Είναι σημαντικό όμως γιατί στην πρώτη ακρόαση είχαμε μια καρποφόρα συνάντηση μαζί τους και με μια συμπαθητική μορφή. Θα ακολουθήσουμε το ίδιο. Λοιπόν, καλωσορίζω όλους τους προσκεκλημένους μας ε, εδώ που συνήθως δεν είναι εδώ. Ελπίζω ότι θα προσθεθούν και άλλα μέλη των διάφορων επιτροπών. Είναι Δευτέρα και ίσως ταξιδεύουν ακόμα, αλλά θα έρθουν. Λοιπόν, μετά την απόφαση της Διάσκεψης των Πρόεδρων στις 12 Απριλίου 2018 και τη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Τσούκεμπεργκ σε επίπεδο διάσκεψης των Προέδρων, αποφασίσαμε το Κοινοβούλιο δηλαδή αποφάσισε να οργανώσει τρεις σε βάθος κοινοβουλευτικές ακροάσεις των επιτροπών μας με ε, συνομιλητές μας από την Cambridge Analytica όσον αφορά το σκάδαλο του Facebook. Στόχος είναι να μπούμε περισσότερο σε βάθος, να δούμε τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε από όλη αυτή την ε, ιστορία και τι μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχετε ίσως ακούσει ότι ε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε τους καταλληλότερους ομιλητές τη ακροάσεις αυτές. Είναι πολύ σημαντικό πράγματι να ακούσουμε από αυτού που είναι υπεύθυνοι από τα διάφορα τμήματα που έχουν θέσει ευθύνης στο facebook και αλλού. Και σήμερα ελπίζω ότι όντως θα ακούσουμε τους προσκεκλημένους μας. Το δεύτερο τμήμα θα επικεντρωθεί κυρίως στις συνέπειες, δηλαδή ποιες είναι οι επιπτώσεις από την προστασία δεδομένων στο ιδιωτικό βία, βίο, τις διάφορες διαδικασίες, τι γίνεται με τις ψηφιακές πλατφόρμες, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την ε, θέση στην αγορά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Το τρίτο τμήμα της ακρόασης αυτή που θα είναι στις 2 Ιουλίου θα ακούσουμε διάφορους επιτρόπους για τις λύσεις, τις πολιτικές και άλλες λύσεις προκειμένου να μην επαναληφθούν ε, τέτοια φαινόμενα όπως είχαμε. Ε, κυρία Σάμπερκ θα είναι εδώ που είναι διευθύνων σύμβουλο ή κάποιος που θα την αντικαταστήσει. Αρχίζουμε λοιπόν με την σημερινή μας ακρόαση. Και έχουμε σημαντικούς ομιλητές. Προηγουμένως να σας επενθυμίσω τους κανόνες που έχουμε αποφασίσει για τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Την προηγούμενη φορά ήταν πολύ επιτυχής αυτή η μορφή της ακρόασης, οπότε να τηρήσετε τους κανόνες. Πριν από τη συνάντηση, οι πολιτικές ομάδες αποφάσισαν να υποβάλουν ερωτήσεις, 15 ερωτήσεις η κάθε ομάδα βάσει του συστήματος DONT. Όλα λοιπόν βασίζονται σε αυτό το κανόνα, DONT. Μετά από κάθε ερώτηση ζητούμε από τους προσκεκλημένους μας να δώσουν απάντηση. Μετά τις παρουσιάσεις του πάνελ θα δώσω το λόγο στους προέδρους των εμπλεκόμενων εδώ κοινοβουλευτικών επιτροπών και μετά θα καθορίσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ο καθένας που βρίσκεται στον κατάλογο ομιλητών αλλά και οι πρόεδροι μια ερώτηση μπορούν να υποβάλουν προς έναν από το πάνελ. Οπότε πρέπει να πείτε σε ποιον απευθύνεται την ερώτησή σας. Ένα λεπτό. Και ο προσκεκλημένος από το πάνελ πρέπει να απαντήσει σε δύο λεπτά. Πρέπει να τηρηθεί αυτός ο χρόνος, για τελείως θα σας κόβω. Αν τώρα δεν είναι παρόν αυτός που έχει ζητήσει το λόγο από τους ευρωβουλευτές, θα περάσουμε στον επόμενο αυτόματα. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχω τίποτα άλλο να ρωτήσω μπορούμε να περάσουμε στους ομιλητές. Ωραία. Περνάμε λοιπόν στους προσκεκλημένους μας. Ανδρέα και είναι πρώτα απ' όλα πρόεδρος EDB από την Αυστρία. Και στη συνέχεια ο κύριος ΔΕ που είναι επικεφαλής του Personal Data IO και ο κύριος Σάτερφιλντ επίσης που είναι πρόεδρος για την ε, πολιτική προστασία του βίου στο Facebook. Θα αρχίσουμε λοιπόν με το πρώτο αυτό τμήμα που είναι οι ερωτήσεις, ο πρόεδρος. Α, πρώτα θα δώσω το λόγο Α, λάθος λέει ο πρόεδρος. Όχι, όχι, όχι. Πρώτα, θα ζητήσω από τους προέδρους και αντιπροέδρους των άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών να μας πούνε αν θέλουν κάτι να πούνε. Μάντι, έχεις κάτι να πεις. Ευχαριστώ, Κλοντ. Εδώ εκπροσωπώ την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή μας εξετάζει ζητήματα τα οποία έχουν ε, να κάνουν με τα θέματα της νομολογίας, ε, της ε, φαρμαζόμενης νομοθεσίας, ποιος είναι υπεύθυνο για να πάρει προσφυγές και να τις εξετάσει κτλ. Τι γίνεται με την εθνική δικαιοσύνη και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες, δεδομένα φορολογικά, αλλά και πνευματική διοκτησία. Εκ μέρους λοιπόν της Επιτροπής Γιούρι και εγώ σας καλωσορίζω εδώ όλους τους εμπειρογνώμονες. Ελπίζω και εγώ ότι θα έχουμε μια ανοιχτή και επικοδομητική συζήτηση όσον αφορά θέματα δικαιοδοσίας για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την περίπτωση και τι δυνατότητες έχουμε για να μην επαναληφθούν τα ίδια στο μέλλον. Τίποτα άλλο. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως. Πάντα είσαστε σύντομοι, Μάντι. Ευχαριστώ πολύ και την Τζούρι που ήρθε. Αν έρθουν και άλλοι πρόεδροι των άλλων επιτροπών, φαντάζομαι θα θέλουν και αυτοί να πάρουν τον λόγο. Ωραία, αρχίζουμε την ακρόαση. Και ξεκινούμε με τον πρώτο μιλητή, Ανδρέα Γελινέκε, πρόεδρος EDPB Αυστρία. Δέκα λεπτά παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, <clears throat> αγαπητέ πρόεδρε αξιότιμες ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτές, ο GDPR άρχισε προ λίγων ημερών να ισχύει και με τον κανονισμό GDPR το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων δημιουργήθηκε από, συντίθεται από τις Εθνικές Αρχές, των EDPS και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υπόθεση Cambridge Analytica Facebook ελέγχεται από τον ICO στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι εκεί έχει την έδρα του η Cambridge Analytica. Μέχρι να αρχίσει να ισχύει ο GDPR, ο ICO θα ήταν η leading authority. Θα συνέτασε την απόφαση και θα την διαβίβαζε στις άλλες συναρμόδιες αρχές. Εν τέλει θα μπορούσαν να επιβληθούν πρόστιμα μέχρι 4% του κύκλου εργασιών της επιχειρήσεως. Επειδή όμως η υπόθεση έγινε, προέκυψε πριν από την, ε, πριν από την ε, εμφάνιση της υποθέσεως, ο ICO είναι όχι μόνο leading authority αλλά και investigating authority, δηλαδή η αρχή που διεξάγει τις έρευνες και θα συντάξει μελέτη. Ο ICO όμως μας ενημερώνει διαρκώς, δηλαδή τις άλλες εθνικές αρχές προστασία δεδομένων και εμεί συνεργαζόμαστε στενά μαζί του. Οι έρευνε έχουν διεξαχθεί και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν Ιούνιο ή Ιούλιο. Ένα από τα κέρια θέματα του GDPR είναι και η λογοδοσία και οι επιχειρήσεις και εν προκειμένου η Facebook πρέπει να αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τους κανόνες και την λογοδοσία. Ο κανονισμός, ο GDPR δηλαδή, δίνει πάλι στα υποκείμενά του, δηλαδή στους πολίτες, τον έλεγχο των δεδομένων τους. Έχουμε πλέον ισχυρότερη εργαλειοθήκη από ό,τι πριν. Η προστασία δεδομένων δεν έπεσε στις 25 Μαΐου από τον ουρανό. Η οδηγία που έχει προηγηθεί του κανονισμού ισχύει ήδη από μια 20 ετία και είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών και πελατών τους εάν συμμορφώνονται με τον GDPR, διότι αυτό είναι και επιχείρημα πωλήσεων, αλλά είναι και αναγκαίο σύμφωνα με τον νόμο. Εάν μια επιχείρηση επενδύει στην προστασία δεδομένων και αναλαμβάνει τις ευθύνες η ελεγκτική αρχή ως ελεγκτική αρχή, δεν χρειάζεται μετά να επενδύσει η επιχείρηση σε εκστρατείες ε, για να ζητήσει γνώμη από το κοινό, κάτι το οποίο δεν αρκεί. Ο EDPP, όπως δηλαδή το Συμβούλιο ε, Προστασίας Δεδομένων, έχει ήδη στα χέρια του 30 υποθέσεις. Θα τις διερευνήσουμε πολύ προσεκτικά σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού GDPR και η ηγετική δηλαδή αρχή προστασίας δεδομένων και οι υπόλοιπε που συνεργάζονται. Η υπόθεση Facebook Cambridge Analytica είναι η κορυφή του παγόβουνου, όπως έχουν πει και άλλοι προηγουμένως. Αυτό που είναι το ανησυχητικό, ωστόσο, είναι οι αποκαλύψεις που γίνονται πρώτα και μετά το Facebook δέχεται ότι έχει διαβιβάσει αλλού τα δεδομένα των χρηστών του. Και κάθε φορά που γίνεται κάποια αποκάλυψη υπάρχει και ε, μία ε, αποδοχή και δεν ξέρουμε ακριβώς πόσες είναι οι ψηφίδες του Μωσαϊκού. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων ενισχύει τα άτομα και τα δικαιώματά τους. Δεν είναι το ζήτημα αν καταχράται κανείς δεδομένα τα οποία δεν θα έπρεπε να έχει καν στη διάθεσή του. Εάν δεν έχει δώσει ο χρήστης ελεύθερα την συνένεσή του, την συγκατάθεσή του, δεν μπορείτε να συλλέγετε τα δεδομένα. Όπως διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, εβδομάδα το Wall Street Journal, τη μεγάλη αυτή εφημερίδα, διεξάγει σχετική έρευνα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, διότι είναι η πρώτη φορά που αρχίζουν τώρα και οι Αμερικανοί να αντιλαμβάνονται τη σημασία της χρήσης των δεδομένων τους. Υπάρχει ενδιαφέρον από πολλά μέρη του κόσμου σε ό,τι αφορά τον κανονισμό GDPR. Και η Ευρώπη παίζει ρόλο πρωτοπόρου. Επίσης, οι αμερικανικές επιχειρήσεις όχι μόνο προσπαθούν να συμμορφωθούν, όπως άλλωστε οφείλουν, ακολουθούν και η συνειδητοποίηση είναι όλο και μεγαλύτερη για την ανάγκη προστασία των δεδομένων και όπως βλέπετε και από Αμερικανούς πολίτες. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Να έρθουμε τώρα στον Paul DeHay, Πρόεδρο της Personal Data I.O. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Εγώ άρχισα να ανακατεύομαι με την ε, Cambridge Analytica εδώ και καιρό. Το Δεκέμβριο του 2015 διάβασα ένα άρθρο του Harry Davis στην Guardian που εξηγούσε ότι η Βρετανική εταιρεία είχε ασχοληθεί με πολιτικά δεδομένα εκατοντάδων ε, χιλιάδων ε, Αμερικανών και αμέσως άρχισα να σκέφτομαι πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια τέτοια συζήτηση για την προστασία δεδομένων από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ε, μετά άρχισα να ερευνώ τη δικιά μου περίπτωση και συγκέντρωσα πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ήταν πάρα πολύ ανησυχητικά. Φάνηκε μάλιστα ότι ήταν ακόμα περισσότερο σημαντικά εξαιτία των όσων διαβάζαμε για το Brexit και για τις αμερικανικές εκλογές. Ή μάλλον για να το πω αλλιώ, γιατί ήταν ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης κάλυπταν ε, όλα αυτά. Πήγα σε δημοσιογράφους λοιπόν με τα στοιχεία μου και έτσι σιγά σιγά ξαναφανίζονται τα στοιχεία για την Cambridge Analytica. Σε κάθε στάδιο όμως, μέσα σε λίγα χρόνια, διαπίστωσα ότι άρχισαν και στο Facebook να μην αισθάνονται πολύ καλά γιατί φαινόταν ότι αυτά που έλεγα ήταν αλήθεια. Και όλα πηγαίνανε καλά για αυτού μέχρι το Μάρτιο του 2018. Κάποιοι συνόψαν την περίοδο αυτή λέγοντα ότι το Facebook είναι απλώ ό,τι και η Cambridge Analytica, απλώ έχει καλύτερε προσωπικέ σχέσει. Και ίσω να ισχύει κάτι τέτοιο, μια που αυτά που προσπάθησε να κάνει η Cambridge Analytica τα κάνει και το Facebook έτσι κι αλλιώς. Είναι μια ρουτίνα για αυτούς, μόνο που μέχρι τώρα δεν είχαν βγει και πολύ στο φως. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, αυτού του είδους την κάλυψη από τον τύπο θα την έλεγα top-down transparency, από πάνω προς τα κάτω διαφάνεια δηλαδή. Ε, στην πραγματικότητα δηλαδή δεν συμμετέχει καθόλου ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Τι θα ήταν το αντίστοιχο. Ε, θα έλεγα ότι ο στόχος είναι να αντιλαμβάνονται τα άτομα πώς διαμορφώνεται το δικό τους οικοσύστημα πληροφόρησης. Γιατί να μην έχουν απάντηση στις ερωτήσεις τους λοιπόν οι χρήστες. Στην περίπτωση της Cambridge Analytica ακούσαμε τον καθηγητή David Carroll στην πρώτη μας ε, ακρόαση όσον αφορά το δικό του subject access request. Και εγώ άρχισα να προσπαθώ να αναλύσω τα πράγματα όσον αφορά την δικιά μου αίτηση πρόσβαση από το Δεκέμβριο του 2016 και ζήτησα από το Facebook να μπορέσω να έχω πρόσβαση στα custom audiences και στα pixel δεδομένα μου. Από την πλευρά των διαφημιστών, λοιπόν, βλέπουμε ότι μπορούν αυτοί να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία όσων έχουν το email τους ή το τηλέφωνό τους. Μετά από επιμονή το Facebook δημιούργησε ένα εργαλείο ώστε να μπορούν να κάνουν το αντίθετο. Δηλαδή οι χρήστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στου διαφημιστέ που χρησιμοποιούν το δεδομένο του. Και εντελώ αυθαίρετα όμω το Facebook στη συνέχεια περιόρισε σε δύο μήνες αυτή τη δυνατότητα. Οπότε ήταν άχρηστο και δεν μπορούσε κανεί αναδρομικά να ψάξει να βρει τι είχαν γίνει τα στοιχεία του στις προηγούμενε εκλογέ. Όμω, παρόλα αυτά διαπίστωσαν πολλοί χρήστε πω εκατοντάδε διαφημιστέ χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους παριστάνοντας ότι έχουν τη συνένεσή τους. Έγιναν λοιπόν πολλά άρθρα όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες όταν αρχίσαμε να συζητάμε για το Facebook. Τώρα όσον αφορά τα δεδομένα Pixel. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει κατάλογος με σελίδες εκτός στο Facebook από διαφορετικές δηλαδή πηγές που χρησιμοποιούμε στο Facebook. Και θα μπορούσε να ήταν ενδιαφέρον και αναδρομικά να το κοιτάξει κανείς για να δει τελικά τι ισχύει, ποια είναι η δυναμική. 18 μήνες αργότερα όμως δεν έχω πάρει ακόμα αυτό το κατάλογο. Οι προσπάθειες αυτές όμως οδήγησαν σε ερωτήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο τα σχόλια του κυρίου Τζίκεμπερκ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Κογκρέσο. Όμως οι απαντήσεις που έδωσαν όλοι αυτοί οι αρμόδιοι είναι αντιφατικές σε σχέση με τις απαντήσεις που είχα πάρει εγώ νωρίτερα. Και αυτό υπογραμμίστηκε από τον ε, κύριο Μπλούκεμπερκ στο Κογκρέσο. Γιατί τελικά η Facebook αυτό που κάνει είναι ότι παρουσιάζει ένα καινούργιο εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιήσει στο μέλλον, με σαφή όμω στοιχεία. Και το οποίο εργαλείο χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν πιστεύουμε ότι θα είναι αποτελεσματικός. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα εμφανιστεί σαν σε θελοντική βάση και όχι σαν κάτι υποχρεωτικό, όπως θα έπρεπε και όπως έλεγε Facebook πριν από 18 μήνες. Αξίζει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε μέσα από το Privacy Shield. Στη θεωρία τουλάχιστον είχα την ευκαιρία να τα όλα αυτά σε ένα εξάρτητο τρίτο μέρος που ονομάζεται τραστή. Όμως μετά από λίγο η Facebook μίλησε στην τραστή και βρήκε τρόπο να απαλλαγεί από τις κατηγορίες μου. Οπότε έπρεπε να περάσω σε κάτι άλλο, σε μια επιτροπή στην Ιρλανδική Προστασία Δεδομένων. Χωρίς όμως δυστυχώς να πετύχω τίποτα πώς να σας το πω, κατά τη γνώμη μου και δεν είναι μόνο δικιά μου γνώμη, η Irish Data Protection, η υπεύθυνη δηλαδή, είναι εκείνοι η οποία επέτρεψαν στην Facebook να κάνει αυτά που κάνει και να παρακάμπτει την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Συνεπώς, η Facebook είναι πραγματικά η Cambridge Analytica, αλλά με καλύτερες δημόσιες σχέσεις, με καλύτερους δικηγόρους και καλύτερο lobbying. Και είναι κρίμα. Εδώ δεν ψάχνω τη διαφάνεια για τη διαφάνεια. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να καταλάβω καλύτερα πώς λειτουργούν τα συστήματα αυτά και να μάθω και τους άλλους να καταλαβαίνουν καλύτερα τα ψηφιακά. Και βρήκα μια δουλειά στην Personal Data I.O., μη κερδοσκοπική, και προσπαθώ να βοηθήσω. Περιμένω βέβαια να έρθουν και άλλες γραπτές μαρτυρίες στην Επιτροπή σας. Τέλος, τα δεδομένα του Facebook είναι πολύ σημαντικά για να εντοπίσει κανείς και να λύσει τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Όμως δεν είναι η ίδια εταιρεία Facebook το κλειδί. Ο ίδιος ο Μάρκ Zuckerberg ζήτησε συγγνώμη και μας ζήτησε περισσότερη εμπιστοσύνη για να διορθώσει την κατάσταση. Όμως στην πραγματικότητα έτσι αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη εξουσία πάνω σε ένα οικοσύστημα πληροφοριών το οποίο όμως κάνει κακό αντί για καλό. Όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια θα μπορούσαν να συλλέγονται εκτός της Facebook και να υπάρχουν δικαιώματα για αυτά και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και άλλες υπηρεσίες που να προσφέρουν ένα αντιστάθμισμα στις εξουσίες και τη δύναμη της Facebook. Για παράδειγμα, το Facebook Pixel Data θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Θα μπορούσε επίσης να ανατεθεί σε δημοσιογράφους για να καταλάβουν και αυτοί καλύτερα πώς λειτουργούν τα πράγματα. Η καινοτομία αυτή όμως βρίσκει φραγμούς στην Facebook. Η Facebook θέλει να δώσει επιλεκτικά πρόσβαση στα δεδομένα για να δημιουργήσει τον ε, περίγυρο πληροφορίες έτσι όπως θέλει και βάσει το δικό της στόχων. Οπότε τη μεταφορά αυτή της δύναμης των δεδομένων θα ήθελα να την εξετάσετε και αντί να γίνεται η ανακατανομή μέσω φόρων θα έπρεπε να καταλάβετε ότι πρόκειται για νέες ευκαιρίες για τη στάθμιση δυνάμεων και εξουσίας. Ο Μάρκ Τσούγκερμπερκ μας αρνείται την ευκαιρία αυτή και τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση, να μπορούν να μεταφέρονται τα δεδομένα. Και δεν διορθώνει το πρόβλημα για το οποίο είναι υπεύθυνο. Ε, εννοείται, επιμένει σε ένα παλιό μοντέλο το οποίο δεν θα έπρεπε να εμπιστευόμαστε, όπως κάνει και αυτός. Σας ευχαριστούμε πολύ και περνάμε απευθείας στον Steve Satterfield, ε, τον Διευθυντή για την ε, Πολιτική Ιδιωτικότητα και υπεύθυνο της ε, Διαφημιστικής Πολιτικής του Facebook. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Το όνομά μου είναι Steve Satterfield Είμαι διευθυντή τη πολιτική ιδιωτικότητα και διαφημίσεων του Facebook. Είμαι υπεύθυνο για τα θέματα ιδιωτικού βίου και προστασία δεδομένων σε ό,τι αφορά τι διαφημίσει στις σχετικές μας εφαρμογές και πλατφόρμες. Δουλεύουμε μάνατζερ και μηχανικούς για να δούμε τα προβλήματα ιδιωτικότητας και ε, προστασίας δεδομένων όταν προτείνουμε τα προϊόντα μας. Όταν σχεδιάζουμε προϊόντα μας θέλουμε ε, ο κόσμος των, ε, οι άνθρωποι τον κόσμο να διασυνδέονται με τους γνωστούς τους αλλά και με έναν τρόπο που να προστατεύει την ιδιωτικότητά τους, να μπορούν να συνδέονται με εφαρμογές και ιστότοπους που τους ενδιαφέρουν. Με σεβασμό της ιδιωτικότητας και των δεδομένων τώρα, έχουμε ένα συγκεκριμένο επεισόδιο για την πλατφόρμα του Facebook, παραβίαση των πολιτικών σχεδιασμού, όταν ο Αλεξάνδρ Κόγκαν μετέφερε πληροφορίες προς την Cambridge Analytica. Θα σα δείξω τι μέτρα αναλήφθηκαν για να βεβαιωθούμε ότι η υπόθεση Cambridge Analytica δεν θα ξανασυμβεί. Όμω θα ήθελα η συζήτηση αυτή κάπω να διευρυνθεί και να μιλήσουμε και για τι πολιτικέ σχετικά με την ειδικότητα και την προστασία δεδομένων τη Facebook και το πώ συμμορφωνόμαστε με την GDPR τον νέο κανονισμό. Επίση, τι παρανοήσει για τι πρακτικέ του Facebook ω τώρα σε σχέση με τι διαφημίσει και τη συλλογή δεδομένων. Πολλά από τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα αφορούν την εμπιστοσύνη. Η υπήρξε μια ε, διακοπή, μια διαταραχή της, της σχέσης εμπιστοσύνης ε, με την υπόθεση της Cambridge Analytica. Θέλουμε να υπάρχουν διαρκείς βελτιώσεις στα προϊόντα μας και τις εσωτερικές μας διαδικασίες. Θα μας χρειαστεί καιρό για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που τώρα προέκυψαν. και να στραφώ και στο αντικείμενο της σημερινή ακρόσης τώρα, την Cambridge Analytica, να ξεκινήσω λέγοντας ότι οι καλύτερες πληροφορίες που διαθέτουμε ε, καταδεικνύουν ότι καμία ε, ε, καθόλου ευρωπαϊκά δεδομένα δεν πέρασαν από τον Dr. Kogan προς την Cambridge Analytica. Αυτό βάσει συμβάσεων. Η εταιρεία του Dr. Αλλά αυτό το μα το είπε και η Cambridge Analytica και η μαρτυρία του, του Dr. Kogan και η δική μας η ανάλυση. Δεν είναι εύκολο βέβαια να το ε, διαπιστώσουμε οριστικά πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, η νομική έρευνα και οι σχετικοί υπεύθυνοι της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου εκδώσουν τις γνωμοδοτήσεις τους, τα πορίσματά τους. Ο αντίκτυπος όμως της υπόθεσης και με τις αναλύτικα στους Ευρωπαίους πολίτες είναι σημαντική, σημαντικός, παρόλο που είναι περιορισμένος. Και σίγουρα το πλήγμα ήταν στη σχέση εμπιστοσύνη. Τι κάνουμε λοιπόν από εδώ και μπρος. Το πρώτο είναι να δούμε τι έγινε το 2014 όταν αλλάξαμε τι πολιτικές μας για να είμαστε αυστηρότεροι με την τήρηση πληροφοριών και να ζητάμε συνένεση των χρηστών. Και επίσης να αναθεωρήσουμε μάλιστα με πολύ δραστηριό τρόπο το τι απαιτείται στα διάφορα πεδία δεδομένων. Τώρα πάμε πολύ μακρύτερα. Όποιο χρησιμοποιεί την εφαρμογή θα πρέπει να έχει μία ε, αποδοχή, να του ζητάτε δηλαδή συγκατάθεσή του για να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες του με τη διεύθυνση email και ούτω καθεξής. Και υπάρχει ολόκληρη ομάδα συνεργατών που ασχολείται με αυτό. Επίσης, μετά από τρεις μήνες μη χρήση της εφαρμογής, απαγορεύεται η πρόσβαση στις πληροφορίες. Τον Απρίλιο, στην αρχή του Newsfeed, δείχναμε ένα κατάλογο του τι εφαρμογές ε, μπορούσε κανείς να χρησιμοποιεί, ε, αλλά τώρα δίνουμε τη δυνατότητα να αποσύρει κανείς και την ε, έγκρισή του προς την κάθε εφαρμογή. Και επίσης ε, είναι πολύ λιγότερες οι εφαρμογές που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες τώρα σε σχέση με τις αλλαγές που είχαν γίνει το 2014. Όταν έχουμε υποψίες, διακόπτουμε την πρόσβαση μιας εφαρμογής και την απομακρύνουμε εντελώ μέχρι να ελεγχθούν τα προσωπικά δεδομένα όλων όσοι χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή. Όμω πριν κάνουμε αυτή την αλλαγή στην πλατφόρμα μα, χρειάστηκε μια διετία για να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές που προέκυπταν από την συμμόρφωση με το GDPR. Ήταν τεράστια προσπάθεια για το Facebook. Η ομάδα συνεργατών που συνεργάστηκε από όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας ήταν από τις μεγαλύτερες. Όλοι αντάλλαξαν την πολύτιμη εμπειρία τους και χρησιμοποίησαμε και τις γνώσεις εμπειρογνωμών και πολιτικών ενθυνόντων για το θέμα αυτό. Κάποια παραδείγματα του τι κάναμε ως τώρα. Απλουστεύσαμε τους ελέγχους, τις ρυθμίσεις. Δηλαδή, αντί να έχει κάνει 20 οθόνε στις ρυθμίσεις, τώρα μπορεί να έχει πρόσβαση από ένα σημείο και μόνο. Υπάρχει ένα νέο πόρταλ όπου μπορεί ο καθένας να σχέσει τα δικαιώματά του, να περάσει σε διορθώσεις, και επικαιροποιήσαμε και τη φορητότητα σε σχέση με τι ε, πληροφορίε που μπορεί κανεί να κατεβάσει. Όλα αυτά επίση είναι διαθέσιμα σε όλου ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Ε, επίση υπάρχει και η ε, λεγόμενη engagement flow, δηλαδή η συγκατάθεση που ζητάτε από όλου του Ευρωπαίου για να επιτρέψουν την πρόσβαση στι προσωπικέ του πληροφορίε, του προφίλ του ή την αναγνώριση μέσω του προσώπου. Και επίση τα δεδομένα τρίτων μερών που είναι ένα παράδειγμα για να δουν αν θέλουν να δώσουν τη συγκατάθεση του ή όχι. Μπορεί κανείς να πει όχι σε όλα αυτά και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Facebook. Επίσης οι όροι του Facebook αναθεωρήθηκαν και η σύμβαση χρήσης μας ε, απαιτεί τη συγκατάθεση του χρήστη πρωτού συνεχίσει να χρησιμοποιεί το προϊόν μας. Και αυτό είναι διαφορετικό από τη διαδικασία συγκατάθεση που περιέγραψα προηγουμένω. Εγώ ασχολούμαι με την προστασία δεδομένων και την ιδιωτικότητα και όλα αυτά δεν σταμάτησαν στις 25 Μαΐου. Ίσα ίσα ε, σχηματίσαμε μια ομάδα για το GDPR. Τώρα έχουμε δημιουργήσει μια κεντρική υπηρεσία που Αγγλία από διάφορε ομάδε του Facebook ανά τον κόσμο για να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε τα σχετικά διαφημιστικά προϊόντα στο μέλλον. Με περισσότερο έλεγχο και προστασία. Σκοπεύουμε λοιπόν να ε, μπορούμε να δούμε και το ιστορικό ε, τη χρήση ενό ε, συγκεκριμένου καταναλωτή. Δηλαδή να μπορεί κανεί να δει τι έχει γίνει από το Facebook από την αρχή και όταν κανεί να σταματήσει να χρησιμοποιεί το λογαριασμό του όλα αυτά να καταργούνται πλήρω. Έχουμε λοιπόν κάποιες γενικές γραμμές για το πώς θα λειτουργεί όλο αυτό, αλλά θέλουμε προηγουμένως να έχουμε και τις αντιδράσεις στον κόσμο, που τον κόσμο, για να δούμε πώς συγκεκριμένα θα σχεδιάσουμε το συγκεκριμένο εργαλείο. Κάποιες λεπτομέρειες για το πώς λειτουργούν ε, τα διαφημιστικά μας προϊόντα τώρα, εντός ολίγου. Τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε όμως πρώτα. Πρώτα απ' όλα για τι διαφημίσει. Να ξεκινήσω λέγοντά το σαφώ. Το δικό μα business model βασίζεται στι διαφημίσει. Νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερο τρόπο να πετύχουμε του στόχου μα. Οι διαφημίσει που βλέπει ο κόσμο στο Facebook σίγουρα είναι στοχευμένε. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για να μπορούμε να τι κάνουμε προσωποποιημένε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ε, ο κόσμο θέλει να βλέπει διαφημίσει που να τον αφορούν. Και ξέρουμε ότι οι διαφημίσει ε, διευκολύνουν τι επιχειρήσει να φτάσουν στου καταναλωτέ ε, και να πουλήσουν τα προϊόντα του. Οι διαφημίσει συνολικά ήταν πολύ σημαντικέ, ιδίω για τι μικρέ εταιρείε και μικρού προπολογισμού για να διαφημιστούν. Όμω η διαφήμιση και η ιδιωτικότητα δεν είναι αντικρουόμενα στοιχεία. Μπορούμε να δείξουμε στου διαφημιστέ κάποια στοιχεία χωρί να του πούμε ποιοι είστε ή να δώσουμε όλε τι πληροφορίε. σα. Όπω είπα λοιπόν προηγουμένω, ζητάμε τη ρητή συγκατάθεση πρωτού χρησιμοποιήσουμε δεδομένα τρίτων μερών για τι διαφημίσει. και έχουμε και ένα εργαλείο που λέγεται προτιμήσει διαφημίσεων και επιτρέπει στου χρήστε να δουν ποια είναι τα ενδιαφέροντα ε, που του αφορούν περισσότερο και όπου θα θέλανε να λαμβάνουν διαφημίσει. Επίση, μπορεί κανεί να μην δει καθόλου διαφημίσει ε, στο Facebook ή να κρύψει τι ε, διαφημίσει ενό ε, διαφημιστή μελλοντικά πλήρω. Επίση, για το πώ το Facebook επεξεργάζεται τα λεγόμενα παράλληλα προφίλ όταν κάποιος δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Για να είμαι σαφής, δεν δημιουργεί προφίλ για κόσμο χωρίς προφίλ στο Facebook. Το Facebook. Θέλουμε οι διαφημίσει να είναι πιο, σχέδιο, πιο σκόπιμες και πιο ε, ενδιαφέρουσε για τον κόσμο που το χρησιμοποιεί το Facebook και τα διαφημιστικά εργαλεία να είναι πιο αποτελεσματικά για το business model του Facebook επίση και πολλέ εταιρείε προτείνουν τέτοιου είδου υπηρεσίε ούτω ή άλλω. Αλλά όταν χρησιμοποιεί κανεί μια εφαρμογή, έναν ιστότοπο που χρησιμοποιεί τι υπηρεσίε μα, ε, θα λάβουμε και εμεί πληροφορίε από αυτού. Αλλά δεν ξέρει απαραίτητο ο, χρήστη, ο συγκεκριμένο ιστότοπο αν είστε χρήστη του Facebook ή όχι. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν την αδειά του πριν μα στείλουν τι πληροφορίε ούτω ή άλλω και τι πληροφορίε μπορεί να τι χρησιμοποιήσουμε για πολλού σκοπού. Μπορώ να τι συζητήσω με περισσότερα λεπτομέρεια στη συνέχεια. Αλλά δεν δημιουργούμε παράλληλα προφίλ για κανέναν. Και πέραν αυτού, η προστασία δεδομένων είναι η καρδιά της, ε, του έργου μα. Όπω είπε και ο Μάρκο Ζουκεμπέργκ, δεν μπορεί να προστατεύσει κανεί τα δεδομένα του κόσμου, δεν ε, χρειάζεται να του προσφέρουμε τίποτα τότε. Η υπόθεση Cambridge Analytica ήταν ένας τρόπος να δούμε πώς αναπτύσσουμε και πώς λειτουργεί η πλατφόρμα μας και με τον κανονισμό GDPR ε, είχαμε και περισσότερη έμπνευση τα τελευταία χρόνια για να ψάξουμε τρόπου να βελτιώσουμε το πώ προσφέρουμε όλε μα τι υπηρεσίε. Να γίνουν σοβαρέ βελτιώσει στι πρακτικέ μα και, να... και βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μα. Σα ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να σα απευθύνω σήμερα το λόγο και είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Και τώρα να περάσουμε τι ερωτήσει. Ένα λεπτό για τον καθένα. Δύο λεπτά για την απάντηση. Στον κατάλογο μου μεθοδικά έχει καταρτιστεί κατά τη μέθοδο Ντεόντ, έχουμε μία αντικατάσταση. Ένα θα, ζητήσει, θα ρωτήσει δύο ερωτήσει, αυτό έχει συμφωνηθεί πριν την έναρξη τη ακρόαση. Και αυτό γιατί σε μία ομάδα λείπει κάποιο και έδωσε την ερώτηση του σε άλλον. Έχει κανονιστεί πριν αρχίσει καν η ακρόαση από τι πολιτικέ ομάδε. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Ντελβό, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Γιούρι Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ε, ερώτηση προς τον κύριο Ζάκελφιλντ. Δώσατε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει το Facebook τώρα για να προστατεύσει τα δεδομένα των χρηστών και λέτε ότι δεν αφορά τους Ευρωπαίους. Εφαρμόζεται την ίδια πολιτική και για πολίτες άλλων υπήρων. Ή πρόκειται για πολιτική που ασκείται ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέποντας το τι έγινε, πώς διευκολύνεται την πρόσβαση στη δικαιοσύνη χριστών οι οποίοι έχουν υποστεί ζημία. Ή αυτό πάλι έχει σχέση με τη δικαιοδοσία όπου κατοικούν οι χρήστες αυτοί. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Νομίζω εννοείται αν προσφέρουμε την ίδια προστασία στην Ευρώπη όπως και αλλού του κόσμου. Ναι, τις, τους ίδιους ελέγχους προσφέρουμε σε όποιον βρίσκεται απανταχού του κόσμου. Έχουμε διάφορες εφαρμογές που είναι, επιτρέπουν τον έλεγχο των δεδομένων. Ε, άλλο πρόγραμμα για την Ευρώπη, άλλα για, τους, για, τους, ε, για, την, για τον υπόλοιπο κόσμο. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν χώρες εκτός Ευρώπης που έχουν αναφιόμενα συστήματα προστασία δεδομένων και θέλουμε να ανταποκριθούμε και σε αυτά. Η δεύτερη ερώτησή σας είναι τι πράττουμε για να ανταποκριθούμε σε όσους ζητούν feedback για τις υπηρεσίες μας. Μα βασιζόμαστε σε αυτό, δηλαδή στο να ακρόμεθα τους ανθρώπους που ε, ε, έρχονται να μας μιλήσουν και συζητούμε και με νομοθέτες και με αυτούς που ε, ζητούν την προστασία της προσωπικής σφαίρας κλπ. Τους ακούμε και έτσι διαμορφώνουμε το προϊόν μας. Μάλιστα, ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση από εμένα, πρόεδρο της Επιτροπής Εμελιδών. Κύριε Σάτερφιλτ, προημερών ο New York Times δήλωσε ότι δίνει το Facebook τώρα πρόσβαση στην, ε, στη, στα δεδομένα. Ποιες είναι αυτές οι σχέσεις και ισχύουν ακόμα. η Cambridge Analytica έχει λάβει δεδομένα από το Facebook ως αποτέλεσμα της στόχευσης και τι είδους πληροφορίες ήταν αυτές. Τρίτο, σε ποιες πλατφόρμες στοχεύτηκαν χρήστες από πολιτικές ε, διαφημίσεις που είχε φτιάξει η Cambridge Analytica στο Facebook, σε άλλες πλατφόρμες ή και στα δύο. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω στην πρώτη σας ερώτηση ε, αναφέρεστε σε ειδήσει στο New York Times για σχέσεις που έχουμε με αυτούς που κατασκευάζουν συσκευές κλπ. για να προσαρμόζονται στο Facebook. Είναι σημαντικό να εξηγήσουμε τις σχέσεις που έχουμε με τρίτους που αναπτύσσουν εφαρμογές αρχίσαν αυτά το 2008-2010 όταν το οικοσύστημα εντό εισαγωγικών των κινητών τηλεφώνων ήταν πολύ διαφορετικό. Τώρα όλοι χρησιμοποιούμε διάφορα συστήματα Google, κατεβάζεται από ένα App Store την εφαρμογή και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε αμέσω. Αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα πάντοτε. Το 2010 υπήρχε πλήθος διαφορετικών ε, συσκευών και συστημάτων, BlackBerry, Palm... Ε, άλλα ε, συστήματα, άλλα λειτουργικά συστήματα και πλήθος τρόπων ε, να μπει κανείς στο διαδίκτυο. Και το Facebook ήταν ακόμα μια σχετικά νέα εταιρεία. Δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε εφαρμογές Facebook για όλες αυτές τις συσκευές και όλα αυτά τα λειτουργικά συστήματα. Γι' αυτό ήρθαμε σε εταιρικέ σχέσεις, δηλαδή κάναμε συμβάσεις με τρίτα μέρη για να αναπτύξουμε σχετικές εφαρμογές. Το ερώτημά σας είναι πόσες από αυτές έχουν παραμείνει. Νομίζω στην αρχή του έτους θα πρέπει να ήταν περίπου 55 60. Τις μειώνουμε σιγά σιγά όπως ανακοινώσαμε ήδη τον Απρίλη διότι και το iOS ως λειτουργικό σύστημα και το Android έχουν τροποποιηθεί. Έχουμε μειώσει στο μισό και στην ουσία θα τις τελειώσουμε όλες μέχρι τέλος του έτους. Η επόμενη ερώτησή σας αναφέρθηκε στην Cambridge Analytica και τις διαφημίσεις και αν ένας διαφημιστής λαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τους ε, ε καταναλωτές. Η Cambridge Analytica, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έλαβε δεδομένα Ευρωπαίων χρηστών. Εάν κάνουν διαφημίσεις θα λαμβάνουν ό,τι άλλο. Δηλαδή, ποιοι έκαναν κλικ στις διαφημίσεις, μια γενική δημογραφική ανάλυση των προσώπων αυτών και για ποιο λόγο συμβουλεύτηκαν τις διαφημίσεις αυτές οι χρήστες. Και η τελευταία σας ερώτηση, σε ποιες ιστοσελίδες έχει διαφημιστεί Cambridge Analytica. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν και τις δικές μας υπηρεσίες, Facebook κλπ. για διαφημίσεις. Ευχαριστώ. Ξεπεράσατε λίγο το χρόνο σας, αλλά απαντήσατε τις ερωτήσεις. Τώρα, η κυρία Μεσόλα από το Λαϊκό Κόμμα. Εμένα μου αρέσει το Facebook, γι' αυτό θα κάνω μια κάπως αντιδημοφιλή παρατήρηση και θεωρώ ότι είναι δύναμη καλού. Προέρχομαι από μια χώρα, τη Μάλτα εννοεί, όπου μέγα ποσοστό του πληθυσμού μας είναι χρήστης. Υπάρχουν όμως εγγενείς αδυναμίες και αυτό το απευθύνω σε εσάς κύριε Σέτερφιλτ. και αυτές οι αδυναμίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γνωρίζουμε ότι συλλέγονται δεδομένα από επιχειρήσεις όπως η Cambridge Analytica και χρησιμοποιήθηκαν μετά και στις Αμερικανικές εκλογές και στο δημοψήφισμα για το Brexit και χιλιάδες Μαλτέζοι έδωσαν δεδομένα τα οποία μετά χρησιμοποίησε κακώς ε, η Cambridge Analytica. Στη συζήτηση δεν τα έχω ακούσει ακόμα αυτό όμω. Να υποσχεθείτε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί δηλαδή. Ότι οι προσωπικέ πληροφορίε του καθενό είναι ασφαλεί στο διαδίκτυο. Και τι γίνεται για να προστατεύσουν καλόπιστε ιστοσελίδε ε, ειδήσεων οι οποίε δίνουν ε, σχετικά δεδομένα και μετά να προστατευτούν από τα λεγόμενα τρόλ που παρουσιάζουν ψευδείς ειδήσει. Μάλιστα. Το πρώτο για την Cambridge Analytica που επηρεάζει το Brexit. Επαναλαμβάνω ότι εξ όσων γνωρίζουμε η Cambridge Analytica δεν έχει λάβει πληροφορίες Ευρωπαίων χρηστών. Για τη δεύτερη ερώτησή σας, τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε την χρήση των εργαλείων μας. Ο κύριος Κάπλαν θα αναφερθεί σε αυτό σύντομα, αλλά να πω εγώ λίγα λόγια πρώτα. Όπως και εσείς είπατε, πολλές από τις καταχρήσεις των εργαλείων μας γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αποκρύψουν την ταυτότητά τους με ψευδείς λογαριασμούς. Ήδη από χρόνια ε, ρωσικές ιστοσελίδες το κάνουν αυτό. Μειώνουμε τώρα τον αριθμό των fake accounts και τα καταφέρνουμε όλο και καλύτερα. Μπορούμε να ποια από αυτά είναι ρομπότ. Μπλοκάρουμε τότε κάθε μέρα μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο. Ε, τέτοιους λογαριασμούς κάθε μέρα. Μειώνουμε επίσης τις ψευδείς ειδήσει. Κανένας δεν θέλει στο facebook να εμφανίζονται ψευδείς ειδήσει. Ούτε εμείς το θέλουμε, ούτε οι χρήστες μας το θέλουν συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη που ελέγχουν την αλήθεια των ειδήσεων μειώνουμε και τα οικονομικά κίνητρα, δηλαδή αντιδρούμε σε ιστοσελίδες που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία μας για να βγάλουν λεφτά. Έτσι λοιπόν, fake accounts, ψευδείς ειδήσει, η αντιμετώπιση τους αυξάνει τη διαφάνεια. Κάποιοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και τα εργαλεία μας διαφήμισης για να κυκλοφορήσουν ψευδείς ειδήσει. Το καλύτερο λοιπόν να φωτιστούν οι προσπάθειές τους αυτές. Μέσα στην εβδομάδα ήδη θα δώσουμε μια εφαρμογή View Ads που μπορείς να μπορεί να δείξει όλες τις αγγελίες που εμφανίζονται σε μια ιστοσελίδα. Εγώ βέβαια ξεπέρασα επίση τον χρόνο. Α παραμείνουμε όμω εντό των οριών ένα λεπτό και δύο λεπτά για την απάντηση. Λυπούμε και εγώ και εγώ μακρηγόρησα. Η κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω ερώτηση προς τον κύριο Σέταφιλ. Οι όροι χρήσης, το ακούσαμε, λένε σαφώς ότι η συλλογή δεδομένων μπορεί να καταλήξει σε άλλα μέρη. Δηλαδή το Facebook το ήξερε, έκανε συμφωνία με κάποιον περιλαμβάνοντας το σημείο αυτό ότι δηλαδή θα μπορούσαν να δοθούν τα δεδομένα σε τρίτο μέρος. Και αυτό πώς ευθυγραμμίζεται με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τότε για την προστασία δεδομένων και πώς μπορείτε να σχολιάσετε το γεγονός της μεταφοράς των δεδομένων αυτών, όχι μόνο εκεί, αλλά και σε όλους τους φίλους φίλων. Και επιτρέψτε μου εδώ να αναφερθώ και στην διαφήμιση, η οποία επηρεάζει τον ιδιωτικό βίο, γιατί το είδαμε. Μπορεί κανείς να τύχει χειραγώγηση σε ατομικό επίπεδο εξαιτία της διαφήμισης. Οπότε δεν είναι αλήθεια αυτό που λέτε για το ότι δεν είναι η διαφήμιση με την προστασία του ιδιωτικού βίου. Απάντηση. Πρώτον, ναι, η πολιτική προστασία ιδιωτικού βίου όντω ζητάει τη συνένεση για να μπορούν τα δεδομένα να βγουν πέρα από την ε, application αυτή του Facebook. Βέβαια, οι κανόνες δεν περιλαμβάνουν το τι μπορεί ο καθένας να συμπεριλαμβάνει στη δικιά του την πολιτική. Δηλαδή δεν μπορούμε τις δικές μας τις πολιτικές να τις εφαρμόσουμε πέρα από το δικό μας ε, το πεδίο. Και αυτά που έλεγαν οι δικοί μας οι κανόνες προφανώς και απαγόρευαν να πάνε τα δεδομένα των χρηστών μας ε, στην ε, Cambridge Analytica. Όπως επίσης απαγορεύεται και η πώληση δεδομένων η μεταφορά σε άλλες εταιρείε κλπ. Τώρα για το φράνστετ εδώ οι διάφοροι developers κανονικά ζητούν την άδεια των χρηστών. Μπορούν να μεταφέρουν τα δίκτυά τους σε άλλες εφαρμογές. Όμως ακούσαμε από πολλούς για αρκετό καιρό να λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα και το κάναμε το 2014, αλλάξαμε την πλατφόρμα μας. Ακούσαμε πιο πρόσφατα ότι πολλοί θα ήθελαν να είναι πιο εύκολο να έχουν το δίκτυο φίλων και εκτός ε, Facebook. Οπότε αυτά είναι θέματα με τα οποία προβληματόσατε ακόμα. Τώρα για τη σχέση τη προστασία ιδιωτικού βίου με τη διαφήμιση. Είναι εντάξει, φυσικά και υπάρχει κάθε φορά που χρησιμοποιείτε προσωπικά δεδομένα για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να έχετε υπόψη στην προστασία δεδομένων. Και κάνουμε πολλά για να υπάρχει διαφάνεια και να έχει έλεγχο ο χρήστη. Ευχαριστούμε. ECR Dalton. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σάταλφιτ και εγώ για εσά έχω ερώτηση. Ακούμε πολλά εδώ για τις ανησυχίες του κόσμου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων τους και δεδομένης της φύσης του σκανδάλου, ότι δηλαδή έγινε κατάχρηση των δεδομένων, θέλω να ξέρω στην πράξη ποιες είναι οι επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη των χρηστών. Οπότε, πέσανε τα έσοδά σας στην Ευρώπη μετά το σκάνδαλο αυτό και πώς εγκατέλειψαν το Facebook από τους χρήστες, έκλεισαν του λογαριασμούς του μετά το σκάνδαλο αυτό. Θα ήθελα νούμερα, παρακαλώ. Απάντηση. Τα νούμερα τα δώσαμε στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Και αυτά μπορώ να σας δώσω και ήταν θετικά. Συνεχίζουμε βέβαια να τηρούμε τις προδιαγραφές για όλα και θα υπάρξει και μετά το επόμενο τρίμηνο και νέα, θα υπάρξουν νέα δεδομένα, νέα στοιχεία. Άξελ Φως, ΕΛΚ, μέλος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Γέλινεκ. Αλλά πρώτα μια διευκρίνηση. Με συγχωρείτε κύριε Βος, ποια στιγμή να φορέσουν τα ακουστικά τους οι, οι παριστάμενοι ε, διακόπτη πρόεδρος. Έλεγα λοιπόν, συνεχίζει ο ότι έχω την αίσθηση ότι αυτή η καταστρατήγηση των διατάξεων του GDPR δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ακόμα περισσότερους νόμους. Χρειάζεται να αυξηθεί το επίπεδο των ελέγχων. Δεν ξέρω πώς βέβαια μπορεί να γίνει αυτό, διότι ούτε και το ποινικό δίκαιο έχει ε, δύναμη εδώ. Διότι λέει και εκεί απαγορεύεται το κλέπτην και όμως ε, οι κλοπές γίνονται. Ερώτηση προς την κυρία Γέλινεκ. Έχει εγγύψει στο θέμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και εάν έχει ασχοληθεί και έχετε ασχοληθεί και εσείς επομένως ποια είναι τα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τους ελέγχους και πώς είναι ενδεχομένως δυνατόν να βελτιωθεί ο έλεγχος στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Ευρωβουλευτά για την ερώτηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έχει συνέλθει μία φορά στις 25 Μαΐου επόμενη συνεδρίαση ναι, υπάρχει μόλις από την 25η Μαΐου. Η επόμενη συνάντηση προβλέπεται 4 και 5 Ιουλίου. Στην ομάδα εργασίας άρθρου 29 έχουμε ήδη συζητήσει διάφορα θέματα, βεβαίως και τους ελέγχους και στο εθνικό επίπεδο, αλλά η κοινοτική διάσταση της εργασίας άρχισε στις 25 Μαΐου, διότι πρόκειται και για όργανο το οποίο έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις. Το ερώτημα θα είναι πώς μπορούμε όχι μόνο να αντιδράσουμε, αλλά να δρούμε και προληπτικά. Διότι ως τώρα έχουμε 29 υποθέσεις διαμεθοριακού χαρακτήρα, τις οποίες έχουμε αναρτήσει στο κοινό μας σύστημα και οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φάση της έρευνας. Πέραν όμως από τις υποθέσεις οι οποίες μας γίνονται γνωστές μετά από καταγγελίες, θα προχωρήσουμε όπως σας είπα και προληπτικά. Ευχαριστώ κυρία Αναγκόμες των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ε, προς τον κύριο Σάτερφελτ και εγώ. Η Cambridge Analytica ήταν μια περιορισμένη ευθύνη ε, στη Μεγάλη Βρετανία και με ε, δράση για την προεκλογική εκστρατεία. Και στην Καραϊβική ανέλαβε δράση και πολλές φορές χρησιμοποίησε παράνομα στοιχεία των ε, μελών της αντιπολίτευσης. Έχετε καθόλου πληροφορίες για το κατά πόσο αυτά τα δεδομένα που αρχικά τα ψάρεψαν στο Facebook και πρόσφατα σε επιστολή με ημερομηνία 13 Ιουνίου παροτρύνεται το Facebook να υποβληθεί σε εξωτερικό ανεξάρτητο, έλεγχο. Ε, δεν ακούσαμε καμιά απάντηση από το Facebook. Θα το δεχόσαστε αυτό, ε, κάποιον εξωτερικό έλεγχο για την πρακτική σας σε σχέση με τα δεδομένα. Και αν όχι, γιατί. Ε, μιλήσατε για την ε, ποινική ε, έρευνα του Ηνωμένου Βασιλείου γιατί όχι για αυτήν την ε, αίτηση, το νέο αίτημα που έχει υποβληθεί. Ναι, για τις πρακτικές ε, της ACL στο KITS και στα, στις νήσους Νίβεν δεν γνωρίζω ακριβώς τι συνέβη, με συγχωρείτε. Είναι ανησυχητικό αυτό που λέτε, αλλά δεν τις γνωρίζω αυτές τις κατηγορίες και δεν μπορώ να τις σχολιάσω. Όσο για την ερώτησή σας για εξωτερικό έλεγχο θα έλεγα ότι το Facebook ελέγχεται συστηματικά και από εξενάρτητο τους ελεγκτές στις ίπα και από την αρχή προστασία των δεδομένων στην Ιρλανδία. Δύο-τρεις φορές έχει γίνει αυτό τουλάχιστον. Υπάρχει σχετικός ε, υπεύθυνο στην Ιρλανδία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε με τον ε, επόπτη προστασίας δεδομένων της Ιρλανδίας στενά και βεβαίως ξέρω ότι με το GDPR σε ισχύ, σε ισχύ αυτή η διαρκής παρακολούθηση θα συνεχιστεί. Το ίδιο και η αρμόδια αρχή στις ΗΠΑ που μας απαιτεί, μας ε, υποχρώνει ε, αναδιαιτία να σε έλεγχο. κυρία Ιντφελτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούω το ίδιο το Facebook να μιλάει. Και είναι περίεργο να είμαι εδώ και να το ρωτάω εάν θα τους πείραζε να ακολουθήσουν τον νόμο και να τον τηρήσουν και αν τους ε, ενοχλεί αυτό. Πραγματικά η αφοσίωσή σα στον ιδιωτικό βίο πολύ με συγκινεί, αλλά θα ήθελα να μπορούμε να επαφιόμαστε στον νόμο και στου φορεί ε, που είναι υπεύθυνοι για την τήρησή του. Γιατί σα πήρε τόσο καιρό ε, πρωτού να αρχίσουν οι επόπτε προστασία δεδομένων να κινούνται και γιατί λέτε ότι από εδώ και μπρο θα είστε και προ όπω λέγεται, δραστήριοι για όλο το θέμα αυτό, διότι το Facebook έχει και πολύ θετικέ πτυχέ. Δηλαδή, μην τα πετάξουμε όλα στον κάλαθο των αχρήστων με τη μία, αλλά πραγματικά είσαστε μια εξαιρετική ε, δύναμη από μόνοι σα. Έχετε πολλέ δυνατότητε. Δεν πρέπει κάπω ε, διανοητικό να προσαρμοστείτε στη νέα κατάσταση. Τι θα κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί και ότι αυτέ οι σπάνιε υποθέσει που έδειξαν ότι το Facebook δεν είναι τόσο αφοσιωμένο και ταγμένο στην ιδιωτικότητα όπω ακούσαμε, εσεί τι θα κάνετε για να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να προστατευτούν τα δικαιώματά μα. Αυτή η ερώτηση πηγαίνει προφανώς σε έναν και μόνο άνθρωπο την κυρία Γέλινεκ. Κύριε Γέλινεκ, απαντά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ευρωβουλευτά. Όλες οι κυβερνήσεις πριν από την θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού αύξησαν το προσωπικό των Εθνικών Αρχών Εποπτείας. Είναι προφανές ότι δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό ακόμη παρόλα αυτά όλες οι Εθνικές Αρχές Εποπτείας Δεδομένων. Ωστόσο, βάζουμε τώρα μπρος τον μηχανισμό που προβλέπει και επιτρέπει τη λειτουργία του η, ο βασικός κανονισμός. Δηλαδή θα υπάρχει μία αρμόδια επί αρχή η οποία συντάσσει ένα σχέδιο και όλες οι ενδιαφερόμενες, όλες οι θυγόμενες δηλαδή εθνικές αρχές μπορούν να συμμετάσχουν και ενδεχομένως και με ερωτήσει ή και με προβολή επιφυλάξεων. Και εάν δεν αρκέσει αυτό, τότε φτάνουν πλέον οι υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, Εποπτείας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτή του είδους συνεργασία δεν υπήρχε ως τώρα. Προβλέπεται τώρα από τον βασικό κανονισμό και στην βάση των εργασιών της ομάδας ε, εργασίας Άρθρο 29 που παίζει συμβουλευτικό ρόλο και η οποία και πριν από την θέση σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού έχει εκδώσει πολλές κατευθυντήρες γραμμές. Αφενός, αφετέρου, έχει βεβαίως και όλες τις δεκαετίες προηγουμένως εκδώσει γνωμοδοτήσεις και έχει συμβουλεύσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις. Όμως, δεσμευτικές αποφάσεις μόνο από τούδε έχουμε δυνατότητα και δικαίωμα να λαμβάνουμε. Ένα πράγμα είναι σαφές. Διερευνούμε ακριβώς και δεν μπορούμε από την πρώτη μέρα κιόλας να βγούμε να επιβάλλουμε ποινές. Έχουμε διαδικασίες κράτους δικαίου και είναι απαραίτητο να τηρούνται οι διαδικασίες αυτές και να, υπάρχει προστασ... Ε, να υπάρχουν μηχανισμοί προστασίας της ένωμης τάξης στην Ευρώπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το προβλέπει ο βασικός κανονισμός. Δώστε μας μια ευκαιρία να αποδείξουμε αυτά που λέμε. Ευχαριστούμε ο Κάρλος Κουέλιο για το ΕΛΚ και τη ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ προς τον κύριο Σάτερφιλ θέλω να θέσω ερώτηση. Υπάρχουν περισσότεροι Ευρωπαίοι χρήστε στο Facebook από τα Αμερικανοί. Και ο κύριο Ζούκερμπεκ είπε ότι το GDPR θα είναι πηγή έμπνευση που πρέπει να ακολουθηθεί. Και το είπατε και εσεί στην ομιλία σα. Το θυμήσατε. Στην πράξη όμω ε, είπε ότι θα πρέπει να περάσουν οι περισσότεροι χρήστε ε, στο καθεστώ προστασία των. Ε, μάλλον το καθεστώ προστασία αυτό πρέπει να ισχύσει και για του χρήστε τη ΕΠΑ. Γιατί όμω δεν έγινε αυτό ακόμα. Και για του Ευρωπαίου πολίτε, πώ μπορείτε να, να βεβαιώσετε ότι ακολουθείτε το GDPR. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Και πάλι πρέπει να πω ότι τα ίδιες ρυθμίσει και τα ίδια στοιχεία ελέγχου που ισχύουν στην Ευρώπη ισχύουν και αλλού. Αυτά τα setting, αυτά τα control τα αναπτύξαμε λόγω του GDPR και ισχύουν για όλους τους χρήστες παγκοσμίω. Η δεύτερη ερώτησή σας ήταν νομίζω... Για το τι εγγυήσει μπορούμε να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους χρήστες ότι θα ακολουθήσουμε τον νόμο και θα τηρήσουμε τον GDPR. Μα το τηρούμε. Δύο χρόνια μας πήρε η συμμόρφωση. Ξέρω όμω ότι δεν σα ενδιαφέρει να με ακούσετε απλώ. Θέλετε να το δείτε και στην πράξη. Άρα, τι να πω. Απλώ θα πρέπει να το δείξουμε. Ε, Σχεδιάζοντα τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση. Η πρόσβαση και η φορητότητα των δεδομένων είναι στοιχεία τα οποία τα συζητούμε πολύ. Ε, τώρα μεν, αλλά για να τα διασφαλίσουμε αυτά τα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, πραγματικά και χρόνο και χρήμα να σπαταλήσαμε. Δεν είναι τυχαίο. Είναι κάτι που το λαμβάνουμε υπόψη το GDPR στην πρόσβαση τη πληροφορία σα. Το να μπορεί κανεί να δει τι πληροφορίε του παντού, να τι κατεβάσει, είναι ένα θέμα. Επίση, η πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο πρωτοφορητότητα η ίδια. Δεν έχουμε περιορίσει τι πληροφορίε που μπορείτε να πάρετε εσεί από την πλατφόρμα η πλατφόρμα είναι ένας τρόπος να πάρει κανείς τις πληροφορίες εκτός Facebook εφόσον θέλει να τις μοιραστεί κανείς με άλλους σχεδιαστές προϊόντων για να ζήσουν και αυτή τη δική τους εμπειρία. Αλλά νομίζω πιο πολύ πρέπει να σας πείσουμε με τις πράξεις μας και με τα λόγια μας. Ναι. Ε, έχει γίνει αντικατάσταση στο επόμενο σημείο. Η κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ. Την κυρία Γελίνεκ θέλω να ρωτήσω τώρα. Είπατε ότι έχετε 29 διασυνοριακές υποθέσεις, ίσως είναι πολλές. Για τις έρευνες Πασιζόμαστε στους επόπτες προσωπικών δεδομένων, έτσι. Η συνεργασία μεταξύ τους πώς λειτουργεί. Έχουν αρκετό προσωπικό ή έχουν τη σωστή νοοτροπία την σωστή προσέγγιση. Ο Ιρλανδός, ακούσαμε, ίσως δεν είναι τόσο φιλικός όσον αφορά την προστασία του ιδιωτικού βίου. Οπότε εσείς πώς χειρίζεστε αυτές τις αποκλίνουσες μερικές φορές στάσεις και προσεγγίσεις μεταξύ των εποπτών προσωπικών δεδομένων. Και μια δεύτερη ερώτηση παρακαλώ. Ο κανονισμός τώρα προστασίας ε, ηλεκτρονικών δεδομένων είναι επίση αρμοδιότητα του επόπτη. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές απόψεις των ε, αρχών προστασίας δεδομένων, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ειδικά αυτό είναι από τα πιο σημαντικά σημεία. Δηλαδή, απαιτείται σύγκληση, την οποία σύγκληση θα επιτύχουμε στο Συμβούλιο. Από τα πιο σημαντικά μας καθήκοντα είναι να γεφυρώσουμε τις υφιστάμενες διαφορές και να καταλήξουμε σε ενιαία άποψη και βέβαια σε ενιαία λήψη αποφάσεως. Και η ενιαία αυτή άποψη στην διόδη των περιπτώσεων θα ληφθεί ομόφωνα, αλλιώς προβλέπεται πλειοψηφία δύο τρίτων. Δύο φορές εάν δεν επιτευχθεί αυτό, τότε λαμβάνεται πλέον η απόφαση με απλή πλειοψηφία. Και εάν είναι ισοψηφία, τότε κρίνει την έκβαση η ψήφος του ή της Προέδρου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που περιλαμβάνεται σχετικά στον βασικό κανονισμό. Εξάλλου σημαντικό είναι ότι όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και, στο, και επί το παρόντος, δηλαδή συνεργάζονται στενά όλες οι αρχές προστασίας δεδομένων και στο παρελθόν έχουμε εκδώσει όχι μόνο γνωμοδοτήσεις αλλά και κατευθυντήρες γραμμές οι οποίες επιβεβαιώθηκαν τώρα από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο και που έχουν σχέση με τον βασικό κανονισμό. Έχω δε απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλες και όλους τους συναδέλφους μου ότι θα φροντίσουν να εφαρμοστεί ο κανονισμός κατά γράμμα. Κάτι το, για το οποίο δεσμευόμαστε όλες και όλοι. Γιάνν Άλμπρεχτ των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Σάτερφιλτ και και τους υπολείπους. Λέτε ότι, ότι σέβεστε τον νόμο της χώρας όπου δραστηριοποιείστε. Αν και φαντάζομαι ότι ίσως υπάρχουν και άλλες ιδεοντολογικές ιδέες, διότι ίσως είναι διαφορετική η νόμη προστασίας των δεδομένων στην Ευρώπη και στην Κίνα λέτε ότι συμμορφώνεστε με τον νόμο. Υπάρχουν όμως πλήθος αποφάσεων σχετικά με την χρήση των ε, δεδομένων Facebook εδώ στην Ευρώπη. Διαρωτώ με λοιπόν, ακούγοντας τις απαντήσεις σας, σε ποια νομική βάση το, το κάνετε αυτό. Και αν επικαλείστε ένομο συμφέρον, πώς το δικαιολογείτε εν προκειμένου. Πώς ορίζετε το ένομο συμφέρον στις διαδικασίες σας και στην επεξεργασία δεδομένων δηλαδή. Λέτε ότι επίσης δεν υπάρχουν δεδομένα προσώπων που δεν χρησιμοποιούν τις εφαρμογές. Αλλά χρησιμοποιείτε δεδομένα προσώπων που χρησιμοποιούν ιστοσελίδες. Ε, ποιο είναι το, ποιος είναι όμως ο ταυτοποιητής για, αυτές, για αυτά τα σύνορα δεδομένων. Ευχαριστώ κύριε Άλμπρεχτ απάντηση. Για την νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων και μέσω των υπηρεσιών και εφαρμογών μας. Αυτά τα διακόπτει ο κ. Σάλβος χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Έχουμε συμβάσεις με τους χρήστες ένομο συμφέρον είναι αυτό που απορρέει από τον νόμο. Εξετάζουμε το συμφέρον, εξετάζουμε και τη, τα προσωπικά ε, δεδομένα, δηλαδή τα, συμφέροντα των προσώπων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας και το να προσφέρουμε ασφάλεια βεβαίως είναι και ένα από τα δεδομένα. Μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιον που κάνει ζημιά και να τον εμποδίσουμε από το να κάνει ζημιά και στις άλλες υπηρεσίες και εφαρμογές μας. Χρησιμοποιούμε ωστόσο τη συλλογή δεδομένων μόνο για εσωτερική χρήση για την αποφυγή spam κλπ. Σχετικά με την διαδικασία δεδομένων μη χρηστών και ποιος είναι ο νέος ταυτοποιητής. Όταν ένα, ένας τρίτος ενσωματώνει ας πούμε, το κουμπί like και το χρησιμοποιεί σε μια δική του εφαρμογή και το χρησιμοποιεί σε μια εφαρμογή του. Λαμβάνουμε πληροφορίες όπως άλλωστε η κάθε επιχείρηση. Επομένως και μια διεύθυνση IP και οποιαδήποτε cookies μπορεί να υπάρχει ένα ενέργειο ταυτοποιητή εκεί. Όλες αυτές οι πληροφορίε είναι αναγκαίες για να μπορέσουμε να προσφέρουμε την βασική υπηρεσία. Και πρέπει να υπάρχει και μια διεύθυνση IP για να ξέρουμε πού να στείλουμε το κουμπί like. Υπάρχουν λοιπόν ενιαίοι ταυτοποιητές. Όπως, όπως είπα, και, είπα και πριν, οι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε δεδομένα μη χρηστών είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Κάποιες αναλύσεις και ε, κυρίω για να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίε. Um, next is Joseph Mr. Don't injure yourself. I have to keep to the default list. Okay, calm, stay calm, stay calm. Yeah. Ήρεμα, λέει ο πρόεδρο, ήρεμα. Μην, δεν χρειάζεται να τρέξετε. Ο κύριο Βό του Λαϊκού Κόμματο, που είναι και μέλο τη Επιτροπή Θεμελιών Ελευθεριών. Ερώτηση προ τον κύριο Σάτερφιλτ, αλλά μην ανησυχείτε, θα μιλήσω γερμανικά. Η ερώτηση που θέλω να υποβάλω έχει γίνει και πριν, κυρίως για τις ψευδείς ειδήσει και την διάδοσή τους. Επειδή όμως αυτά λίγο πολύ απαντήθηκαν, έχω να πω ότι με απασχολεί ακόμη το εξή ερώτημα. Τι πρέπει να γίνει ακριβώς στο μέλλον και τι πρέπει ενδεχομένως να κάνουμε εμείς, να βελτιώσουμε εμείς εδώ, ώστε να μην μπορούν να επαναληφθούν τέτοια πράγματα σαν αυτά που έγιναν. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένες ιδέες σχετικά με το πού εντοπίζονται κενά, ποιες δυνατότητες έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το ενδεχόμενο αυτό. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ανέφερα προηγουμένω κάποιε από τι προσπάθειε που κάνουμε για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων. Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα το ερώτημά σα είναι ευρύτερο. Τι μπορούμε να κάνουμε ω κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο κανεί δεν θέλει να δει ούτως ή άλλως στο ίντερνετ. Κάτι που μπορούμε να κάνουμε και θα θέλαμε να το δούμε και περισσότερο είναι κάποια εκπαιδευτική προσπάθεια. Δηλαδή πώς μπορεί κανείς να εντοπίσει τις ψευδείς ειδήσει, πώς μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα τις πηγές τους. Κάτι που κάνει το Facebook είναι να προσπαθούμε να μεταφέρουμε ειδήσει από ευρεία αξιοπιστία πηγέ. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μα αυτό. Χρειάζεται ε, να βοηθήσουμε τον κόσμο να είναι πιο αντικειμενικός κριτής των ειδήσεων. Κάτι όπου μπορούν να βοηθήσουν και οι κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα χρειαστεί όμως μεγάλη προσπάθεια από πλευράς πολλών φορέων. Όμως η εκπαίδευση του κοινού, ώστε να γίνει πιο ε, κριτικός καταναλωτής των ειδήσεων στο ίντερνετ, αυτή έχει κέρια σημασία. Βάιντεν Χόλτσερ Ιωσήφ Ευχαριστώ. Ερώτηση προς την κυρία Γέλινεκ. Προεβδομάδων το Facebook έκανε μια μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία δηλώνοντας ότι θα τηρήσει τον κανονισμό προστασίας δεδομένων. Έχετε να σχολιάσετε κάτι. Δεύτερο, για την εφαρμογή στις διάφορες χώρες μέλη. Διαπιστώνεται ε, προβληματικές καταστάσεις θεωρείτε ότι κάπου υπάρχουν άσχημες πρακτικές. Τρίτο, ενίσχυση των, των δικαιωμάτων των καταναλωτριών σε ό,τι αφορά την... το ενδεχόμενο να δοθεί δυνατότητα συλλογικών αγωγών. Ευχαριστώ για την ερώτηση σας. Αρχίζω με την τελευταία ερώτησή σας. Δικαίωμα συλλογικών αγωγών. Μια δυνατότητα που θα πρέπει να ανοίξουν οι χώρες μέλη. Στην Αυστρία δεν δόθηκε αυτή η δυνατότητα από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Σε άλλες χώρες υπάρχει. Θα ήταν μια δυνατότητα που θα επέτρεπε μια καλύτερη αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών. Δεύτερο, Καλέ πρακτικές. Ο κανονισμό ισχύει εδώ και τέσσερι εβδομάδε. Έχουμε διαπιστώσει ότι η συνεργασία μεταξύ των αρχών είναι καλή. Έχουμε και ένα template, ένα πρότυπο δηλαδή ηλεκτρονική τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιείται. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή στι 28 χώρε μέλη, ένα πράγμα καθίσταται σαφέ. Είναι άμεσα εφαρμοστέο ο κανονισμό, Επομένως, εφαρμόζεται και χωρίς λήψη συνοδευτικών μέτρων ή άλλης νομοθεσίας. Βέβαια χρειάζεται κάποια προσαρμογή των ε, εθνικών νομοθεσιών προστασίας δεδομένων. Η πρώτη σας ερώτηση ήταν, με συγχωρείτε τη λησμόνησα, πέστε μου πάλι. Α, η, η διαφήμιση, η διαφήμιση, ναι. Ναι, ναι, που χάρηκα που την είδα, λέει ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ, αλλά το θέμα είναι το εξής. Συνεχίζει η κυρία Γέλνικ. Εισαγωγικά είπα ότι θα ήταν καλύτερο να κάνουν εξ αρχή επιχειρήσει επιχειρήσεις επενδύσεις στην προστασία δεδομένων, ώστε να αποφύγουν μετά τις δαπάνες για εκστρατείες διαφήμισης που να ζητούν συγγνώμη στην ουσία κλπ. Δεύτερο, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προσπάθειες. Τώρα, αν οι προσπάθειες αυτές είναι επαρκείς, αυτό θα προκύψει από την διερεύνηση των επιμέρους υποθέσεων. Δεν μπορώ να προκαταλάβω τις έρευνες και ούτε θέλω, διότι υπάρχουν αυτές τις στιγμές αυτή τη στιγμή υποθέσεις που ερευνώνται. Τα γνωρίζει αυτά το Facebook, τα γνωρίζετε και εσείς από τις ε, εφημερίδες. Η κυρία Σπινέλη. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια εμπορική εφεύρεση που τελικά δεν τα αποκρίνεται στα δικαιώματα, τα ιδιωτικά δικαιώματα. Έχω κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Ντέι. Πώς μπορεί να ξέρει ένα άτομο ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του και ότι το προφίλ του κάποιος το πειράζει. Οι προσφυγές, οι ατομικές κοστίζουν πολλά. Το δικαστήριο όμως έχει περιορίσει τα δικαιώματα των Χριστών γιατί λένε ότι μόνο ο αρχικός συμβαλόμενος μπορεί να προσφύγει. Υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί αυτό στην ομολογία. Έπειτα, το άρθρο 80 του κανονισμού προστασίας ε, δεδομένων είναι αρκετά σαφές προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς μπορούν να γνωρίζουν ε, οι χρήστες. Το σύστημα πράγματι είναι πάρα πολύ περίπλοκο και μπερδεμένο και για τις επιχειρήσεις που δρούν στον κλάδο. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι φορείς που ο ρόλος τους είναι να ετοιμάσουν πληροφορίες για κάποιον άλλον μπορείτε να πάτε και να ρωτήσετε, να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται, αλλά υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι φορείς οι οποίοι οργανώνουν τις πληροφορίες, αλλά δεν δουλεύουν για σας, δουλεύουν για κάποιον άλλον. Και το πρόβλημα είναι ότι θεωρούνται όχι οι ελεγκτές, αλλά processors, αυτοί οι οποίοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες, οπότε κρύβονται ουσιαστικά, προστατεύονται. Ελπίζω να πετύχουμε στήριξη από τις αρχές προστασίας δεδομένων για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση εκεί. Όσον αφορά τώρα το άρθρο 8 και τις προσφυγές, νομίζω ότι το πρόβλημα τώρα είναι για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να εντοπίσουν τέτοιες περιπτώσεις και νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί κανείς να το προσεγγίσει και τελώς διαφορετικά. Αν έχουμε καλές υπηρεσίες που προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες να οργανώνουν την πληροφορία τους και να μην υπάρχουν κίνητρα να υπάρχουν ε, επιχειρήσεις που να χρησιμοποιούν τα δεδομένα των χρηστών σε βάρος τους, τότε θα κανονιζόταν το πρόβλημα από μόνο του. Οπότε το θέμα είναι να προσανατολίσουμε τον κόσμο στις σωστές διαδικασίες προσφυγής. Γνώμη μου είναι ότι θα δούμε τι θα γίνει και πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει ως άτομα για το τι θα κάνουμε. Υπάρχουν ευκαιρίες. Ευχαριστούμε κυρία Γιούροκα. Έλκα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Δύο-τρεις από τις προτάσεις σας θα ήθελα να μας τις δώσετε συγκεκριμένα για αυτές που μιλάτε στην ομιλία σας που είπατε πριν. Τώρα, άλλο είναι να γίνεται χειραγώγηση γιατί τι θα μπορούσατε να κάνετε παραπάνω για τους χρήστες σας, οι οποίοι όμως είναι ανήλικοι, κάτω το 18. Βλέπετε η ανησυχία μας είναι ότι γίνεται η χειραγώγηση των ε, νέων, των ανήλικων, των παιδιών. Έχετε διαπιστώσει τέτοια φαινόμενα. Γιατί βλέπετε όταν τα παιδιά μας είναι στο facebook πρέπει να μπορούμε να ξέρουμε τα δεδομένα τους που φτάνουν. Εσείς δηλαδή ε, πρέπει να ξέρετε που έφτασαν τα δεδομένα του παιδιού σας και μπορείτε να προσφύγετε εναντίον αυτών που έχουν κλέψει τα δεδομένα μας. Ακόμα και αν δεν μας έχουν χειραγωγήσει πολιτικά. Γιατί αυτό είναι το κύριο πρόβλημα των χρηστών σας. Ε, ναι, δύο ερωτήσεις, ναι. Είναι λίγο γραφικατικό, αλλά παραβαίνει στους κανόνες. 20 seconds, I promise you 20 seconds. So... Ωραία. Πρόεδρο, να είμαστε ευέλικτοι. Ωραία, να είμαστε ευέλικτοι, μια που κάνετε δύο ερωτήσει σε δύο διαφορετικού ε, ομιλητέ. Λοιπόν, το πρώτο φτηνό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προωθηθεί η πρόσβαση. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι θα ήθελαν πάρα πολύ να χρησιμοποιήσουν ε, το δικαίωμα πρόσβασης. Θα πρέπει βέβαια οι αρχές προστασίας δεδομένων να τους αθαρρύνουν. Τότε θα έκαναν ε, τη δουλειά τους και δεν θα κόστιζαν παραπάνω. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση. Δεύτερον, να ψάξουμε τα δεδομένα που έχουν να κάνουν ε, με την διασταύρωση των εφαρμογών με τις πλατφόρμες. Γιατί εκεί έγκυται και το σκάνδαλο της Cambridge Analytica. Ο συνδυασμός λοιπόν των δύο δημοσιογράφων να μπορούν ε, να ε, ψάξουν περισσότερο. Ωραία και ο κύριος Σάταφιλτ. Ευχαριστώ και εγώ για τις ερωτήσεις σας που είναι όντως πολύ σημαντικές μιλάτε για τα δεδομένα των ανηλίκων και πώς χρησιμοποιούνται αυτά για τη διαφήμιση και οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι που παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Φυσικά και ο κανονισμός προστασίας δεδομένων, ε, ε, προσωπικών δεδομένων λέει πάρα πολλά και για τους ανήλικες και την ηλικία. Οι προτάσεις του κανονισμού λένε ότι οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται στους νέους και στα παιδιά με τρόπο που να τις καταλαβαίνουν. Και αυτό προσπαθούμε κι εμείς να κάνουμε, να βοηθήσουμε τους νέους να καταλάβουν τι σημαίνει η πρόσβασή τους, τι σημαίνουν οι πληροφορίες που δίνουν. Και αυτό όμως είναι γενικότερο για το πώς αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες θα έπρεπε έτσι κι να το κάνουμε πάρα πολύ νωρίς, να αρχίσουμε να διδάσκουμε στα παιδιά μας πώς να αντιλαμβάνονται τις ειδήσει, τις πληροφορίες, τα νέα, πώς να είναι επικριτικοί απέναντι σε αυτά. Αυτό είναι κάτι πολύ γενικότερο. Πρόεδρος, ναι, τώρα να τηρούμε το χρόνο μας μέχρι τις 5 για να περάσουμε στο επόμενο. Σοσιαλιστές, η κυρία Σίπελ εκ μέρους της Ήτρε αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σάτερφιλ, προηγουμένως είπατε ότι το Facebook συνήψε εμπορική σχέση με διαφημιστική, της οποίας οι όροι και οι προδιαγραφές προέβλεπαν την πώληση δεδομένων σε τρίτα μέρη. Άρα το τρίτο μέρος ε, παραβίαζε τους κανόνες. Άρα εν γνώση σας ε, προβήκατε στη σύναψη αυτής της εμπορικής σχέσης και βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου εσείς είστε αυτός που ελέγχει νομίμως, εσείς είστε υπόλογοι και υπεύθυνοι. Άρα και πάλι Πώς μπορείτε πραγματικά να δικαιολογήσετε τη συμπεριφορά σας σε εκείνη τη χρονική φάση και να λέτε ότι τότε ακολουθήσατε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ε, είμαι βέβαιος ότι το ακολουθήσαμε. αλλά ο τρόπος που χειριστήκαμε την Cambridge Analytica ήταν ε, τελείως ε, νομοφανής. Ε, θα συζητηθεί πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ακολουθήσαμε τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ακολουθήσαμε τον νόμο. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι θέμα ε, πίστης. Δεν κάνουμε, κάνουμε κουβέντα για θρησκεία εδώ πέρα. Καμιά συγκεκριμένη απόδειξη μπορείτε να μας δώσετε. Πού να λέτε ότι ακολουθείτε τους κανόνες και να λέτε ότι ως αυτός που είναι σε θέση να ελέγξει δεν πέρασε σε παράνομη σχέση. Με όλο το δέοντα σεβασμό, ο τρόπο που χειριστήκαμε την υπόθεση Cambridge Analytica θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο όταν ανακαλύψαμε ότι ο Δρότερ Κόλγαν είχε παρανόμως μεταφέρει πληροφορία στην Cambridge αναλυτικά, παραβιάσαμε τη σχέση εμπιστοσύνη με τον κόσμο που καθημερινά εξυπηρετούμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε τώρα, σε αντιδιαστολή με το παρελθόν. Οι επερωτήσεις δεν επιτρέπονται, αλλά είναι πολύ βαρετό άμα δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν είναι τη ανθρώπινη φύση να μην μπορεί κανεί να διακόψει κανέναν από του ομιλητέ ποτέ. Ο Μάρκο Τζούλο από την EFTD. Ευχαριστώ στον εκπρόσωπο της Personal Data. Μιλάμε τώρα για το Facebook, αλλά είναι ένα παράδειγμα. Το Facebook είναι ένα σύστημα το οποίο αντικατοπτρίζει το κοινωνικό μοντέλο εντό του οποίου ζούμε. Πρέπει να προστατεύσουμε περισσότερο τους χρήστες, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει λίγο αυτό το κοινωνικό business model να ε, το εξετάσουμε. Το Facebook κάνει πολλά για να προσφέρει στους χρήστες την δυνατότητα να ελέγξουν τη ροή των δεδομένων τους και πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Όμως παραμένουμε πάντοτε αγκιστρωμένοι και περιορισμένοι σε ένα σύστημα κλειστό. Ο εκπρόσωπος της Personal Data μα το είπε, το υπενήχθηκε. Μίλησε για τη φορητότητα των δεδομένων. Το να επιμείνουμε λοιπόν στην φορητότητα, δηλαδή το σύστημα να ανοίξει και να υπάρχει και μια νέα ίσως νομοθεσία για ένα ανοιχτό σύστημα. Θα επέλυε το πρόβλημα των παράνομων χρήσεων. Τι μπορείτε να μας προτείνετε σχετικά. Είναι μία ιδέα, μια κατεύθυνση η οποία έχει αρχίσει να εξερευνάται, είτε μας αρέσει είτε όχι. Μπορεί να προκύψουν πολλές παραβιάσεις της συγκατάθεση με τη χρήση της φορητότητας. Και θα είναι πολύ δύσκολο να διερευνηθούν, καθώς και να υπάρξουν και προσφυγές. Πάντω με του καταναλωτέ και τι πληροφορίε που βάζουν στου ιστοτόπου, βλέπουμε περίπου τι βάζουν σε έναν ιστοτόπο και τι συνέπειε μπορεί να προκύψει. Όμω στο μέλλον, αυτά που κάνουν μπορεί να γυρίσουν εναντίον του. και πολύ σοβαρά. Η φορητότητα μπορεί να χρησιμοποιείται επιλεκτικά από τι πηγές τις ίδια των δεδομένων, ώστε να χρησιμοποιείται διαφορετικά για του δικαιούχου Άλλοι να έχουν περισσότερη πρόσβαση από ότι κάποιοι άλλοι ακόμα ακόμη. Οπότε ανοίγει ιδέε δυνατότητε ανταγωνισμού και είναι περισσότεροι οι φορεί που εμπλέκονται εδώ πέραν από του ελεγκτέ προσωπικών δεδομένων. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει σώματα όπω το δικό σα και θα σα δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα από 5.000 εταιρείε στο μάρκετ και την τεχνολογία στο σύστημα ITEC. Οι περισσότεροι έχουν προφίλ ε, όλων των μελών αυτή τη αίθουσα. Μπορείτε να πάτε σε όλου σα και να ζητήσετε το προφίλ σα ε, και τα στοιχεία σα. Αυτό ε, πραγματικά απογοητεύει πάρα πολύ κόσμο να βλέπουν τόσε κατηγορίε δεδομένων και να μην ξέρουν τι είναι νόμιμο και τι όχι. Αυτά τα δεδομένα όμως με τη φορητότητα θα μπορούσαν να περάσουν και σε άλλα συστήματα που να είναι με την, στο δικό σας το πλευρό. Εάν υπήρχε σωστή επιβολή κανόνων και αν μπορούσε να επιτρέψει να υπάρξουν και άλλα βιώσιμα business model από τη σωστή πλευρά. Άρα η φορητότητα είναι ένα πρόβλημα, θα μπορούσε να είναι προβληματική αν δεν πετύχουμε την επιβολή του νόμου. Και τελευταία ομιλήτρια εδώ η κυρία Κάπελ για την ΙΕΝΕΦ e και την Ήτρε. Ευχαριστώ πολύ. Ερώτηση προς την κυρία Γέλινεκ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για την εφαρμογή του βασικού κανονισμού. Είναι μεγάλη η πρόκληση. Είπατε ότι ήδη έχετε 29 υποθέσεις διαμεθοριακού χαρακτήρα που εκκρεμούν για την ερμηνεία και εφαρμογή του βασικού κανονισμού. ασφαλώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο πρότυπο. Είπατε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι διατεθειμένες να συνομιλήσουν μαζί μα για τον βασικό κανονισμό, ότι επίσης το Facebook έχει αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόσει τις διατάξεις του βασικού κανονισμού προστασίας δεδομένων. Ερώτηση. Εάν διαπιστώσετε παραβιάσεις στην εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού, θα συστήσετε την λήψη νομικών μέτρων. Επίσης, για την first conscience ή για την εξαναγκαστική συγκατάθεση. Έχετε εκεί να προτείνετε κάποια μέτρα. Η κυρία Γέλινεκ, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας κυρία Ευρωβουλευτά. Δεν πρόκειται για σύσταση ε, μέτρων, νομοθετικών μέτρων διότι ο ίδιος ο βασικός κανονισμός προβλέπει μέτρα τα, οποία όχι μόνο πρέπει να, ε, όχι μόνο μπορούμε να επιβάλλουμε και να, ε, αλλά και πρέπει να τα επιβάλλουμε και προβλέπει ε, προειδοποιήσεις και πινές οι οποίες πρέπει να είναι και αποτελεσματικές. Δεν είναι ζήτημα λοιπόν συστάσεων, είναι ζήτημα εφαρμογής του νόμου. Όπως είπατε σωστά, πρόκειται για μια ενιαία εφαρμογή του κανονισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα που επιθυμώ να απαντήσω. Το δεύτερο, το παγκόσμιο πρότυπο που αναφέρατε. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση δείχνει τον δρόμο. Υπάρχουν πολλά ενδιαφερόμενα έθνη, πολλές ενδιαφερόμενες χώρες. Διότι οι διατάξει του κανονισμού πρέπει να γίνονται σεβαστέ όχι μόνο όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, αλλά μπορεί να παίξει και τον ρόλο του παγκόσμιου προτύπου και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίω. Και όχι μόνο στην Δύση, αλλά και στην Ανατολή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Εδώ λίγη η πρώτη συνεδρία. Ευχαριστώ τις ομιλίτε και του ομιλητέ, καθώ και τα μέλη ευρωβουλευτέ. θα προχωρήσουμε αμέσω στην δεύτερη συνεδρία τις επιδράσεις στις εκλογικές διαδικασίες. Θα έλθει κοντά μας η πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών, κυρία Χούπνερ. Και θα προσέλθουν και άλλα πρόσωπα όπως η κυρία Μπάσετ, της, ε, Ευρωπαϊκής, ε, συγγνώμη, της ε, Επιτροπής Εκλογών της Μεγάλης Βρετανίας και ο κύριος Κάπλαν, αντιπρόεδρος του Global Public Policy Facebook. So, colleagues, uh, please stay with us. Αγαπητοί συνάδελφοι, μείνετε μαζί μας. Έχουμε σημαντικούς ομιλητές. Η κυρία Χούμπνερ όμως παρακαλώ πρώτα να κάνει μια σύντομη εισαγωγή, μια που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ταγματικών ε, Υποθέσεων και βέβαια ασχολείται πολύ με τα θέματα των εκλογικών διαδικασιών. Παρακαλώ. Ναι, πράγματι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να πω δύο λόγια για ζητήματα που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά για τη συζήτησή μα. Πρώτα απ' όλα, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωεκλογέ που μα έρχονται σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ακόμα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Εκλογική Επιτροπή και ελπίζω να έχουμε συμπεράσματα σύντομα όσον αφορά το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρουμε ότι όταν συμβαίνουν άσχημα πράγματα, καλό είναι να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, πώς γίνανε, γιατί και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε στο μέλλον. Επίσης, όσον αφορά τις ευρωεκλογέ του χρόνου, την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσουμε για νέους κανόνες που θα διέπουν τις επόμενες ευρωεκλογέ για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια. Και θέλω να σας πω επίσης ότι θα πιέσουμε ε, στους κανόνες αυτούς να υπάρξει δυνατότητα ε, ψηφοφορίας online, ηλεκτρονικά δηλαδή. Και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες αλλά και τους υποψηφίους ε, που θα ψηφίσουν, θα χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική αυτή ψηφοφορία όλα να είναι ασφαλή και να πάνε καλά. Οι κανόνες που θα τροποποιηθούν τώρα στον Ευρωπαϊκό Εκλογικό Νόμο θα αλλάξουν και την μορφή, την νομική και θα έχουν πλέον το βάρος ευρωπαϊκής πράξης που σημαίνει ότι επιδέχονται ε, έλεγχο και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεχομένως, που σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν περισσότερα μέσα προσφυγής στη διάθεσή τους. Έπειτα τεχνολογία εννοείται ότι αποτελεί ευχή, αλλά μπορεί να αποτελέσει και κατάρα στην περίπτωση των εκλογών. Μας ε, προσφέρουν φοβερές ευκαιρίες για να φτάσουμε στους ψηφοφόρους. Από την άλλη μεριά όμως ανοίγουν και την πόρτα σε κακόβουλους χειρισμούς από όσου αποφασίσουν να κάνουν τέτοιους χειρισμούς. Ελπίζω λοιπόν ότι ο κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων θα ε, αποτελέσει και το κατάλληλο πλαίσιο προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών, ώστε τα δικαιώματά τους και τα δεδομένα τους να τυχαίνουν προστασίας. Για να τα καταφέρουμε όμως χρειαζόμαστε συνειδητοποίηση και μεταξύ των πολιτών. Πρέπει να θέλουν να... και να ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και τι σημαίνει κάθε φορά που πατάνε ένα κλικ ε, που λέει συμφωνείτε με τους όρους χρήσης. Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να ρυθμίσουμε και να έχουμε κανόνες για το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα στις προεκλογικές εκστρατείες. Και όσοι συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να λογοδοτούν. Άρα χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια. Το πρόβλημα πιστεύω είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν περιορίζεται στην Cambridge Analytica και στο Facebook και πρέπει να λυθεί συνολικά. Γιατί αλλιώς θα ξανά έχουμε το ίδιο πρόβλημα ακόμα και αν ακούει σε διαφορετικό όνομα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χούμπνερ. Θα ακούσουμε τώρα από μια χώρα από αυτές που ακούμε ότι υπήρξαν σημαντικές επιπτώσεις. Ακούμε λοιπόν την κυρία Μπάσετ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε εδώ σήμερα. Αρχίζω υπογραμμίζοντας ποιος είναι ο ρόλος της ε, Επιτροπής Εκλογών του Ηνωμένου Βασιλείου στην προεκλογική εκστρατεία. Είναι πολύ σημαντικό το πλαίσιο τι ρόλο παίζουμε για να καταλάβουμε ποιες είναι οι σημερινές προκλήσεις. Πρόκειται για ένα κοινοβουλευτικό σώμα το οποίο δημιουργήθηκε το 2000 και βοηθάει σε περίπτωση και δημοψηφισμάτων όπως στη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκοτή κτλ. Και βοηθούμε λοιπόν στα δημοψηφίσματα αλλά και στην ε, ρύθμιση των οικονομικών ε, των διαφόρων εκλογικών διαδικασιών. Όταν το Κοινοβούλιο δημιούργησε την εκλογική αυτή επιτροπή, αποφάσισε ότι ο καλύτερο τρόπο να ρυθμιστούν οι πολιτικές εκστρατείε είναι να υπάρχουν κατάλληλοι έλεγχοι όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Με κανόνε συγκεκριμένου για τη χρηματοδότηση, για την προέλευση τη χρηματοδότηση αυτής και για το πώ τα χρήματα δαπανώνται. Έτσι λοιπόν ζητάμε και από τα πολιτικά κόμματα και από όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν αυτούς τους κανόνες. Πώς λειτουργούν τώρα οι ρυθμίσεις. Είναι σημαντικό και αυτό να το ξέρουμε. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Πρώτον, οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα πρέπει να δίνει πληροφορίες όσον αφορά την χρηματοδότηση. Και υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανόνες προεκλογικής εκστρατείας και όλα αυτά καταγράφονται, συμπεριλαμβάνονται δηλαδή σε ένα μητρό το δημοψήφισμα κάθε φορά που θα πάνε πάνω από 10.000 λίρες πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ποιοι συμμετείχαν στην χρηματοδότηση. Όσον αφορά τώρα τα δάνεια και τις δωρές. Ένας δωρητής μπορεί να είναι κάποιος ψηφοφόρος, καταγεγραμμένος ως ψηφοφόρος. Οπωσδήποτε και πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι όλες οι δωρές πρέπει να αναφέρονται από τα πολιτικά κόμματα στην προεκλογική εκστρατεία. Όλες ε, οι δαπάνες πρέπει να αναφέρονται και ελέγχονται από το Κοινοβούλιο. Είχαμε 7 εκατομμύρια για την εκστρατεία του Brexit, σε άλλες περιπτώσεις κατεβαίναμε σε 700.000. Η περίοδος αναφοράς βέβαια επηρεάζει τις δυνατότητές μας να ρυθμίζουμε τις προεκλογικές εκστρατείες. Στις γενικές εκλογές είναι άλλη περίοδος και στο δημοψήφισμα ήταν 10 εβδομάδες. έξι μήνες είχαν στη διάθεσή τους τα πολιτικά κόμματα. Τις επιστροφές φροντίζει η εκλογική επιτροπή να δίνονται στα κόμματα για τα χρήματα που έχουν δαπανήσει και προβλέπονται επιστροφές. Η εκλογική επιτροπή δεν είναι σε θέση να καλύψει το περιεχόμενο των προεκλογικών εκστρατιών. Όμως ελέγχουμε τις διάφορες δραστηριότητες ώστε να ξέρουμε ότι τα πράγματα γίνονται σωστά. Μπορεί να τοπίσουμε ε, κάτι που γίνεται από κάποιον ο οποίος δεν έχει καταγραφεί ε, ως συμμετέχον στην προκλητική εκστρατεία. Όσοι συμμετέχουν πρέπει να ενημερώνουν και τις δαπάνες τους στην προκλητική εκστρατεία και τη διάρκεια της. Και όσοι είχαν πληρώσει πριν την έναρξη της εκστρατείας. Θα πρέπει με τις δαπάνες να βλέπουμε πώς τα ποσά ε, δαπανήθηκαν με βάση συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Τους κανόνες αυτούς τους εφαρμόζουμε σε υποθέσεις που δείχνουν από την προηγούμενη περίοδο πώς όλα αυτά αναπτύχθηκαν και γιατί πρέπει να είναι αποτελεσματικά με τι ψηφιακέ εκστρατείε ιδίω. Όσοι συμμετέχουν σε προεκλογική εκστρατεία ψηφιακά μπορούν να κάνουν τα ίδια σε μεγαλύτερη κλίματα και πιο φθηνά. Πάντοτε είχαμε την ε, ε, προσέγγιση των πολιτών με φυλάδια στα σπίτια τους, στα γραμματοκιβώτια τους και τα συνθήματα, τα μηνύματα που έφταναν έτσι στους πολίτες. Σε αυτή τη φάση όλα αυτά γίνονται ψηφιακά και μπορώ να πω ότι η χρηματοδότηση των εκστρατιών ε, ε και το να γνωρίζουμε πώς έγινε αυτή, είτε είναι για, ότι πρόκειται για εκλογέ είτε για δημοψηφίσματα, είναι πολύ σημαντικό. Και η ψηφιακή διεξαγωγή εκστρατιών είχε πολύ θετικό αντίκτυπο. Επέτρεψε σε όλο και περισσότερους πολίτες να είναι μέρος του δημόσιου διαλόγου. Και είδαμε ε, επίπεδα ρεκόρ ψηφοφόρων στα, στις πρόσφατες περιπτώσεις. Όμω είναι σημαντική και η προστασία των ψηφοφόρων και είναι μέρο επιτυχών εκλογών. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε διαφάνεια και λογοδοσία για όλε τι εκστρατείες, ώστε οι ψηφοφόροι να ξέρουν τι του λέει ποιο. Πάντως πρέπει να πω ότι ήδη έχουμε αυστηρούς κανόνες οι οποίοι μπορούν να βελτιωθούν και πρέπει να βελτιωθούν για να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν. Όπως οι τωρινοί κανόνες δεν λένε πώς ε, ε, τα χρήματα δαπανώνται σε καθημερινή βάση πριν τις εκλογές. και Σημαντικό θα ήταν να μπορούμε να δούμε και τι συμφωνίε πρώτη εκστρατεία για να τα ελέγξουμε. Ας πούμε από το 2003 βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφημίσεις και ψηφιακέ και ε, έντυπε για το δημοψήφισμα. Αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να το δούμε και σε κυβερνητικό επίπεδο. Επίση, θέλουμε να δούμε βελτιώσεις στις κατηγορίες βολής εκθέσεων για τα θέματα αυτά και τη σωστή διεξαγωγή των εκλογών. Αυτή τη στιγμή οι κατηγορίε που έχουμε προβλέψει δεν δείχνουν με λεπτομέρειε πώ τι ψηφιακέ δραστηριότητε δαπανήθηκαν συγκεκριμένα ποσά. Θα χρειάζονταν λογαριασμοί και αποδείξει για να δούμε τι ακριβώ έχει γίνει. Συχνά απλώ ε, αυτά καταχωρίζονται κάτω από την κατηγορία digital consultancy, συμβουλευτική ψηφιακή και τα καλύπτει όλα. Ε, επίσης πρέπει να δούμε το δικαίωμα εκλογή αυτού που διεξαγάγει την εκστρατεία. Πάντω, το κόστο τη εκστρατεία έχει να κάνει και με το ποιοι συνεργάζονται με τον καθένα. Και επίση, τα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει να υπάρχει μια συστηματική καταγραφή όλων των δεδομένων, Όπω η πηγή ε, των ποσών του και το σε ποιου απευθύνονται. Επίση, θα πρέπει να προσφέρουμε στου προφόρου διαφάνεια, αλλά γι' αυτό πρέπει να καταγράφονται ποιοι έκαναν συγκεκριμένε δηλώσει και όχι απλώ ε, υποθετικά. Ε, η πληροφορία, οι πληροφορίε που έχει η, η εκλογική επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου στα χέρια τη ε, είναι σημαντικέ. Το να μοιραζόμαστε όμω τι αρμόδιε αρχέ και να σεβόμαστε τι αρμοδιότητε με τον ΔΕ είναι πολύ σημαντικό. Η εκλογική επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να δει πώ χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα και όπω η Ελίζαμπεθ και η ομάδα τη ε, θα τα μελετήσουν τα θέματα αυτά προσεκτικά για να δούμε πόσα χρήματα δεπανήθηκαν και πώ. Ε, με συγκεκριμένου κανόνε. Πρέπει πάντω να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να έχουμε τι σωστέ πληροφορίε και να λειτουργεί νομοθεσία. Υπάρχουν κανόνε που προβλέπουν περιορισμού στι πηγέ, όχι όμω που μπορούν να δαπανηθούν. Και πρέπει να δαπανούνται σωστά. Οι εμπειρογνώμονε και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να είναι ε, αυτοί που θα πάρουν χρήματα από όσου διεξαγάγουν εκστρατεία. Αλλά όχι σε όλε τι περιπτώσει επίση δεν έχουμε, δεν έχουμε δικαιοδοσία για αυτού που είναι εκτό Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι προβλέπει ο νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου. Κοινωνικά δίκτυα που δεν έχουν δυνατότητα στη χώρα μα δεν μπορούν να επηρεαστούν κατά τη διάρκεια τη διεξαγωγή προεκλογικών εκστρατιών. Και πολύ συχνά η διακοπή των προεκλογικών εκστρατιών, η διατάραξή του είναι μέρο προσπάθεια διατάραξη του δημοσίου βίου γενικότερα. Και τώρα για την ανάγκη να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του το κοινό των ψηφοφόρων. Πρέπει να προσέξουμε και το θέμα της ψηφιακής εκστρατεία. Βλέπουμε τα διδάγματα από τις έρευνες που έγιναν μετά την προεκλογική εκστρατεία. Είμαστε σε διάλογο με τις αρμόδιες αρχές και από το πρωί θα δημοσιοποιήσουμε και μια έκθεση για το θέμα αυτό με τις προτάσεις για αλλαγές. Ε, για το μέλλον. Αυτή θα είναι η πρώτη από τι κινήσει μα και τα πορίσματά μα, αλλά θα υπάρξει και μια σειρά από αλλαγέ, όπω αυτά που προηγουμένω ανέφερα, για να ενισχυθεί η εκλογική επιτροπή μα και δυνατότητα να επιβάλλουμε τι κορώνε που μα διέπουν. Ακόμη και ισχυρότερε κυρώσει, ε, αυστηρότερε κυρώσει. Επίση, ο νόμο μα μπορεί να μην επικεντρώνεται τόσο πολύ στα δεδομένα, αλλά ελπίζουμε ότι θέτει το σωστό πλαίσιο για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο ομιλητή. Κάπλαν, αντιπρόεδρος του Facebook. Καλώς ήλθατε. Προχωρήστε στην παρουσίασή σας. Γεια σας, ευχαριστώ τους Προέδρους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με δέχεται σήμερα εδώ. Ας μιλήσουμε για τα γεγονότα των τελευταίων μηνών και ας δούμε ποια μέτρα έχουμε λάβει ως Facebook για να προστατεύσουμε τις εκλογέ απανταχού του κόσμου. Άλλωστε είναι τιμή μου που ε, βρίσκομαι εδώ μαζί με την κυρία Μπάσετ και άλλε αρχέ που έχουν αναλάβει σχετικέ πρωτοβουλίε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή. Αρχίζω λέγοντα τα όσα είπε ο διευθυντή μα Ζούκερμπεργκ όταν ήρθε εδώ το προηγούμενο μήνα στι Βρυξέλλε. Η προστασία τη ακαιρεότητα των εκλογών εδώ στην Ευρώπη είναι για μα πρώτη στην προτεραιότητα στο Facebook. Η δέσμευσή μα για την ασφάλεια των εκλογών και την ακαιρεότητά του περιλαμβάνει και τι εθνικέ εκλογέ αλλά και τι ευρωεκλογέ που θα γίνουν τον επόμενο Μάιο. Στο Facebook πιστεύουμε απολύτως ότι η πλατφόρμα μας μπορεί να είναι μια δύναμη καλού στη δημοκρατική διαδικασία. Πιστεύουμε ακόμη ότι οι πολιτικές διαφωνίες είναι θεμητές όταν είναι όμως ειλικρινείς και ακριβείς. Βλέπουμε εδώ οι πολίτες στην Ευρώπη να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, τους, πλατφόρμα μας για να διεξαγάγουν συζητήσεις μεταξύ τους ή και με τις κυβερνήσεις τους και βλέπουμε και πολλούς policy makers όπως εσείς να χρησιμοποιείτε εργαλεία μας για να έλθουν σε άμεση επαφή με τους ψηφοφόρους κάτι που θα ήταν αδιανόητο και προ μια δεκαετία, μια δεκαετία. Έχει καταστεί σαφέ όμω τον τελευταίο 1,5 χρόνο ότι η πλατφόρμα μα μπορεί να γίνει και αντικείμενο κατάχρηση από αυτού οι οποίοι προσπαθούν να υποσκάψουν την ακαιρεότητα των εκλογών. Στι εκλογέ των ΗΠΑ το 2016. Αλλοδαποί φορεί χρησιμοποίησαν πλατφόρμες όπως το Facebook για να διασπάσουν τον κόσμο και να του εμφυσίσουν αμφιβολία και φόβο. Ανταποκριθήκαμε με μεγάλη καθυστέρηση εμείς στο Facebook και αντίθετα από ό,τι έχουμε κάνει με το, fish, με το phishing και το malware. Μπορούμε να φροντίσουμε ώστε να μην ξαναγίνουν παρόμοιε επιθέσεις στο μέλλον και αναλαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά αυτή την, την ευθύνη μα. Θέλω να επαναλάβω ήδη από την αρχή κάτι που είπε ο συνάδελφός μου προηγουμένω ότι σε ό,τι αφορά την Cambridge Analytica, οι πιο ακριβεί προφορίες που έχουμε σήμερα έω σήμερα δηλαδή είναι ότι ο Δόκτωρ Κόγκαν δεν είχε στη διάθεσή του δεδομένα άλλων μη Αμερικανών, δηλαδή περιλαμβανομένους αυτών και, και των Ευρωπαίων. Αναμένουμε την πλήρη διερεύνηση της Cambridge Analytica, την οποία θα κάνουμε μόλις μας δώσει την άδεια ο Βρετανικός ICO. Από τις ε, αμερικανικές εκλογές του 2016 έχουμε διδαχθεί σημαντικά μαθήματα σε ό,τι αφορά τη στάση μας απέναντι σε εκλογές. Έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις και σε προσωπικό και σε τεχνολογία για να δυσχεράνουμε πολύ τέτοιου είδου επιθέσει και χρησιμοποιούμε επιτυχώ τα νέα μα αυτά εργαλεία και σε πρόσφατε ευρωπαϊκέ εκλογέ στη Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Εκεί στοχεύουμε σε πέντε βασικούς τομεί Αποτροπή αλλοδαπών επιθέσεων, μείωση των ψευδών λογαριασμών, αντιμετώπιση των ψευδών επιθέσεων, των ψευδών ειδήσεων μάλλον και ενημέρωση του κοινού. Σε κάθε έναν από αυτού του τομεί θα εξηγήσω τι νοοτροπία διαθέτουμε και τι ακριβώ πρόοδο έχουμε επιτύχει ω τώρα. Πρώτο, αντιμετώπιση των λαδαπών παρεμβάσεων. Είναι η πραγματικότητα ότι σε κάθε ε, ε, εκλογή έχουμε διαφορετικέ απειλέ και βεβαίω αντιμετωπίζουμε διαφορετικού φορεί. Η ομάδα μας που ασχολείται με την ασφάλεια εξετάζει πριν από τις εκλογές συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονε και με τους κυβερνητικούς φορείς να αντιληφθούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι και απειλέ σε κάθε χώρα. Για να αντιμετωπίσουμε τι αλλοδαπέ παρεμβάσει. χρειάζεται να κάνουμε πολύ σοβαρότερες επενδύσει σε ασφάλεια. Έχουμε διπλασιάσει το προσωπικό μα που ασχολείται με θέματα ασφαλείας από 10.000 σε 20.000 πρόσωπα που χρησιμοποιούμε και επίση το machine learning και την ε, ε, τεχνητή νοημοσύνη που μα επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε δράσει που ενδεχομένως έχουν δυνατότητα να επηρεάσουν εκλογέ. Όπως ε, ιστο, ε, αλλοδαπές ιστοσελίδες που διοχετεύουν πληροφορίε. Σημαντική δραστηριότητα αυτή για μας για να αντιμετωπίσουμε τη ε, διάδοση ψευδών ειδήσεων. Πέρσι αυτά έγιναν στις δευτερεύουσες εκλογές στην πολιτεία της Αλαμπάμα. Μπορέσαμε εκεί να εντοπίσουμε σπαμ που προέρχονταν από την Μακεδονία, εννοεί την του Γουδουμού, και φαίνεται πως γινόντουσαν για, και για την αποκόμιση κέρδους. Δεύτερος τομέας είναι η αντιμετώπιση των ψευδών λογαριασμών. Πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι bad actors κρύβονται πίσω από ψευδείς ταυτότητες. Μέσα στον τελευταίο χρόνο έχουμε βελτιώσει σημαντικά την διερεύνησή του και μπλοκάρουμε εκατομμύρια ψευδεί λογαριασμού κάθε μέρα πριν προλάβουν να κάνουν κακό. Αυτό λόγω του ότι ε, χρησιμοποιούμε την μηχανική μάθηση, τη μάθηση των μηχανών δηλαδή, που μας, επιτρέπει, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιους λογαριασμούς. Τρίτος τομέας, μείωση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Βεβαίω το κοινό επιθυμεί να βλέπει ακριβεί ειδήσει στο Facebook και το ίδιο και εμεί. Έχουμε χρησιμοποιήσει διάφορου τρόπου ε, ε, και αντιμετωπίζουμε ε, τα fake news που συνήθως έχουν οικονομικά κίνητρα. Μπλοκάρουμε ιστοσελίδες που προωθούν fake news για την αποκόμιση κέρδους. Και αντιμετωπίζουμε και το λεγόμενο clickbait και sensationalism. Γνωρίζουμε ότι μόνοι μας δεν θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό αναζητούμε εταιρικέ σχέσεις για την εκπαίδευση των χρηστών μας. Από τότε που αρχίσαμε το πρόγραμμά μας Third Party Fact Checking το έχουμε επεκτείνει σε 14 χώρες και μέχρι τέλος του έτους θα το επεκτείνουμε και σε άλλες χώρες. Πρόκειται για πιστοποιημένους ε, φορείς οι οποίοι διαρευνούν την αλήθεια των ειδήσεων και μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε την διάδοση ψευδών ειδήσεων και το έχουμε καταφέρει τώρα αυτό στα 80%. Επιπροσθέτως, προωθούμε και την εκπαίδευση των χρηστών μας δίνουμε ε, τρόπους, γνωστοποιούμε τρόπους για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων και αυτό το κάνουμε και μέσα στο facebook σε όλη την ε, παντού. Επίσης, προώθηση της διαφάνειας. Εμείς θεωρούμε ότι ο κόσμος πρέπει να αντιλαμβάνεται ποιος πληρώνει τις διαφημίσεις, ποιες άλλες διαφημίσεις προωθεί ο ίδιος διαφημιστής και αυτό ισχύει βεβαίως ιδίως για πολιτικές διαφημίσεις. Έχουμε κάνει πολλά βήματα τους τελευταίους μήνες και έχουμε δημιουργήσει και ένα νέο εργαλείο που λέγεται View Ads που σας επιτρέπει να εξετάσετε όλες τις διαφημίσεις και τα μηνύματα που προωθεί ένας συγκεκριμένος διαφημιστής. Είτε εσείς λαμβάνετε τη διαφήμιση, είτε ε, παρακολουθείτε τη σελίδα. Ε, έτσι χρησιμοποιούμε πολύ, ε, εξασφαλίζουμε πολύ καλύτερη διαφάνεια. Η εφαρμογή αυτή θα είναι παγκόσμια ισχύω σύντομα. Τέλος, η εμπλοκή μας με την κοινωνία των πολιτών. Η Συζητήσει η διαφωνία μέσα ε, στην πολιτική είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε. Διότι θέλουμε ενήμερο κοινό. Έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Megaphone και στο οποίο καλούμε το κοινό να συμμετέχει στις εκλογές και έχουμε έτσι βελτιώσει τη συμμετοχή των εκλογέων. Δημιουργούμε επίση προϊόντα που βοηθούν τον κόσμο να αντιληφθεί καλύτερα το νόημα των ψηφοδελτίων και τα προγράμματα των κομμάτων. Πριν από τις γαλλικές και τις βρετανικές εκλογές, επιτρέπουμε με τα εργαλεία μας στον κόσμο να, να αντιληφθούν καλύτερα το μήνυμα των κομμάτων. Δημιουργούμε και διαδικασίες μάθησης για πολιτικούς, για το προσωπικό των γραφείων τους κτλ. για να δουν πώς μπορεί να γίνει η κατάχρηση των λογαριασμών και πώ μπορεί να βελτιωθεί η ασφάλεια στη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατιών. Δίνουμε προτεραιότητα σε όλα αυτά, σε όλο το Facebook. Γνωρίζουμε όμω ότι η προστασία τη δημοκρατική διαδικασία είναι μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει συνολικά. Δεν αρκεί μια επιχείρηση ή ένα κλάδο τη οικονομία. Χρειάζεται συνεργασία με κυβερνητικού φορεί, με πανεπιστήμια και ούτε καθεξής, για να γίνουν αντιληπτέ οι συγκεκριμένε μοναδικέ απειλέ σε κάθε χώρα. Στι γερμανικέ εκλογέ πέρσι συνεργαστήκαμε από κοντά με το Ομοσπονδιακό ε, Γραφείο Προστασία τη Προφορίας, BSI, πριν από τις Ιταλικέ εκλογέ του Μαρτίου συνεργαστήκαμε στενά με τον Ιταλό νομοθέτη για να δημιουργήσουμε κατευθυντήρε γραμμέ για το πώ θα χρησιμοποιούν οι πολιτικοί τα επιγραμμικά εργαλεία και να διοχετεύσουμε τι προφορίες αυτέ στο διαδίκτυο. Και τέλο, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ, φροντίσαμε το πλήθο των ε, παρατηρητών ΟΑΣΕ να μπορεί να έχει στη διάθεση τι αναγκαίε πληροφορίε. Συνεργαζόμαστε συχνά και με εξωτερικούς φορείς, με το Ατλαντικό Συμβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες και με το αρμόδιο εργαστήριό του, το οποίο σε συνεργασία με τις δικέ μας ομάδες δίνει άμεσε πληροφορίες στο διαδίκτυο για αναφιόμενε απειλέ. Σημαντική και ισχυρή εταιρική σχέση για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουμε χρήση του δικτύου μα. Τέλος, τον Απρίλιο ξεκινήσαμε νέα πρωτοβουλία για την αξιολόγηση του ρόλου των social media στις εκλογές που θα επιτρέψει στο Facebook να, ε, να διδαχθεί από αναλύσεις πανεπιστημιακών ώστε να μπορέσουμε να λαμβάνουμε καλύτερες και ταχύτερα αποφάσεις. Η προστασία της ακαιρότητας των εκλογών ποτέ δεν θα λύθει ως πρόβλημα. Ως φορέας και ως κλάδος αντιλαμβανόμαστε ποιες είναι οι απειλές. Έχουμε επιθέσεις από φορείς που είναι όλο και ισχυρότεροι. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε απόλυτα την ακυρότητα των εκλογών, μπορούμε όμως να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας. Και συνεργαζόμαστε με πολιτικά κόμματα, με ε, τους νομοθέτες, με τις κυβερνήσεις και με τους πανεπιστημιακούς φορείς για να αυξήσουμε τη συνεργασία αυτή μεταξύ αυτών και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα πράξουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε την ακυρότητα των επικειμένων ευρωεκλογών. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Να πάμε τώρα αμέσως στις ερωτήσεις, για τις οποίες έχετε ένα λεπτό και δύο λεπτά για τις απαντήσεις. τανούτα Χύπνερ πρώτη. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Πάσετ. Η περίπτωση αυτή που μας έχει φέρει και εδώ σήμερα ε, κυκλοφόρησε πολύ στον τύπο, στα μέσα ενημέρωσης παντού. Μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ψηφιοποίηση. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχει και αρνητικέ επιπτώσει στη συμμετοχή των πολιτών στι επόμενε εκλογέ. Πιστεύετε πω υπάρχει τέτοια περίπτωση, ναι ή όχι. Καλή ερώτηση θα έλεγα, λέει η κυρία Μπάσετ. Το πρώτο που πρέπει να θυμόμαστε για όλα αυτά είναι ότι μπορεί κανείς να πει ό,τι θέλει για το τι κάνει, τι δεν κάνει ο κόσμος, τι νομίζουμε κτλ. Αλλά η σχέση αυτών με τις αποφάσεις του κόσμου να αποφασίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε έρευνες που δείχνουν πως δεν έχουν δεδομένα οι ανεξάρτητοι ερευνητές για να το ξέρουν. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην ε, βιαζόμαστε και να νοπίζουμε να νομίζουμε ότι οι άνθρωποι που έκαναν πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν έχουν τόσο μεγάλη εξουσία στα χέρια του. Αυτό που κάνουμε εμεί στην Εκλογική Επιτροπή με τι έρευνέ μα είναι ότι κάνουμε έρευνε στην ε, κοινή γνώμη για να δούμε ποια είναι η συμπεριφορά του απέναντι στα ψηφιακά, στην ψηφιακή τεχνολογία. Και σίγουρα υπάρχει μεγάλη επιθυμία οι άνθρωποι να παίξουν πιο ενεργό ρόλο. Χρειάζεται συνειδητοποίηση και είναι ένα ευρύτερο θέμα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη συμμετοχή στις εκλογές. Ο κόσμος αρχίζει επικριτικά να τα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα ζητήματα και είναι θετικό. Να αναρωτιέται πολύ περισσότερο ε, για τον ε, ψηφιακό του περίγυρο. Το και πριν ότι έχουμε δει ρεκόρ συμμετοχή στις εκλογές. Το είδαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και μεταξύ των νέων κυρίως υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή. Οπότε δεν θα έλεγα ότι θα πάει προς τα κάτω η συμμετοχή. Πρόεδρος, εγώ εκ μέρους των ε, σοσιαλιστών. Θα ήθελα να πάμε περισσότερο σε βάθος όσον αφορά την ανάμειξη στις εκλογές μας. Υπήρχε έκθεση πρόσφατα που έλεγε ότι προσλάβατε ως προσωπικό τέος ερευνητές των υπηρεσιών ε, πληροφοριών. Πώς όλα αυτά επηρεάζουν την ε, ανάμειξη που κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπήρξε στις εκλογές, είτε αυτή είναι ρωσική ή σε άλλες εκλογές. Για πείτε μας με δύο λόγια. Τι προκύπτει από όλα αυτά. Ευχαριστώ. Είναι στην καρδιά του ζητήματος αυτή η ερώτηση. Πρόκειται για ένα άρθρο πράγματι που λέει τι πόροι χρησιμοποιήθηκαν από τις ομάδες μας για να έχουμε πραγματογνωμοσύνη για το πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε σε σχέση με τις εκλογές παγκοσμίως. Πρέπει να έχουμε αυτή την ικανότητα, αλλά όπως είπα και στην αρχή, επίσης θέλουμε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες επιτόπου στις χώρες όπου γίνονται οι εκλογές. Οπότε πρέπει να έχουμε αρκετό προσωπικό για συνεργασία με τις εκλογικές επιτροπές κλπ. Πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι απειλές που προκύπτουν σε κάθε χώρα. Δεν είχαμε αναπτύξει πλήρω τις δυνατότητές μας αυτές το 2006 για τις αμερικανικές εκλογές και μάθαμε πολλά για το εύρος εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιούμε στην περίπτωση εκλογών. Όσο προχωράμε με διάφορες εκλογές και χρησιμοποιούμε τις ομάδες μας σε συνεργασία και χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να εντοπίσουμε τους ψεύτικους λογαριασμούς, τις ε, ε, παρεμβάσεις, την έλλειψη διαφάνειας ε, και λοιπόν και λοιπά. Όλα αυτά τα μέσα λοιπόν θα τα χρησιμοποιούμε για κάθε εκλογική διαδικασία. Χρησιμοποιούμε την εμπειρία που αποκτήσαμε τους τελευταίους μήνες, είδαμε με τις γαλλικές εκλογές που 30 τόσες χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς κατεβάσαμε πριν από τις εκλογές ή στις γερμανικές εκλογές όπου συνεργαστήκαμε στενά με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια. Ή αλλού που πάλι συνεργαστήκαμε για ελέγχους ώστε να μην υπάρχουν ε, ψευδείς ειδήσει. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας σε κάθε εκλογική διαδικασία και το κάνουμε. Ευχαριστούμε κύριο Ζοντόφσκι. ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. που μου δίνετε το λόγο πρώτα απ' όλα και σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ, κύριε Κάπλαν. Περιμέναμε βέβαια και άλλους ανώτερους, αλλά εντάξει, μας ικανοποιεί δικιά σας παρουσία σήμερα. Είπατε ότι το Facebook αποτελεί δημοκρατική πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών. Ναι, αλλά πώς μπορώ εγώ να έχω εμπιστοσύνη σε μια εμπιστοσύνη η οποία χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο για να κλείσει ψεύτικους λογαριασμούς οι οποίοι εμφανίζονται σαν είμαι εγώ που χρησιμοποιούν τη δικιά μου τη φωτογραφία. Τι κάνετε για να σταματήσετε μια τέτοια κατάσταση ώστε να μην επαναλαμβάνονται αυτοί οι ψεύτικοι λογαριασμοί. Και και η Bridge Analytica φάνηκε ότι επηρέασε την εκλογική διαδικασία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και στην Τσεχία μάλιστα. Ο συνάδελφός σας είπε κάτι μόνο για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Όταν πήγαμε στο Facebook όλοι είπαν ότι είσαστε μια εταιρεία κοινωνικά υπεύθυνη. Κάνετε πράγματι τα πάντα ώστε να σας πιστέψουμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Απαντήστε μας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Όσον αφορά τους ψεύτικους λογαριασμούς, είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, αλλά έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ τεχνολογική έρευνα σε αυτό και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Όπως είπε και ο συνάδελφος στο προηγούμενο πάνελ, τώρα φερούμε εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς, τους μπλοκάρουμε ώστε να μην ε, καταγραφούν πριν καν μπορέσει κανείς να τους δει αυτούς τους ψεύτικους λογαριασμούς. 500 εκατομμύρια πρόσφατα. Άρα λοιπόν αναλαμβάνουμε δράση και κατά τη γνώμη μου δεν θα λυθεί ποτέ πλήρως το παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά και συνεχίζουμε να επενδύουμε και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε νέα τεχνολογία και νέες εφαρμογές για να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή. Αυτό κάνουμε, γι' αυτό και διπλωσιάσαμε τους ανθρώπους που δουλεύουν για την ασφάλεια σε εμά. Όσον αφορά την επιρροή της Cambridge Analytica σε άλλες εκλογικές διαδικασίες στην Ευρώπη, θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή και που είπε και ο κύριος Σάτερφιντ νωρίτερα, ότι οι καλύτερες πληροφορίε που έχουμε σήμερα είναι ότι τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών δεν δόθηκαν στην Cambridge Analytica. Οπότε δεν βλέπω πώς θα μπορούσε η Cambridge Analytica να έχει επηρεάσει εκλογές διαδικασίε στην Ευρώπη. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο δεδομένο για να πιστέψουμε αυτό. Φυσικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει να γίνει εξωτερικός έλεγχος, γιατί στο κάτω-κάτω μόνο η Cambridge Analytica η ίδια γνωρίζει τι ακριβώς έκανε. Τέλος για το τελευταίο που ρωτήσατε αν είμαστε κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεσή μας. Και όπως είπε και ο κύριος Σάτεφιλτ νωρίτερα, ε, στο τέλο δεν έχει σημασία αν εγώ ή κάποιος άλλος λέει ότι είμαστε κοινωνικά υπεύθυνοι ή όχι. Αυτό που παίζει ρόλο είναι εσείς να συμπεράνετε από τη δράση μα ότι όντω κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και για να αντιμετωπίσουμε ό,τι προβλήματα διαπιστώνουμε με καταχρήσεις στην πλατφόρμα μας. Εσείς πρέπει να πιστείτε γι' αυτό. Η Mercedes Μπρέσο για την ΑΦΚΟ και τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να επανέλθω σε αυτό που υπόθηκε 500, εκατομμύρια λογαριασμοί σε λίγους μήνες με παράνομη χρήση. Μήπως πρέπει να φτάσουμε στην ψηφιακή ταυτότητα, την προσωπική ψηφιακή ταυτότητα, λόγω χάρη στην Εστονία, για να μπορεί κανείς να κάνει σχόλιο σε online εφημερίδα, πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δική του ηλεκτρονική ταυτότητα, πράγμα που πιστοποιεί το ποιος είναι ποιος. Αυτό θα έπρεπε να γίνει όχι στο επίπεδο μια χώρα μόνο, αλλά να κοιτάξουμε να δημιουργήσουμε μια ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτό θα διευκόλυνε πολύ τα πράγματα ίσω. Διότι λέτε 500 εκατομμύρια, αλλά το πρόβλημα είναι πόσοι ήταν οι λογαριασμοί τελικά. Ε? Πόσα εκατομμύρια πιστεύετε ότι μπορεί να σας διέφυγαν. Και μετά έχω και άλλη μια ερώτηση, αλλά θα την κάνω μετά. «500 εκατομμύρια καταγράψαμε στο πρώτο τρίμηνο. Ένα από τα πράγματα που κάναμε πρόσφατα για να δείξουμε την αφοσίωσή μας είναι ότι δημοσίευσαμε περισσότερα δεδομένα, περισσότερα στοιχεία για το πόσε ε, παραβιάσεις και προνομές κρίσεις εντοπίσαμε στο Facebook και μπορέσαμε να προσφύγουμε εναντίον τους. Η εκτίμησή μα σε σχέση με την ετήσια έκθεση είναι ότι είναι, υπάρχουν 3-4% ε, λογαριασμοί που είναι ψεύτικοι. Μεγάλο αριθμό είναι αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο στη διάθεσή μα για να του αποκρούσουμε. Τεχνητή νοημοσύνη, ε, το machine loading, Προωρούμε να δούμε από τη συμπεριφορά των ε, λογαριασμών και του πώς κινούνται, αν είναι ψεύτικοι ή όχι. Δεν είναι πραγματικός άνθρωπος πίσω του. Το θέμα της ψηφιακή ταυτότητας για όλους. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο κόσμο στι διαφορετικέ χώρε, οι πολιτικοί ηθήνοντε και όσοι χαράζουν πολιτική μπορούν να έχουν διαφορετικέ απόψει για τη σοφία, τη σύνεση και την ε, σκοπιμότητα ενό τέτοιου μέτρου πάλι ανακύπτουν ζητήματα όπως αυτά που σχολιάζουμε σήμερα για τα δεδομένα και την προστασία των δεδομένων αλλά όταν μιλάμε για πραγματική πιστοποίηση κάποιου στο διαδίκτυο αυτό έχει ζητήματα. Και θα απασχολήσει πολύ τι κυβερνήσει ποιο είναι ο σωστό τρόπο να το κάνουμε. Όταν έχουμε μια υποψία ότι κάποιο λογαριασμό είναι ψεύτικο, πολλέ φορέ θα τον περάσουμε από ένα checkpoint, δηλαδή θα τον μπλοκάρουμε από την περαιτέρω πρόσβαση στο Facebook, εκτό και να μα δείξει μια ταυτότητα και ταυτοποιήσει κάπω τον εαυτό μου για να δούμε ότι είναι το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι. Αλλά προτιμάμε να κινούμαστε βάσει των υποψιών μα αυτή τη στιγμή αντί να ζητάμε από όλου του χρήστε επισήμω μια ταυτότητα. De facto. Ο κύριο Σέφλιν, παρακαλώ, από το ΕΛΚ και την ΑΦΚΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι πραγματικά έχω εκπλαγεί ιδιαίτερος από όσα ακούω με, την, με το καθεστώς ασφάλειας στην ψηφιοποίηση. Όπως είπε ο κ. Κάπλαν, ποτέ θα λυθεί πλήρως το πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν κάποιο μέλλον για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Κύριε Κάπλαν, θέλετε μήπως να πείτε κάτι για τις ουγγρικές εκλογές. Όταν λέω δεν θα λυθεί ποτέ πλήρω το πρόβλημα, νομίζω ότι είναι σαφή αποτίμηση τη μάχη που κάθε εταιρεία που κινείται στο διαδίκτυο και κάθε φορέα επιβολή του νόμου έχει να κάνει κατά τη εγκληματική δραστηριότητα και των δόλειων ε, χρηστών, το τομέα των ψηφιακών κυρίω. Έχουμε αντιπάλου που και χρήμα έχουν και προηγμένα μέσα και θα συνεχίσουν να ε, ε, χρησιμοποιούν τι πιο εξελιγμένε τεχνικέ και δυνατότητες. Εμείς λοιπόν ως Facebook και ως αρχές και φορείς επιβολής του νόμου ανά τον κόσμο θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και εμείς πολύ προηγμένα μέσα και εργαλεία για να μείνουμε ένα βήμα μπροστά τους αν γίνεται. Αυτή είναι αφοσίωσή μας. Επενδύουμε τεράστιους πόρους ως προς το προσωπικό που προσλαμβάνουμε, την τεχνολογία στην οποία επενδύουμε, τους ε, ε, τρόπους που Βέβαια μπορεί να, έχουν, ε, να πλήξουν και τα δική μας κερδοφορία, αλλά πρέπει να προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερη προστασία σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ηλεκτρονική διεξαγωγή εκλογών. Αυτή την υπηρεσία δεν την προσφέρουμε στο Facebook, πρέπει να το κάνουν μόνο του οι κυβερνήσεις. Εκείνες να σκεφτούν αν μπορούν να έχουν το απαραίτητο ε, επίπεδο ασφαλεία για να γίνουν ηλεκτρονικέ εκλογέ. Τώρα το να συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι στι εκλογέ και περισσότεροι να ψηφίζουν, αυτό να το επιδιώξουν οι κυβερνήσει. Νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν, αλλά θα εξαρτηθεί και από το επίπεδο εμπιστοσύνη τη υπηρεσία που θα προσφέρονται. Ο κύριο Σίλβα Περέιρα για, την, για του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε και την ΑΦΚΟ. Για τον κύριο Κάπλαν πάλι. Μετά την υπόθεση Cambridge Analytica, το σκάνδαλο αυτό είναι σαφέ ότι αναγνωρίσατε ότι υπήρξε σοβαρή παραβίαση τη σχέση εμπιστοσύνη και πρέπει να αναλάβετε περισσότερη δράση. Αναγνωρίζουμε τι προσπαθίε σα. Όμω η ερώτησή μου είναι, έχετε πλήρη επίγνωση της μαζικής χρήσης της πλατφόρμας σα ανά τον κόσμο για να διαδοθούν τεράστια κύματα ψευδών πληροφοριών και αντιδραστικές εκστρατείε πολιτικής σκοπιμότητας να εξαπλώνονται παντού. Διότι η ερώτησή μου είναι τόσο μπορείτε να κάνετε ή μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι αυτό που κάνετε απλώς δεν αρκεί. Μπροστά στον όγκο του φαινομένου που αντιμετωπίζουμε, του προβλήματος. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, έχουμε επίγνωση και έχουμε όλο και μεγαλύτερη του τελευταίου 18 μήνε για το τι είδου απειλέ κατά των εκλογών ε, μπορεί να αντιμετωπίζουμε. Ιδίω από τι ψευδέ ειδήσει και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Και έχουμε αναλάβει πολλά σημαντικά βήματα, ξεκινώντα ε, με την κατάργηση των ψευδών λογαριασμών που σα προανέφερα και που πολύ συχνά είναι υπεύθυνοι για πολλέ από τι ψευδεί πληροφορίε που διαδίδονται στο Facebook. Εδώ έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο ε, Επίση, καταργούμε τα χρηματοδοτικά κίνητρα αν μπορούμε. Πολλοί από το περιεχόμενο που βλέπουμε με την παραπληροφόρηση και διαδέτε στο facebook ε, δεν είναι σαφές ότι έχει πολιτική σκοπιμότητα γιατί αγγίζει πολιτικά θέματα αλλά πολλέ φορές αυτοί είναι και σπάμερ που βγάζουν χρήματα και με email ε, καταφέρνουν να περάσουν σε άλλη πλατφόρμα. Προσπαθούμε λοιπόν να τους ε, απομακρύνουμε για να μην κερδίζουν τίποτα από το Facebook, να πάνε στην άλλη τους πλατφόρμα και να κάνουν ό,τι εκεί, ε, να κάνουν εκεί ό,τι θέλουν. Έχουμε και εδώ μεγάλη επιτυχία, έχουμε αλλάξει τους αλγορίθμους μας για να μην προάγουμε τον αισθησιασμό και τις προκλητικές ειδήσει, αλλά να προάγουμε τις πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές και με πολλούς αξιόπιστους συλλεκτές δεδομένων από τον κόσμο έχουμε αναλύσει το περιεχόμενο του Facebook για να δούμε αν είναι ψευδές ή όχι. Τότε να λαμβάνουμε αμέσω δράση, φροντίζοντα να μην εξαπλωθεί και να μην διαδοθεί. Έχουμε κάνει λοιπόν τεράστιε προσπάθειε το τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου, από τι εκλογέ ε, στη ΣΥΠΑ το 2016. Ξέρουμε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά. Πρέπει να συνεργαστούμε με κυβερνήσει, εμπειρογνώμονε, πανεπιστημιακού, αλλά πρόοδο έχει γίνει σε πολλές από τι μεγάλες εκλογές, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, είδαμε ότι τα βήματα που αναλάβαμε είχαν και αποτέλεσμα στο να βελτιωθεί η προστασία αυτών των εκλογών. Και για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από το τόσο και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε Κάλα καλά από το, την Άλντα και την Ήτρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Μιλάτε για το πώς θα εντοπίζεται η παράνομη χρήση η... στις εκλογές, η παράνομη χρήση δεδομένων ή παραπληροφόρηση. Η Ιταλία, Γερμανία, ε, Γαλλία λόγω χάρη. Όμως τι γίνεται με τις μικρότερες χώρες. Εγώ έρχομαι από μια μικρή χώρα. Ένα εκατομμύριο κόσμος μιλάει τη γλώσσα μας. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι και εκεί προσπαθείτε να εντοπίσετε τις ε, κακοχρησίες ή είμαστε πολύ μικροί για σας. Γιατί και εμείς έχουμε εκλογές και έχουμε ένα γείτονα που οπωσδήποτε ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα των εκλογών μας. Και ο κόσμος στη χώρα μας ενδιαφέρεται για το Facebook και το χρησιμοποιεί. Ποια είναι λοιπόν η απάντησή σας για τις μικρότερες χώρες. Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά ζωτική σημασία η ερώτηση. Ξέρουμε ότι οι κοινοβουλευτικέ εκλογέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη πρόκληση διότι θα ψηφίσουν ταυτόχρονα 27 χώρε. Ε, μια, σειρά από τα, μια σειρά από εργαλεία από αυτά που περιέγραψα δεν επικεντρώνονται καθόλου στο σε τη γλώσσα είναι γραμμένα τα σχόλια. Οι ψευδείς λογαριασμοί που χρησιμοποιούμε ε, και τα εργαλεία μας βασίζονται στη συμπεριφορά του κατόχου του λογαριασμού. Το πώς ε, κινείται στο Facebook. Δεν μας απασχολεί το γλωσσικό κομμάτι του λογαριασμού, σε τι γλώσσα εκφράζεται. Το ίδιο και τα χρηματικά, τα οικονομικά κίνητρα. Δεν χρειάζεται να δούμε αν οι σελίδες και αυτά τα περιεχόμενα ε, μπορεί να μάλλον ε, κοιτάζουμε αν προσελκύουν διαφημιστικό περιεχόμενο, ε, περιεχόμενο που έχει σχέση με οικονομικό κέρδος. Και έχουμε και τις δημόσιες αναγγελίες και το σχετικό περιεχόμενο, το οποίο μπορούμε να το δούμε σε διάφορες χώρες και να συνεργαστούμε και εκεί σε με εκλογικές επιτροπές και σε πολύ μικρές χώρες, για να δούμε αν στη διεξαγωγή των εκλογών ε, οι ψηφοφόροι βγάζουν νόημα και μπορούν να ε, κρίνουν το περιεχόμενο που βρίσκουν στο Facebook. Ευχαριστούμε Γκόμε, S&D και Λίμπε. Κύριε Μπάσετ, βρήκατε αποδεκτικά στοιχεία για παρέμβαση στι βρετανικέ εκλογέ μεταξύ των οποίων του δημοψηφίσματο μέσω τη Cambridge Analytica, τη ε, περιορισμένη ευθύνη εταιρεία και άλλων παρόμοιων που να έχουν σχέση με άλλες εταιρείες όπως η Henley Partners ή άλλες λογιστικές εταιρείες και οι οποίες βάσει της ηθαγένειας και της κατοικίας και των σχετικών θεωρήσεων που δίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρούν τις κυβερνήσεις να το λάβουν αυτό υπόψη Τι μέτρα μπορείτε να αναλάβετε ώστε οι δημοσιογράφοι κατά των οποίων προσέφηγαν τέτοιου είδους εταιρείες θα πάψουν να είναι θύματα εκφοβισμού. Και θέλω και τον κύριο Κάπλα να ρωτήσω κάτι. Όχι, όχι. Η Cambridge Analytica από αφέλεια, δεξιότητα, πληστία, ε, δολιότητα τα έκανε όσο έκανε. Πήρατε δύο ερωτήσει πάλι. Θα απαντήσω στη δικιά μου. Θα πω αυτό που είπα στην αρχή. Το γεγονό ότι Cambridge Analytica και άλλε εταιρείε ήταν πάροχοι υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των εκλογών ήταν κάτι το νόμιμο βάσει του εκλογικού νόμου. Δεν ερευνήσαμε πέραν αυτού εάν οι συμμετέχοντες ε, κατέγραφαν σωστά τα όσα δαπάνησαν για τι εταιρείε αυτέ. Υπάρχουν άλλε έρευνε που τρέχουν για το παραδεκτόν σε δωρές. Αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω για έρευνες εν εξελίξη. Μόνο για αυτές που έχουμε ήδη ολοκληρώσει. Και δείχνουν ότι οι συζητήσεις υπήρξαν, αλλά σωστά είχαν καταγραφεί. Για τις προσφυγές κατά των δημοσιογράφων αυτό είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της Εκλογικής μας Επιτροπής. Οπότε δεν είναι δικός μας ο ρόλος να διερευνήσουμε την συμπεριφορά μεγάλων οργανισμών ως προς τους δημοσιογράφους και εκτός των χρονικών ορίων των εκλογών. Δεν έχουμε τις αρμοδιότητες για να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστούμε ο κύριο Άντερσον για τους Πρασίνους και την ΑΦΚΟ. Ευχαριστώ. Το δημοψήφισμα του Brexit επέφερε μια τεράστια αλλαγή, αλλά μόνο με ένα περιθώριο 4%. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι διεξήχθη νομίμως το Facebook έχει πληροφορίες που μας επέτρεπε να το συμπεράνουμε αυτό, αλλά μέχρι τώρα δεν τις έχει ε, παραδώσει. Δεν έχει δώσει το σχετικό υλικό στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν αποδείξεις ότι δημιουργήθηκαν ε, προφίλ ε, περιθωριακών ψηφοφόρων που βομβάρδιζαν τους υπόλοιπους κάνοντας πίσω κεφάλαιο υπέρ του ΛΙΒ και της ε, αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της προλογικής εκστρατείας. Μαζί με όλη τη διαφήμιση που πουλήθηκε τότε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν το δημοψήφισμα και έξι μήνες πριν την προφορία δεν πρέπει να έχετε συγκεντρωμένες αυτές τις πληροφορίε και να τις παραδώσετε στους αρμοδίους ώστε και οι χρήστε και οι ερευνητές για μελλοντικέ εκστρατείε να είναι προστατευμένοι, να ξέρουμε τι δαπανήθηκε από ποιον, για ποιο σκοπό και βάση δεδομένων. Ευχαριστώ. Thanks for the question. Um... Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Έχουμε απαντήσει ένα τεράστιο αριθμό ερωτήσεων από τη Βρετανική Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Στείλαμε και τον αξιωματούχο μας να μαρτυρήσει επί τέσσερις ώρες, ερωτήσεις επί ερωτήσεων. Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στην αρμόδια Βρετανική Κοινοβουλευτική Επιτροπή στην προσπάθεια που κάνει να διερευνήσει Ποιε ε, ήταν οι πτυχές γύρω από το Brexit. Συμφωνούμε ότι υπάρχει πραγματική αξία στη διαφάνεια γύρω από τις ε, διαφημίσεις ή τις αγγελίες και θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε εργαλεία που θα επιτρέπουν στο κοινό να βλέπει ποιον στοχεύουν οι διάφορες διαφημίσεις αγγελίες που έχουμε ξεκινήσει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένουμε να το κάνουμε το ίδιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος και να δημιουργήσουμε εργαλεία που θα επιτρέπουν στο κοινό να κατανοεί γιατί βλέπει άρα για την διαφήμιση, πού βλέπει στην οθόνη του εκείνη την ώρα και άλλον, ε, σε ποιον άλλον έχει φτάσει η διαφήμιση έχοντας, για να δώσουμε τώρα όλες τις αναδρομικές προφορίες για όλες τις διαφημίσεις που έχουν και σε όλους όσοι συμμετείχαν στις εκλογές, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό έχοντας αναλάβει δεσμεύσεις για την προστασία της προσωπικής σφαίρας των Χριστών. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό ειδοποιώντας όλους πρώτα. Έχουμε δώσει πληροφορίες σχετικά με οποιασδήποτε διαφημίσεις σχετικές με τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό βρήκαμε ελάχιστες σχετικές προφορίες και από ρωσικούς φορείς πριν από το Βρετανικό δημοψήφισμα. Εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε και να παρέχουμε όσο δυνατόν περισσότερες προφορίες στην αρμόδια Βρετανική Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η κυρία Μπρέσο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Ερώτηση για την κυρία Μπάσετ. Μετά την... Με ακούτε? Μετά την ανακάλυψη της χρήσης, ε, υπεξαίρεσης δεδομένων και παράνομες χρήσεις τους από την Cambridge Analytica για τους χρήστες του Facebook θεωρείται ότι μέσω εκλογικών ε, νόμων, κανόνων μπορούμε να αρχίσουμε να περιορίζουμε αυτές τις πρακτικές που είναι υψηλού κινδύνου. Είναι σαν μια γέλη λύκων που ε, κάνει έφοδο τους πιο ευάλωτους στα εύκολα θύματα. Εδώ τα προφίλ των ψηφοφόρων βλέπουμε ότι είναι τόσο ευπαθή που είναι λες και υπάρχουν ε, οι επιτίδοι λύκοι που κανονίζουν τι θα κάνουν. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε γι' αυτό με βάση κάποιον εκλογικό νόμο. Ε, thank you. I mean, I think... Ευχαριστώ. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Το είπα όμως προηγουμένως. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι καμία οργάνωση μόνη της είτε είναι ρυθμιστή είτε στην κυβέρνηση δεν μπορεί να το λύσει μόνη της το πρόβλημα. Εάν επιτεθούμε σε έναν τομέα και ασχοληθούμε με αυτόν, θα μετακινηθεί σε έναν άλλον το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να το δούμε σφαιρικά. Νομίζω η λύση για την καλή νομοθεσία είναι να έχουμε πραγματικά ισχυρούς ελέγχους δεδομένων. Η παρακολούθηση να εφαρμόζεται σωστά. Οι αλλαγέ που είδαμε στη Βρετανική κυβέρνηση πρόσφατα ήταν πολύ θετικέ. Πρέπει όμως οι σχετικοί κανόνες για τις εκλογές να υπάρξουν σύντομα με ενισχυμένες αρμοδότητες για την εκλογική επιτροπή. Και πληροφορίες να μπορούμε να πάρουμε όχι μόνο από όσους συμμετέχουν στην εκστατεία, αλλά ε, να μπορούμε να ζητήσουμε δεδομένα και από άλλες πηγές. Να έχουμε δηλαδή ισχυρότερη εντολή. Και μετά τη δυνατότητα να ε, ανακόψουμε τη δράση κάποιων όταν έχουμε την υποψία ότι παραβιάζουν τον νόμο. Ακούγοντα τίποτα από αυτά, μάλλον δεν είναι τίποτα τόσο κλονιστικό, ούτε είναι κάποια φανταστική αποκάλυψη. Αλλά πρέπει οι εταιρείε κοινωνικών δικτύων να αναλάβουν ευθύνη. Να ακολουθούν αυστηρό του κανόνε του και οι ρυθμιστέ να έχουν τι δυνατότητε να τα επιβάλλουν με κυρώσει, εάν προκύψουν παραβιάσει. Αυτό ζητούμε. Η κυρία Έρνστ για την ΚΟΕ e και την Ήτρα. Ε, Ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλά σχετικά με τα όσα έχετε αναλάβει και κάνετε ως Facebook. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό που είπε η Βρετανίδα συναδελφό σας. Έχω την ερώτηση τώρα. Πώς διακρίνετε απλά διαφήμιση προϊόντων από την πολιτική διαφήμιση. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, πώς ε, την εννοείτε αυτή τη διαφήμιση και ποιε διαφορέ υπάρχουν κατά την άποψή σα, Υπάρχει ε, προεκλογική διαφήμιση, επανέρχομαι στην τηλεόραση, όπου ισχύουν κάποιοι κανόνε, αναλογικότητα σχετικά με τη δύναμη των κομμάτων κτλ. Μπορείτε να φανταστείτε εφαρμογή παρόμοιων κανόνων ανεπροχημένο. Και εδώ συμπληρώνω την εξή ερώτηση. Χειραγώγηση εκλογών, κάτι για το οποίο μιλούμε τόσο πολύ. Θέλω να μάθω χειραγώγηση εκλογών, ναι, αυτό σημαίνει και τα fake news. Αλλά στο αφήσουμε αυτό για την ώρα. Τι σημαίνει για σας χειραγώγηση εκλογών, από ποιο σημείο και μετά αρχίζει και πώς την αντιμετωπίζετε. Είπατε κάποια πράγματα, αλλά τι ακριβώς σημαίνει, εκτός τώρα από τα fake news. Είπαμε, αυτό είναι η μία πτυχή. Υπάρχουν εδώ ε, κάποια στοιχεία τα οποία βάζετε στην ερώτησή σας και το πρώτο πώς διακρίνεται ανάμεσα σε εμπορική διαφήμιση και πολιτική διαφήμιση και ε, ποια μεταχείριση επιφυλάσσεται στις μεν και στις δε. Κάτι που έχουμε κάνει και το είπα αρχικά είναι ότι φτιάξαμε ένα εργαλείο που λέγεται View Ads, το οποίο αντιμετωπίζει όλες τις διαφημίσεις ως ίδιες, ε, βασιζόμενο στην πεποίθηση ότι ο καθένας θα πρέπει να μπορεί να βλέπει όλες τις διαφημίσεις τις οποίες ε, προωθεί ένας συγκεκριμένο διαφημιστής διότι έχουν τη δυνατότητα οι διαφημιστές να μικροστοχεύουν κάποια τμήματα του κοινού χωρί να γνωρίζει όμω ο υπόλοιπο εκλογικό πληθυσμό ότι αυτό συμβαίνει. Εμεί προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό μέσω του εργαλείου View Ads ώστε όλοι να μπορούν να παίξουν το ρόλο του πολιτικού ε, χωροφύλακα εντό εισαγωγικών, watchdog, δηλαδή να μπορεί να παρακολουθεί τι ακριβώ κάνουν αυτοί οι διαφημιστέ. Αυτού του είδου η διαφάνεια θα συμβάλλει σημαντικά στην ικανότητα του κοινού να ζητεί από τους ε, πολιτικά δρόντες να λογοδοτούν σχετικά με το τι κάνουν με τις εκλογικές διαφημίσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι εμείς θεωρούμε εκλογική χειραγώγηση, εκεί ε, στοχεύουμε σε πράγματα τα οποία βλέπουμε, δηλαδή παραπληροφόρηση, clip baiters, sensationalism και ούτω καθεξής. Βλέπουμε δηλαδή τι γίνεται στην πλατφόρμα μας, πράγματα που μπορούμε να εντοπίσουμε και αναλαμβάνουμε δράση κατά αυτόν. Εγώ εξήγησα προηγουμένως διαφόρους τρόπους με τους οποίους προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και να καταπολεμήσουμε διάφορα είδη χειραγώγησης και εκμετάλλευσης και θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, να τα κάνουμε αυτά και όταν εντοπίζουμε μια συμπεριφορά που θεωρούμε ότι δεν είναι γνήσια ή προσπαθεί να παραπλανήσει να λαμβάνουμε την κατάλληλη δράση εναντίον της. Πέντρο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ πολύ για τον κύριο Κάπλαν. για κάποιους από τους πιο προηγμένους τρόπους κακό μεταχείρι, ε, ε, κακής μεταχείρι, ε, χρησιμοποίησης του Facebook για σκοπούς προεκλογικών εκστρατείας ε, με μεταφορά πληροφοριών σε στο ιστοτόπους. Εγώ θα σας έλεγα ότι υπάρχουν και απλούστεροι τρόποι κακές χρήσεις για πολιτικούς σκοπούς της πλατφόρμας σας. Διάδοση ψευδών πληροφοριών, ε, ε, ψεύτικες εκστρατείες, ανώνυμοι σχολιαστές, που σε καθημερινό επίπεδο συναντούμε παντού. Όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς κάποιο μητρό αξιόπιστης καταγραφής ηλεκτρονικής ταυτότητας. Υπάρχει κάποιο μέλλον. Ευχαριστούμε. Και πάλι έχουμε μια σειρά από τρόπους να αντιμετωπίσουμε την εξάπλωση νοθευμένων πληροφοριών για προεκλογικές εκστατείες. Τους ανέφερα εδώ σήμερα. Μίλησα για τους ψευδείς λογαριασμούς, τα χρηματικά κίνητρα, την άρση των κινήτρων, για να πάψουν να έχουν δραστηριότητα στο Facebook ε, με τους ελεγκτές από τρίτη πηγή για να μπορούν να ε, επαληθεύσουν την, ε, την αλήθεια, το βάσιμο μιας πληροφορίας. Ε, και να δούμε αν μπορούμε να περιορίσουμε την εξάπλωση της είδηση αυτής. Επίσης κοιτάζουμε τη διάδοση άλλου περιεχομένου χαμηλής ποιότητας, το clickbait, τον αισθησιασμό. Κοιτάζουμε να περιορίσουμε τη διάδοση στο newsfeed και προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε την διάδοση και διανομή αξιόπιστων πληροφοριών από πηγές που ο κόσμος στο facebook θεωρεί αξιόπιστες. Ειδήσει που ενημερώνουν, που έρχονται από τοπικές ελεγμένες πηγές και που ε, είναι μια μάχη που όλοι μας θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε για τον ψηφιακό ρόλο των κυβερνήσεων για την ιδιότητα του πολίτη και στο ψηφιακό περιβάλλον, για όσα θέλουν να βλέπουν στο διαδίκτυο και για να διαδραματίζουμε το ρόλο μας στην διάδοση αυτού του περιεχομένου. Θα προσπαθήσουμε να εκπαιδεύουμε τον κόσμο και εντός πλατφόρμας και εκτός για το πώς να ε, αφομοιώνουν τις διάφορες ειδήσει. Βεβαίω, αν ήταν άλλο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο και η Χιλάρη Κλίντον είχε βγει πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν θα βρισκόμαστε εδώ να συζητάμε όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά είμαστε εδώ και για την κυρία Μπάσχατ και την εκλογική τη επιτροπή. Είπε ότι παρά το ρόλο της Επιτροπής να επιβάλλει τους κανόνε και να διασφαλίσει ότι οι δωρεέ ήταν ε, νόμιμε. Έχουμε δύο εκστρατείε ε, κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματο που χρησιμοποίησαν παραδοσιακότερα μέσα. Η κυβέρνηση τη αυτή μεγαλειότητα ξόδεψε περίπου 10 εκατομμύρια στελίνε, ένα φυλάδι που πήγε σε κάθε νοικοκυριό του Ηνωμένου Βασιλείου και για ένα μόνο ε, μέρο του επιχειρήματο, το Remain. Ε, αυτά καταγράφηκαν και έπειτα ως προς την εξωτερική παρέμβαση στο δημοψήφισμα. Ο πρόεδρος Ομπάμα έκανε μια δική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να επηρεάσει απευθεία το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την πλευρά του Remain. Ε, ήταν εκατομμύρια τα δολάρια που δαπανήθηκαν για αυτή την επίσκεψη. Καταγράφτηκαν αυτά ως ε, ενδεχομένω δωρεά. Και πώς ο πρόεδρος Ομπάμα μπορεί να είναι ένας παραδεκτός δωρητής. Κοιτάξτε, το φυλάδιο που διένει με κυβέρνηση έγινε πριν από τις 10 εβδομάδες ε, και την περίοδο που καταγράφουν τις δαπάνες, οπότε δεν μπορούσε να καταμετρηθεί έτσι λογιστικά. Όπως οι κανόνες πέρναγαν από το Κοινοβούλιο, ισχυριστήκαμε ότι έπρεπε να είναι μεγαλύτερη περίοδος που καταγράφεται ως προεκλογική. Θα το είχαμε καλύψει σε αυτή την περίπτωση. Όμως, σε εκείνο το δημοψήφισμα η δραστηριότητα αυτή έγινε πριν τις 10 εβδομάδες. Την επίσημη προεκλογική περίοδο καταγράψαμε όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Υπάρχουν σχετικές ε, εκθέσεις. Η κυρία Σκοτ Κέιτο για τους Πρασίνους και εγώ για την κυρία Μπάσετ. Καταλαβαίνω ότι έχετε ολοκληρώσει την έκθεσή σας για την ε, παράνομη διαπλοκή μεταξύ των όσων ε, επισήμως υποστήριξαν το ΛΥΒ στο δημοψήφισμα αλλά δεν σχολιάστε το αντίστροφο και τι μαρτυρίε του επίση για κάποια μέλη τη επιτροπή μα. Ε, να μην ξεχνάμε ότι ο Μπόρις Τζόνσον και ο ε, Υπουργό Περιβάλλοντος Γκόπ έχουν κάνει δηλώσει σχετικά. Οι κανόνε δαπανών παραβιάστηκαν ανάλογα με την... Ε, ε, αντίληψη ο καθένα για την εντολή του Ηνωμένου Βασιλείου να φύγει όχι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, αυτά θα δημοσιοποιηθούν ποτέ και εσεί τι μπορείτε να κάνατε για τις ε, διαρροές δημοσιοποιήσεων και κάποιους από αυτούς που μπλέκονταν σε όλα αυτά. Είναι μέρος του όλου δημόσιου διαλόγου για το θέμα αυτό και πρέπει πριν το Ηνωμένο Βασίλειο όντως αποχώρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα γνωρίζουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Για να υπάρχει τουλάχιστον μια σαφής και νόμιμη εντολή. Να εξηγήσω απλώ ότι έχουμε μια πολιτική επιβολή που καταρτίζει πολύ σαφώ πώ προχωρούμε και πώ θα ολοκληρωθούν οι έρευνε είναι μέρος αυτής της διαδικασίας το ε, πώς θα προχωρήσουμε στην ε, εφαρμογή της απόφασης. Έχουμε 28 μόνο ημέρες εντός τις οποίες μπορούν να γίνουν ε, προσφυγές. Οι προσφυγές αυτές λαμβάνουν υπόψη να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Συμπεράσματα τα οποία δημοσιοποιούμε και για τα οποία θα υπάρξουν και λεπτομερέστερες έρευνες ε, στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα. Δεν μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες για ενεξέλιξη έρευνες, είναι σαφής πολιτική της εκλογική μας επιτροπής και είναι νομίζω και πολύ σωστή γιατί αποφεύγουμε τις ακαμπόδεις συζητήσεις. Παρόλα αυτά, Υπάρχουν κάποια στοιχεία που κυκλοφόρησαν για συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία δεν ξέρω από πού προήλθαν. Έχω ακόμη χρόνο. Λέτε ότι δεν έχετε τις αρμοδιότητες διαρεύνησης της ε, ε, Cambridge αναλυτικά. Τότε ποιος την έχει την αρμοδιότητα αυτή και έχετε την αρμοδιότητα και την εξουσία να ανακόψετε αυτές τις αλλοδαπές παρεμβάσει σε εκλογές από ξένες ε, ε, εξουσίες. Και ποιο μπορεί τότε. Είπα καθαρά ποια είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων μας του ICO, Information Commission Officer. Πολλά από τα πράγματα που ακούσαμε σήμερα εδώ αναφέρονται σε παραβιάσεις της νομοθεσίας της προστασίας δεδομένων και είναι αντικείμενο συνεχιζόμενων ερευνών, την έκβαση των οποίων θα πληροφορηθούμε σύντομα. Έχουμε διαφορετικούς ρυθμιστές σε διαφορετικούς τόπους που συνεργάζονται για την αντιμετώπιση πάρα πολύ σοβαρών θεμάτων. Οι έρευνές μας αναφέρονται στο πότε γίνεται η χρηματοδότηση, αλλά επισημαίνω και πάλι ότι πρόκειται για συνεχιζόμενες έρευνες, οπότε κολλείομαι να σχολιάσω. Hang me, you know, whatever. It's just so boring to, stick to Μάλιστα, συνεχίζει ο πρόεδρο. Βεβαίω, ε, ερωτήσεις, απαντήσεις αποτελούν ήδη μια βελτίωση. Θα ευχαριστήσω όλες τις ομιλήτριες και ομιλητές για τις ε, ε, μαρτυρίες τους θα ευχαριστήσω και τα μέλη ευρωβουλευτές για την υπομονή και πειθαρχία που έδειξαν. Να περάσουμε στην τρίτη συνεδρία. Θα έχουμε και άλλα μέλη που θα προσέλθουν, δηλαδή ευρωβουλευτές. Στην επόμενη συνεδρία πάντως θα αρχίσουμε 18 και 15, ώστε να προλάβουν να προσέλθουν όσοι βρίσκονται καθοδόν. Σύντομο διάλειμμα λοιπόν λίγων λεπτών για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν οι ομιλητές μας. Και ο πρόεδρος αναφέρει τα ονόματα. Um, and the, and the chair will be Joseph Weidenholzer for this next session. So, colleagues, oh, and th thank you to our AFCO chair, Danuta Hubner, very much. Thank you, Danuta.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 αλλά δεν είναι Ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ, Προεδρεύων. Ε, ευχαριστώ που ήρθατε. Καλό σας απόγευμα. Είναι η τελευταία ε, συνεδρία για σήμερα. Γίνεται μαζί με την Επιτροπή Ήτρε και τον ε, συνάδελφό μου Πάουλ Ρούμπικ, στον οποίο θα δώσω το λόγο για λίγα λεπτά. Πριν όμως του δώσω τον λόγο, θα ήθελα να σας πω ποιοι είναι εδώ. Ο αντιπρόεδρος της ΕΝΙΣΑ, η κυρία Μπάχλ, ο κύριος Σρίμς, privacy activist, Ρίτσαρτ Άλλαν, αντιπρόεδρος άλλου οργανισμού που παρακολουθεί το Facebook. Yes, many thanks. Ο κύριος Ρούμπιχ τώρα, στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ είναι πολύ καλός χρονομέτρης. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Είμαι μέλος της Επιτροπής Ήτρε και της ΣΤΟΑΣ, που είναι η Επιτροπή ε, Αξιολόγηση Τεχνολογίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ασχολείται με την έρευνα στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να δούμε πώς μπορεί να αυξηθεί η ποιότητα των trust instruments. Μέχρι τώρα πράττουν αυτό που ζητούν οι τρίτοι. Η ερώτησή μου είναι πώς μπορούμε να αυξήσουμε την δύναμη των καταναλωτών. Ε, να έχουν δηλαδή εγγυημένη την ταυτότητά τους. Δηλαδή, ποια εγγύηση μπορούμε να προσφέρουμε για την ψηφιακή ταυτότητα, διότι είναι πολύ εύκολο να πλαστογραφηθεί η ταυτότητα κάποιου που εισέρχεται στο διαδίκτυο. Εφόσον συμβεί αυτό, πώς μπορώ να διατηρήσω την κυριότητα των δεδομένων μου και πώς μπορούμε επίσης να βγάλουμε έξω από τα κοινωνικά μέσα τις ψευδείς ειδήσει. Επαναλαμβάνω τα ερωτήματα, εγγύηση της ε, ψηφιακής ταυτότητας, κυριότητα των δεδομένων και δραστηριοτήτων μου. Εγώ μπορώ να διοδοτήσω ένα τρίτο μέρος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει την ταυτότητά μου και τη γνώση των δεδομένων μου. Τι μπορώ να κάνω κατά των λεγόμενων avatar, οι οποίες μπορούν, με τα οποία avatar μπορούν, ως γνωρίζετε, να αντιγράψουν ένα προς ένα τις ε, ψηφιακές ταυτότητες και πώς μπορεί η ε, Ένωση να εγγυηθεί την ε, ψηφιακή μας ταυτότητα. Our first speaker is now ο κύριος Στίβ Πέρσερ πρώτος. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους και σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να σας απευθύνω το λόγο. Κινδυνεύω να σας απογοητεύσω όμως διότι εμείς έχουμε έρθει εδώ ως ακροατές και έχοντας ακούσει την συζήτηση του σημερινού απογεύματος εντυπωσιάστηκα για το πόσο λίγα από τα ζητήματα που συζητείτε εδώ είναι μέσα στο πρόγραμμα MSO. Διότι αυτά είναι σημαντικά πράγματα και τα περισσότερα που άκουσα σήμερα δεν εμπλέκουν τον οργανισμό ίσα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει στο μέλλον και αυτό είναι το μήνυμα που έχω να σας μεταφέρω. Θα κάνω λίγα σχόλια πάντως και θα είμαι στη διαθεσή σας για ερωτήσεις. Ας αρχίσουμε με τα θετικά πρώτα. Το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα ασφαλώς έχουν ανοίξει νέες δυνατότητες για την διάδοση της δημοκρατίας, των ελευθεριών και των αξιών. Α μην το αυτό στη συζήτηση αυτή, διότι το χειρότερο μπορούμε να κάνουμε, ε, καθώ θα βάζουμε κάποια, κάποια μέτρα ελέγχου, είναι να ανακόψουμε αυτή τη θετική εξέλιξη. Αν το σκεφτείτε καλά, τα κοινωνικά μέσα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη λεγόμενη αραβική άνοιξη του 2011 και μετά αργότερα το 2014 στην Ουκρανία. Το μήνυμα ήταν ότι εν τέλει ο λόγος είναι ισχυρότερος από το ξύφο. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα που προσφέρει, ε, προσφέρουν αυτά τα νέα κοινωνικά μέσα. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι βέβαια εκτός από τις παλαιές απειλές τις οποίες γνωρίζουμε από ετών, ε, βλέπουμε και ένα νέο είδος απειλών, αν θέλετε, το οποίο είναι ας πούμε απειλητικότερο από τις παλαιές ε, επιθέσεις ιών και κάτι τέτοια διότι τουλάχιστον ε, μπορούσε κανείς να εντοπίσει τον ιό, ε, μιλούμε, μιλούμε πάντως στο διαδίκτυο. Μιλούμε όμως τώρα για ψευδείς ειδήσει, για εγκληματική χρήση ε, των δεδομένων άλλων και ούτω καθεξής. Εκτός από αυτό, εδώ ωστόσο υπάρχει μία διαφορά. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι είναι πολύ ανεπαίσθητες οι ε, αλλαγές αυτές, οι απειλές αυτές και συνήθως δεν το αντιλαμβάνεται για κανείς ότι πέφτει θύμα των απειλών αυτών. Και αυτό υποσκάπτει ωστόσο την εμπιστοσύνη. Ψηφιακός κόσμος χωρίς εμπιστοσύνη είναι ψηφιακός κόσμος ο οποίος δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Και αν επιβιώσει ακόμη, ίσως να επιβιώσει με έναν τρόπο που να μην είναι χρήσιμος για τους ε, πολίτες είναι τεράστιο το θέμα της εμπιστοσύνης. Μιλώντας για εμπιστοσύνη βέβαια, η εμπιστοσύνη δεν αρκεί. Είναι αναγκαία συνθήκη, ωστόσο δεν είναι επαρκής. Και εκεί μπαίνει η διάσταση της κυβερνοασφάλειας, όπου παίζει ένα ρόλο ο οργανισμός ΕΝΙΣΑ. Η κυβερνοασφάλεια είναι οι τεχνικές εκείνες που χρησιμοποιούμε για να περιορίσουμε την πρόσβαση σε δεδομένα στη βάση κάποιων αρχών. Οι αρχές αυτές μπορεί να παραλλάσσουν από περίπτωση σε περίπτωση και ανάλογα με το πλαίσιο. Αυτό όμως είναι που κάνει και την ασφάλεια δύσκολη υπόθεση. Το πλαίσιο είναι πολύ σημαντική υπόθεση στην ασφάλεια και η λήψη υπόψη είναι επίσης δύσκολη. Υπό ορισμένες συνθήκες η κυβερνοασφάλεια μπορεί να περιορίσει και την χρήση των δεδομένων. Το άσχημο νέο βέβαια είναι ότι αυτή τη βγάλετε το δεδομένο από το πλαίσιο του συστήματος που χρησιμοποιείτε είναι game over. Αυτή τη στιγμή το δεδομένο φύγει από το πλαίσιο, έχει φύγει και από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει με αυτό. Αυτό είναι και η υπόθεση της Cambridge Analytica και σε κάποιο βαθμό και το τι γίνεται με όλα τα δεδομένα και όλο και περισσότερο καθώς περνά ο χρόνος. Από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε τώρα είναι η συλλογή και παραπέρα διάδοση των δεδομένων στο διαδίκτυο που είναι απολύτως διαδομένη είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι και πάλι, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή στο δεδομένο βγει έξω από το πλαίσιο, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί η χρήση του. Βέβαια, ο GDPR δεν επιτρέπει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση. Πώς όμως να ελέγξει κανείς όταν γνωρίζει τι γίνεται. Επανέρχομαι τώρα στην ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι πάντοτε συνδυασμό τριών ε, παραγόντων. Άνθρωποι, διαδικασίε, τεχνολογία. Γενικά, ένα από τα σφάλματα που έχουμε κάνει στο παρελθόν και εξακολουθούμε να διαπράττουμε σήμερα είναι ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τεχνολογία, ε, στην τεχνολογία, στην υπερβολική βαρύτητα στην τεχνολογία. Ενώ τα περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα, προβλήματα ασφάλεια, ε, έχουν σχέση με ανθρώπου και με διαδικασίε. Βλέπουμε δηλαδή αποτυχία των διαδικασιών όπου μία επιχείρηση μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσει με παράνομο τρόπο. Επίση, πολιτικέ. Τι νόημα έχει να υπάρχει μια πολιτική όταν δεν μπορεί να επιβληθεί. Ούτε μπορώ να θεωρήσω, ε, μπορώ να θεωρήσω μάλλον ότι μια πολιτική είναι δύσκολο να εφαρμοστεί όταν υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι. Όμω, ε, ένα από τα μηνύματα αυτόν που πρέπει να πούμε τώρα δηλαδή, είναι ότι η ισορροπία ανάμεσα σε ευκαιρία και κίνδυνο πρέπει να αλλάξει. Μπορεί να μην μπορέσουμε ίσως να ελέγξουμε τα πάντα στο λεγόμενο διαδίκτυο των πραγμάτων όπως τώρα, αλλά έχουμε ένα καθήκον προφύλαξης και να θεσπίσουμε διαδικασίες μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, ρήτρας προφύλαξης. Για να επανέλθω στην αρχή, ε, πρόκειται για παραβίαση όχι μόνο διαδικασιών και πολιτικής, αλλά και για παραβίαση εμπιστοσύνης και αυτό μπορεί να είναι πραγματική καταδίκη σε θάνατον του διαδικτύου. Θεωρούμε ότι ο κανονισμός GDPR είναι φιλόδοξο σχέδιο και πραγματικά ε, απόλυτα χρήσιμο νομοθέτημα. Είμαστε απολύτως στην υπηρεσία του GDPR. Θα παρακολουθήσουμε τι θα μας πείτε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την εφαρμογή του GDPR και επαναλαμβάνω το μήνυμα ότι ο κόσμος αλλάζει. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος δεν είναι τα προβλήματα για τα οποία δημιουργήθηκε ο ΕΝΙΣΑ. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι δεν μπορούμε να ε, αλλάξουμε και εμείς ώστε να παρακολουθούμε τις αλλαγές για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, για την αντιμετώπιση της κλοπής ψηφιακών ταυτοτήτων κλπ. Εσείς έχετε τη δυνατότητα και την εξουσία να τα αλλάξετε. Ας ολοκληρώσω λέγοντας ότι Υπάρχει το άρθρο 14 του, ε, της αρχικής οδηγίας που επιτρέπει στις χώρες μέλη ε, να ζητούν ανάληψη ειδικών καθηκόντων από τον ΕΛΙΣΑ. Να κάνετε χρήση του μηχανισμού αυτού που επιτρέπει κινητοποίηση βραχυπρόθεσμα και έχει μεγάλη ισχύ. Εδώ θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου και σας ευχαριστώ και πάλι. Yes, many thanks to you and... Σας ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής η Ούρσουλα Πάχλ αναπληρώτη διευθύντρια στην Μπεούκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτά που αποκαλύπτει το σκάνδαλο Facebook Cambridge Analytica έχουν και θα έχουν σοβαρές συνέπειες στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Το σκάνδαλο αυτό δεν έχει σχέση απλώ με την εμπιστοσύνη προ το Facebook, αλλά με όλο το αρχιτεκτόνιμα τη ψηφιακή οικονομία. Και αυτή είναι η προοπτική που πρέπει να υιοθετήσουμε όταν βλέπουμε την κατάσταση. Ο τρόπο που τα πράγματα λειτουργούν τώρα είναι ότι η εκμετάλλευση των δεδομένων, η αξιοποίησή του είναι μια βασική πηγή εισοδήματο στο διαδίκτυο και όχι μόνο από το Facebook. Οι παράνομε χρήσει περιεχομένου μπορούν να συμβούν παντού, σε πολλέ πλατφόρμε του διαδίκτυου. Το γενικό λοιπόν αίσθημα των καταναλωτών και των υπερασπιστών του είναι ότι η διαφάνεια που χρειαζόμαστε δεν υπάρχει στι πλατφόρμε και ότι η προστασία των δεδομένων καθώ και τα δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά. Δεύτερον, και θα ήθελα εδώ να τονίσω, δεν είναι μόνο θέμα εμπιστοσύνη και με συγχωρείτε κιόλα θα το πω, είναι πολύ βασικότερο. Είναι θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία δεν γίνονται σεβαστά και αυτό φαίνεται ανάγλυφα από την περίπτωση του Facebook Cambridge Analytica, διότι δεν διακυβεύεται μόνο η εμπιστοσύνη, είναι θέμα παρανομίας. Ε, η περίπτωση Facebook, βάσει των επίσημων ανακοινώσεων του Facebook, αφορά 2,7 εκατομμύρια ε, Ευρωπαίους μόνον. Εμένα αυτό κάπως με φνηδίασε, με δηλώσεις που ακούστηκαν ότι τα δεδομένα των Ευρωπαίων καθόλου δεν επλήγησαν. Είναι μια αντίφαση αυτό που προέκυψε σήμερα εδώ. Μου θυμίζει λίγο την περίπτωση Volkswagen που ε, ζήτησαν συγγνώμη αρχικά και μετά είπαν ότι μερικά πράγματα ήταν εκτός των, ε, της δικαιοδοσίας τους. Εδώ λοιπόν, <clears throat> χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των καταναλωτών, τη συγκατάθεσή τους, δεδομένα τους πωλήθηκαν σε άλλους για σκοπούς διαφορετικούς από τους αρχικούς. Η υπόθεση Cambridge Analytica είναι ε, μια υπόθεση που ε, ήδη οδήγησε στην διακοπή 200.000 αδειών για ενδεχόμενη κακή και παράνομη χρήση δεδομένων. Μιλάμε για την κορυφή του παγόβουνου. Αν δει ε, αν σκεφτεί το Facebook, σίγουρα θα πρέπει να είναι βέβαιο τα δεδομένα του κάποιο τα χρησιμοποίησε παράνομα κάποια στιγμή στον χρόνο. Και αν όχι, κάποια στιγμή τα δεδομένα του ε, σίγουρα έχουν περάσει εκεί που δεν έπρεπε. Υπήρξε λοιπόν πρόσβαση σε τρίτα μέρη για να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά και με τη γνώση ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά παράνομα. Το Facebook λοιπόν δεν ανέλαβε τα ε, απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Και η απόκριση τη εταιρεία ω τώρα δεν είναι ικανοποιητική. Μόνο κάποιε καλοπιστικέ αλλαγέ στην πλατφόρμα έγιναν και αυτό δεν είναι ε, αρκετά ικανοποιητικό κατά την άποψή Προφανώ. Οι αλλαγέ στην πολιτική ιδιωτικότητα του Facebook μπορεί να έχουν περιγραφεί ω άμεση αντίδραση στο σκάνδαλο αυτό. Και εδώ η εφαρμογή του GDPR ε, έχει να κάνει και με το πώς εφαρμόζει τώρα την πολιτική του περιδιωτικότητα στο Facebook δεν αρκεί απλώς να κάνουμε καλοπιστικές αλλαγές, αλλά να κοιτάξουμε και την ουσία της πολιτικής του Facebook και τη δομή της πλατφόρμας. Η δομή του business model του Facebook και το πώς ε, βγάζει χρήμα το Facebook είναι ένα θέμα. Οι διαφημίσεις είναι φυσικά το βασικό όφελος των ε, ψηφιακών εταιριών και βεβαίω και για του καταναλωτέ είναι σημαντικό να αποφύγουν κάθε σύγκρουση συμφερόντων. Πώ όμω αισθάνονται γι' αυτό οι καταναλωτέ, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν γίνει ενδιαφέρουσες μελέτες για την χρήση των δεδομένων που έχουν δείξει ότι υπάρχει η αίσθηση ότι οι καταναλωτές δεν έχουν καθόλου την κατάσταση στα χέρια τους. Ο κόσμος είναι ανασφαλής για το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα από αυτές τις πλατφόρμες και κατά πόσον είναι νόμιμη η χρήση ή κατά πόσον μπορούν να αναλάβουν δράση για τις διάφορες πρακτικές. Ε, ε, αισθανούνται αποδυναμωμένοι διότι η συμπεριφορά τους μπορεί κατά λάθο να τους προκαλέσει προβλήματα. Και οι μελέτες δείχνουν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι καταναλωτές συνήθως τα παρατάνε. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ερωτήσεις μεταξύ των καταναλωτών αλλά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το Facebook διότι σε τελική ανάλυση κάνουν σαν να μην τους ενδιαφέρει αλλά οι πραγματικοί λόγοι δεν είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει είναι ότι αισθάνονται αδύναμοι ότι έχουν υποταχθεί και υπάρχει, δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν υπάρχει κάτι που να αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή το Facebook. Φυσικά το σκάνδαλο άνοιξε τα μάτια πολλών ε, καταναλωτών φυσικά. Ένα σημείο το οποίο εκπλήσει στην ε, όλη συζήτηση είναι ότι στο σκάνδαλο της Cambridge Analytica με το Facebook δεν δόθηκε επαρκής προσοχή στη ζημιά που έχουν υποστεί οι καταναλωτές διότι τα δικά του δεδομένα καταχράστηκαν αυτές οι εταιρείε. Γι' αυτό το λόγο σήμερα ε, ε, τα μέλη από Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία ε, από τις ενώσεις καταναλωτών αυτών των χωρών ε, ξεκίνησαν μια ομαδική δράση συλλογικής αποζημίωσης κατά του Facebook. Σήμερα ήταν το Βέλγιο, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλοι τις επόμενες μέρες. Ζήτησαν αποζημίωση στο Βέλγιο από το Facebook το Βέλγιο ήδη 20.000 άνθρωποι συνυπέγραψαν αυτή τη δράση. Ζητούν ε, αποζημίωση όχι μόνο για όσους υπέστησαν ζημία από την Cambridge Analytica, ζήτησαν ε, να αντιπροσωπεύσουν όλους τους χρήστες του Facebook για τους λόγους που μόλις εξήγησα. Δύο λόγοι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Είναι ένα θέμα στενά συνδεδεμένο με το ιδιωτικό απόρριτο φυσικά. Τα δεδομένα που έχετε, που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι ασφαλή. Ε, πρέπει να είναι ασφαλή από ανεπιθύμητη εισβολή. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς μια υπηρεσία αν ξέρει ότι είναι ανασφαλής. Αλλά όπως ξέρουμε εδώ, στην περίπτωση του Facebook και της Cambridge Analytica, το θέμα δεν ήταν ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ήταν ότι απλά το Facebook άνοιξε τις πόρτες του σε τρίτα μέρη και τους έδωσε τα δεδομένα. Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι τι είδους υποχρεώσεις έχουμε για να ε, διασφαλίσουμε την προστασία και την ασφάλεια των χρηστών. Πρέπει να πω ότι αυτό που γνωρίζουμε από την έρευνα μεταξύ των καταναλωτών είναι ότι ε, όταν μιλάμε για υποταγή των καταναλωτών αυτό ισχύει και για τα θέματα ασφάλειας. Η έρευνα μας δείχνει ότι δεν καταλαβαίνουν οι καταναλωτές τι συμβαίνει με την παραβίαση δεδομένων. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα σύστημα ούτε σε εταιρεία ούτε σε κράτο που να του βοηθά να βρουν κατά πόσο έχουν κλαπεί τα δεδομένα του ή κατά πόσο έχουν πουληθεί ή δημοσιευτεί κατά κάποιο τρόπο. Αφού λοιπόν αρχίζουν να κυκλοφορούν τα δεδομένα, κυκλοφορούν ελεύθερα και κανεί δεν ξέρει τι γίνεται με αυτά τα δεδομένα αφού δοθούν. Και οι καταναλωτέ τελικά είναι μόνοι του με αυτή την κατάσταση. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι έχουμε διάφορα, θα έχουμε συνδεδεμένα προϊόντα στα σπίτια μα πολύ σύντομα και ε, όχι απλά θα σας βοηθούν αυτά, αλλά είναι εύκολο να τα παραβιάσει κανείς. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χάσει την ευκαιρία να θεσπίσει ε, δεσμευτική νομοθεσία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αυτή τη στιγμή ρυθμίζεται μόνο με εθελοντικά μέτρα. Κάτι που δεν υποχρεώνει κανέναν να εφαρμόζει ασφάλεια ε, ως προεπιλογή και να την ενσωματώνει στα συνδεδεμένα προϊόντα, για παράδειγμα. Αυτό είναι δυστυχές διότι ξέρουμε όλοι ε, ως τώρα ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην αυτορύθμιση και στην ε, υποτιθέμενη καλή θέληση αυτών των εταιριών χρειαζόμαστε ε, παγιωμένη νομοθεσία. Συμπερασματικά τώρα να σας πω δύο παρατηρήσει. Πρώτον, οι καταναλωτέ χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη για επανεξορρόψη τη ε, δύναμη που έχουν, του ελέγχου που έχουν των δεδομένων του. Έχουμε το GDPR, αυτό είναι πολύ καλό. Σύντομα θα έχουμε, ελπίζουμε, και την οδηγία για, την, ε, για το ηλεκτρονικό απόρριτο, αλλά χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα. Πιστεύουμε ότι η GDPR θα επηρεάσει θετικά την κατάσταση, αλλά χρειαζόμαστε πραγματική τη υλοποίηση, εφαρμογή. Και εδώ επανέλθουμε σε αυτά που είπε η κυρία Γέλνεκ για το μηχανισμό συνοχή, διότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκέ απαντήσει σε αυτέ τι μεγάλε εταιρείε και στι ε, παραβιάσει που κάνουν σε ευρωπαϊκό αν όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε σχέση με το Facebook πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο όχι μόνο να λαμβάνουμε υπόψη μα το σκάνδαλο τη Cambridge Analytica αλλά να κάνουμε και μια ευρεία έρευνα, ειδικότερα όσον αφορά τις σημερινές πρακτικές του Facebook, κάτι που θα επιτρέψει να βασιστούμε και στους ε, σημερινούς κανόνες του GDPR και να λάβουμε μια απόφαση που πραγματικά να αλλάξει την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει μια έρευνα αγοράς στις ψηφιακές ε, αγορές. Το έχουμε ήδη ζητήσει αυτό στην ομάδα υψηλού επίπεδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά το αίτημά μας δεν έγινε δεκτό η αποζημίωση των καταναλωτών για την απώλεια των προσωπικών του δεδομένων θα πρέπει να είναι κάτι αυτονόητο. Και ήθελα να πω ότι έχουμε μία πρόταση συλλογική αποζημίωση ε, για του καταναλωτέ, ε, την οποία θα σα ζητήσουμε να υποστηρίξετε. Έχω σχεδόν τελειώσει. Το τελευταίο Χρειαζόμαστε πιο δυνατά μέτρα για να διασφαλίζεται ε, η υπευθυνότητα όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα από τρίτα μέρη. Όπω φαίνεται, δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Υπάρχουν μόνο όροι και προποθέσει ε, για την παρακολούθηση και για την χρήση αυτών των δεδομένων. Δηλαδή, ουσιαστικά τι λέμε, ότι ο καθένα έχει τα, τη δική του πολιτική, η Cambridge Analytica έχει μια άλλη πολιτική, το Facebook άλλη πολιτική και τι θέλετε να κάνουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερη λογοδοσία από αυτήν την άποψη. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι οι καταναλωτών θα πρέπει να συμβάλλουν με ε, διαμαρτυρίες και νομική δράση, αλλά χρειαζόμαστε συλλογική, ε, συλλογικά ένδικα μέσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειαζόμαστε μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη, κάτι που δεν είναι αυτονόητο ούτε δεδομένο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλήτή ο Μαξ Schrems. Γεια σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρέπει να πω ότι με μεγάλη χαρά ε, προσήλθα σήμερα σε αυτή την ακρόαση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντικό το γεγονό ότι το Ευρωκοινοβούλιο διοργανώνει αυτή τη συνεδρίαση. Όσον αφορά την εμπιστοσύνη, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτε και οι χρήστε να έχουν εμπιστοσύνη γενικά στην ψηφιοποίηση και πρέπει να το πετύχουμε. Ο λόγος για τον οποίο προσέβλεπα σε αυτήν την ε, συνεδρίαση σήμερα είναι ότι τα πάντα όλα αυτά τα στοιχεία ήταν γνωστά από το 2011 και μάλιστα ε, είχαμε συζητήσει για 7 ώρες το 2011 τα προβλήματα ε, αυτά με τις εφαρμογές το 2011 ξαναλέω. Φαίνεται λοιπόν ότι 7 χρόνια αργότερα ερχόμαστε και διαπιστώνουμε ότι τελικά υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ποιος κοιμόταν λοιπόν το Facebook ή οι αρχές. Και μιας και το αναφέρω να σας εξηγήσω τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχει λοιπόν το Facebook το οποίο ε, ε, τότε το 2011 έστελνε δεδομένα χρηστών ε, μέσω της Facebook Ireland, Ιρλανδίας, σε εταιρεία που έφτιαχνε συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτό ήταν ε, νόμιμο ή παράνομο. Γι' αυτό άλλωστε είχαμε υποβάλει τότε εκείνη την καταγγελία. Είχαμε πει ότι δεν υπήρχε καμία συνένεση συγκατάθεση των χρηστών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να διαβιβαστούν τα προσωπικά του στοιχεία, τα προσωπικά τους δεδομένα. Και τελικά ακριβώς αυτό συνέβαινε. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι όλη αυτή η κατάσταση ήταν πρόβλημα. Τότε υπήρχαν 20 εκατομμύρια ε, ε, περιπτώσεις εγκατάστασης της εφαρμογής αυτής μέσω του, ε, Facebook. Τι να, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς ε, μάλιστα φτιάξαμε μια εφαρμογή για να ασκήσουμε αγωγή κατά της Facebook. 25.000 προσυπέγραψαν και εγκατέστησαν τη σχετική εφαρμογή. Έχω 25.000 ε, ομάδες δεδομένων, προσωπικών δεδομένων στον υπολογιστή μου. Και η Facebook ποτέ δεν με ρώτησε από πού τα πήρα, για ποιο, τι θα τα κάνω, σε ποιον θα τα διαβεβάσω. Αυτό λοιπόν αποτελούσε παραβίαση ε, μια σειρά άρθρων της οδηγίας. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι έγινε λογιστικός έλεγχος το 2012, ο οποίος στην, στην ε, Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία κατέληξε σε κάποιες συστάσεις προς το Πρέσβουκ, τα κάνει λίγο πιο όμορφα τα πράγματα, λίγο πιο εύχριστα. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιες, κάποιες, ε, σύνδεσμοι οι οποίοι να μην είναι ανενεργοί προς τις ε, πολιτικές απορρίτου του Facebook. Ποτέ όμως δεν εξέτασε η αρχή αυτή τη νομική βάση, ούτε τον νόμο ε, που διέπει αυτά τα πράγματα. Η Facebook ε, ε, ισχυρίστηκε ότι όλα αυτά εντάσσονται εντός της συμφωνίας που υπογράφουν οι χρήστες μαζί της όταν ε, φτιάχνουν λογαριασμό ότι σε τελική ανάλυση η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων αποτελεί πτυχή της κοινωνικής διάστασης της πλατφόρμας αυτής. Η Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων είχε πει τότε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωση, να τα φτιάξει το Facebook σα παρακαλούμε πολύ και ότι ε, αρκεί η συνεργασία μέσω των ε, κατασκευαστών των εφαρμογών ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κάναμε και μια συνάντηση του 2012 με τον Ρίτσαρντ Άλανμπεκ. Υπάρχει και πρακτικό τη συνάντηση αυτή και τότε ο Ρίτσαρντ ανέφερε ότι πιστεύουν ότι υπάρχει γενική συγκατάθεση. Δηλαδή όταν χρησιμοποιεί κανείς το Facebook συνενεί στο να διαβιβάζουν τα προσωπικά του στοιχεία σε τρίτους ακόμη και αν δεν τον γνωρίζει καν αυτόν τον τρίτο. Και αυτό μάλιστα αποτελεί και ενημερωμένη ε, συγκατάθεση του χρήστη. Κάτι που εμένα φυσικά δεν με έπεισε καθόλου. Ενδιαφέρον ήταν ότι υπήρχε και ε, γινόταν λόγος για την συγκατάθεση τρίτου που είναι και αυτό μια πολύ περίεργη και, και, και καινοφανής έννοια. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, κατά τη Facebook και αυτή η συγκατάθεση τρίτου. Ε, και ότι ο χρήστης είναι εκείνο που πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εφαρμογές που εγκαθιστά στο λογαριασμό του είναι εκείνε που συμμορφώνονται με τον νόμο και όχι η Facebook. Βάσει όλων αυτών έγινε εκ νέου έλεγχος και το 2012 η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιρλανδίας κατέληξε στο ότι η Facebook πρέπει να εξετάσει το ζήτημα και να βρει μια λύση. Το 2012 όλα αυτά, ε, πριν από 6 χρόνια η Facebook απάντησε στο ότι πλέον βασίζεται στις καταγγελίες ή στις αναφορές που κάνουν οι ίδιοι οι χρήστες. Ότι αν κάποιο χρήστη δηλαδή διαπιστώσει ένα πρόβλημα, έχει πλέον τη δυνατότητα να υποβάλει αναφορά στη Facebook. Που μάλλον δεν είναι και ότι καλύτερο που μπορεί κανεί να φανταστεί. Αυτά όλα δείχνουν διάφορα πράγματα. Πρώτον, επρόκειτο για κατάφορη παραβίαση της ισχύουσα νομοθεσία. Νομίζω ότι τα ίδια πράγματα περίπου πάνω κάτω συμβαίνουν και σήμερα με τη Facebook. Και βλέπουμε ότι οι αρχές απλά κλείνουν το μάτι. Κοιτάζουν από την άλλη μεριά. Γιατί πέρασαν χρόνια, τρία χρόνια, έως ότου η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιρλανδίας ε, μου έδωσε τελικά το πρακτικό των συναντήσεων με την Facebook ενδιαφέρον δεν είναι μόνο οι αλλαγές που θα επιφέρει ο GDPR. Αν δείτε την ε, πολιτική του και ιδιωτικότητας που εφαρμόζει η ε, Facebook, για παράδειγμα το ότι ε, να βγάζουν χρήματα από τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως συνέβη και με την υπόθεση του WhatsApp, τότε πραγματικά νομίζω ότι ούτε το γράμμα ούτε το πνεύμα του νόμου του GDPR ακολουθούν. Αλλά θα δούμε αν οι αρχές καταφέρουν να επιβάλλουν ε, την, ε, την νομοθεσία. Βεβαίως, μακροπρόθεσμα θα χρειαστεί και οι χρήστες να μπορούν να ε, εφαρμόζουν ή να, να ασκούν τα δικαιώματά τους. Για παράδειγμα, η υπόθεση που εκκρεμεί εναντίον του Facebook ε, έχει, ε, θα, θα επιφέρει 10 εκατομμύρια ε, ευρώ κόστος σε όποιον χάσει την υπόθεση, σε δικηγορικά έξοδα. Οπότε είναι και αυτό μια διάσταση. Χρειάζεται λοιπόν χρηματοδότηση για την επιβολή του νόμου τόσο στα κράτη-μέλη αλλά και σε πανενωσιακό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης προκειμένου να επιβάλλει την νομοθεσία διότι προφανώς το να ε, προσφύγει μια μη κυβερνητική οργάνωση ε, στα δικαστήρια λόγω του ότι το Facebook παραβιάζει την νομοθεσία είναι μια πάρα πολύ δαπανηρή υπόθεση. Διαφορετικό κεφάλαιο που επίσης θέλω να ανοίξω είναι το ζήτημα των ανοιχτών δικτύων. Επί της ε, ουσίας έχουμε μια αποτυχία στην αγορά. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μισούν το Facebook αλλά δεν έχουν εναλλακτικέ ε, που αναγκαστικά χρησιμοποιούν το Facebook γιατί δεν υπάρχει αναλυτική. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ε, δυστυχώς την χάνει της, της υποστήριξης των μεγαλύτερων και περισσότερων πολιτικών ομάδων. Δεν ανοίγουμε δηλαδή τα ανοιχτά δίκτυα. Ε, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο αν θέλουμε πραγματικά να αποκαταστήσουμε και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των χρηστών. Να αναγκάσουμε δηλαδή τις εταιρείε να πάρουν τέτοια μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Λόρδος Λίτσαρτ Ελν είναι πόσο μιλής από το 2009. Ασχολείται με την πώληση Europe γνωρίζει λεπτόμερος το θέμα. Έχετε λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαι εδώ και να είμαι στο πάνελ με τον Μάρξ. Δεν σε εκπλήσει το ότι έχω διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Από πλευρά της εταιρεία που άκουσε επικρίσεις, ήταν ανοιχτή σε επικρίσεις και είδα ότι η διαδικασία λειτουργήσε σωστά και οι ρυθμιστικές αρχές συμμετείχαν. Τελικά οι απόψει ήταν διαφορετικέ όσον αφορά την εφαρμογή τη νομοθεσία. Αυτό είναι το θέμα, την προστασία των δεδομένων. Υπάρχουν αποκλίνουσε απόψει όπως είναι η σύμφωνη γνώμη και λοιπά, η συνένεση. Και στους επόμενου μήνες και χρόνια αυτές οι αρχές θα δοκιμαστούν. κυβέρνηση, ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών αναφέρθηκε και στην προηγούμενη συνεδρίαση θέθηκε το θέμα, το θέμα των ευθυνών. Υπάρχουν σημαντικά θέματα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων να συζητηθούν αλλά και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι θέμα και το έχουμε επεξεργαστεί το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι ευρύτερο πεδίο και σχετίζεται με επιβλαβεί δραστηριότητε σε μια πλατφόρμα. Όσον αφορά τη μετώπιση αυτών, η πρώτη γραμμή άμυνα είναι η πρόληψη αυτοί που έχουν κακή πρόθεση να μην έχουν πρόσβαση στι υπηρεσίε μα στο Facebook. Θα ακούσατε πώ αντιμετωπίζουμε του ψευτικού λογαριασμού. Να βάλουμε το στο πλαίσιο περισσότερε υπηρεσίε στο διαδίκτυο θα έχουν κανόνε ποιο μπορεί να καταχωρηθεί και ποιο όχι, να εγγραφεί και ποιο όχι. Πολλαπλοί λογαριασμοί μπορούν να παραδοθούν ή αυτόματα λογισμικά ρομπότ ή bots ε, που κινούνται αυτόματα και όχι δεν είναι αποτελέσμα ταχύσμου ανθρώπου. Λοιπόν, πρέπει να χρησιμοποιούν στο Facebook την πραγματική του ταυτότητα ή τα μέλη και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τη υπηρεσία του Facebook, όπου έρχονται να μοιραστούν με του φίλου και την οικογένειά του διάφορε πληροφορίε. Και με ρώτησαν πριν το βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίε θα πρέπει να απαιτούν απόδειξη ταυτότητα. Και αυτό καθ' αυτό είναι κάτι επίμαχο στα πλαίσια των συζητήσεων σε αυτή την προστασία των δεδομένων, αλλά σίγουρα αξίζει η διερεύνηση Όπω αναφέρθηκε προηγουμένω, επενδύουμε πολύ στον εντοπισμό και στην πρόληψη εγγραφών παραβίαση στου κανόνες και περιγράψαμε κάποιε μεθόδου που χρησιμοποιούμε, αλλά πέραν από τι τυπικέ μεθόδου, δηλαδή να εξετάσουμε τι πολλαπλές καταχωρήσει από συγκεκριμένη χώρα που γνωρίζουμε ότι είναι υψηλού κινδύνου, Επίση, αντιμετωπίζουμε και πολύ περίπλοκες επιθέσει, προχωρημένε και εταιρείε όπως εμά απασχολούν ε, υπευθύνου για θέματα κυβερνοασφάλεια για να διερευνούν αυτέ τι μορφέ επίθεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητούμε λεπτομερώς δημοσία, διότι δεν θέλουμε να δώσουμε πληροφορίε στου επιτιθέμενους, αλλά θα δείτε από την εμπειρία στο διαδίκτυο και του φορεί έρευνα για το διαδίκτυο στι ΗΠΑ, πληροφορίε που είναι δημόσιε και εκεί θα δείτε ότι δημιούργησαν επί μακρά περίοδο χρονική ε, ρεαλιστικού λογαριασμού για να οδηγηθούν, να εφαρμόσουν τι ε, εκστατείε παραπληροφόρηση. Τώρα έχουμε μια υπογραφή, ένα σήμα αυτή την επίθεση και θα ληφθεί υπόψη στα αντίμετρά μα για την ασφάλεια. Κάποιος ρώτησε για τις ε, ουγγρικές εκλογές. Για κάθε εκλογή μπορώ να πω. Κοιτάμε τις υπογραφές των διαφόρων επιθέσεων ιστορικά, τι έχει γίνει και προσπαθούμε να παρεμποδίσουμε τις επιθέσεις να επαναληφθούν. Όσον αφορά τους ψεύτικους λογαριασμούς, θέλουμε να εμποδίσουμε και την ε, διαγραφή μάλλον να προσπαθούν από δημόσιες σελίδες να συλλέξουν πληροφορίες. Διάφορες ιστοσελίδε μπορεί να δημοσιευσούν και κάποιοι αρπάζουν πληροφορίε και από πληροφορίε πληροφορίες δημιουργούν βάση δεδομένων και δημιουργούμε διάφορα τέτοια σήματα όπω ε, καταχωρήσει εγγραφών. Και στα πλαίσια του θέματος της Cambridge Analytical, ε, πραγματικά όπως περιγράφει έχουν τα πράγματα, θέλουμε να εμποδίσουμε τον κόσμο που νόμιμα έχει πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίε, δημιουργώντας μια εφαρμογή και να χρησιμοποιεί τα στοιχεία για του σκοπούς και δεν συμφωνώ ότι οι αλλαγές είναι διακοσμητικού χαρακτήρα. Εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά βαθιές οι αλλαγές. Ε, το σύστημα που δημιουργήσαμε ε, είχε συγκεκριμένη πρόθεση. Εκείνοι που θέλουν να δημιουργήσουν κάποιες κοινωνικές ε, εφαρμογές, να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές κοινωνικές οι άνθρωποι, να διευκολύνουν κατάσταση, αυτό περιέχει κάποιου κινδύνου και προσπαθούμε να μειώσουμε του κινδύνου και αυτό σημαίνει να μειώσουμε και την πρόσβαση, φυσική πρόσβαση και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στοιχεία οι διάφοροι συμμετέχοντε. Τώρα στου άλλου τομεί, όπου θεωρούμε ότι πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι, πολλού από του εμπλεκόμενου εξετάζουν αυτόματα και ανθρωπίνω τη δραστηριότητα σε μια πλατφόρμα. Πιο προχωρημένο ε, είναι ένα σύστημα είναι κατάχρηση των παιδιών και εκμετάλλευση παιδιών και εκεί έχουμε μπλοκάρει την πρόσβαση σε αυτού του είδους τα στοιχεία. Αυτό είναι κάτι εύκολο, διότι αυτό το υλικό είναι πάντα παράνομο, ούτως ή άλλως δεν τίθεται θέμα. Αν αναρτάται ή όχι, δεν μπορεί να αναρτηθεί νομίμως, αφαιρείται και συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού. Κυρίως με τον πρώτη, την πρώην Επίτροπο κυρία Νέλη Κρούς, η οποία έκανε μια εκστρατεία κάνουμε παρό... και παρόμοιε δραστηριότητε κατά τη τρομοκρατική προπαγάνδα. Συνεργαζόμαστε με εμπλεκόμενου φορεί και τον Επίτροπο Κίνγκ και Αβραμόπουλο εντό του διαδικτύου, του Φόρουμ τη Ευρωπαϊκή Ένωση του Διαδίκτυου και έχουμε κάνει μεγαλύτερη πρόοδο από ό,τι νομίζετε. Και έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε τώρα πάρα πολλέ ε, περιεχόμενο Αλκαίδα και Άισι. Ε, Εμεί πριν μα το καταγγείλουν και πριν το δει κανεί και κατεβάζουμε αυτέ τι αναρτήσει πριν διανεμηθεί και διαδοθεί στην πλατφόρμα μας και θεωρούμε ότι πρωτοβουλίε είναι πάρα πολύ σημαντικέ για εμπιστοσύνη να θεωρήσουν ότι οι υπηρεσίε μα, οι άνθρωποι, είναι προ το κοινό καλό και όχι προ το κοινό κακό. Και άλλου τομεί του οποίου εξετάζουμε αφορούν του λόγου μυσαλλοδοξία με την Επίτροπο Γερόβα. Ε, εδώ είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Πρέπει να καταλαβαίνει κανεί ε, τα υπονοούμενα, ηρωνία κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημειώνουμε και εκεί πρόοδο. Και τέλο, το άλλο θέμα το οποίο συζητήσαμε εκτενώ σήμερα είναι οι ψευδεί ειδήσει εγώ ήμουν στην ομάδα εμπειρογνωμόνων και τώρα συμμετέχουμε στις εργασίες υπό την ηγεσία της Επιτρόπου Γκαμπριέλ και πρέπει να πω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι περιπλοκότερος τομέας ε, διότι κάποιος, ε, κάποιον πολιτική άποψη μπορεί να θεωρηθεί ψευδή είδηση από κάποιον άλλον και πρέπει να δούμε πώς ε, ακριβώς καταλήγουμε στους ορισμούς και έχουμε πρωτοβουλίες ενδιαφέρουσες όπως το γαλλικό κίνημα προ νομοθεσίε σε αυτό το τομέα. Θα είναι κάτι που θα μα βοηθήσει να ενημερωθούμε, αλλά απάντηση και επίλυση του προβλήματο των ειδήσεων πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχει εμπιστοσύνη ο χρήστη. Κεντρικό τομέα όπου εστιάζονται οι προσπάθειε και στο Κοινοβούλιο είναι τα πνευματικά δικαιώματα ότι οι πλατφόρμες δεν χρησιμοποιούνται για να διανέμουν παράνομα έργα που πρέπει να τύχουν προστασίες λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Τελικό τομέα είναι οι διαφημίσεις ε, και η διαφήμιση συζητήθηκε εκτενώς όπως προαναφέρθηκε, πιστεύουμε ότι στο διαδίκτυο διαφήμιση εν γέννη είναι αποδεκτή, αποδεκτός τρόπος για χρηματοδότηση διαφόρων υπηρεσιών του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένη στην δική μας, και έτσι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να πλησιάσουν τους πελάτες που θα πλησιάζαν πριν, διότι η φραγμή ήταν πολύ ψηλή και μπορεί ο κόσμος ε, να έχει κάποιες υπηρεσίες δωρεάν, επειδή χρηματοδοτούνται από τις διαφημίσεις. Μιλάμε για το ψηφιακό χάσμα και όμως Έχουμε υπηρεσίε υψηλής ποιότητα που είναι δωρεάν ε, και έτσι μειώνεται το χάσμα το ψηφιακό και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ευρύτερη πρόσβαση του κοινού αλλά να γνωρίζουμε ότι μπορεί να τύχει κατάχρηση και γι' αυτό έχουμε και όρους για τους ε, που επιβάλλουμε στους διαφημιστές που δεν είναι τους χρήστες για τους διαφημιστές έχουμε υψηλότερες διαγραφέ για το περιεχόμενο από ότι ε, απαγορεύσεις και κάποιο περιεχόμενο που σε ιδιωτικέ αναρτήσεις δεν είναι αποδεκτό σε μια διαφήμιση. Πρέπει να συλλέξουμε και συλλογή πληροφοριών για πληρωμές, πιστοτικές κάρτες κλπ. που κανονικά δεν πρέπει να δώσει ο χρήστης και προσπαθούμε να παρεμποδίσουμε τι απάτες. Επίση στην Ευρώπη συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προστασία του Καταναλωτού, του διάφορου φορεί και υπάρχουν σημεία επαφή του ώστε να μπορούν να δοθούν καταγγελίε όσον αφορά μη αξιοπρεπεί, αν θέλετε, απρεπεί διαφημίσεις και υπάρχουν και διάφορες αυτορυθμιζόμενες πλατφόρμες όσον αφορά τι διαφημίσεις για τον ηχό δεν είναι προ όφελό μα η κατάξυνση των διαφημίσεων και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών να είναι παραπλανητικέ διαφημίσει ή κακή ποιότητα που εμφανίζονται στο σύστημά μα και έχουμε ε, συνεργασίε που έχουμε δημιουργήσει για να το καταπολεμήσουμε. Ένα βασικό σημείο τώρα, όσον αφορά τι εργαλειοθήκε, είναι να διαφανέστερε διαφημίσει. Οι συναδελφοί μου εξήγησαν προηγουμένω πώ το επιτυχάνουμε αυτό. Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια θα βοηθήσει οδήποτε εποπτικό φορέα στον πολιτικό τομέα, στον ευρύτερο τομέα τη προστασία των καταναλωτών εντοπίσει ε, διαφημίσεις που δημιουργούν ανησυχίες ε, που ίσως ε, κρύβουν και κάποιες απάτες. Πού εστιαζόμαστε τώρα όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια. Αυτά, περι... Αυτά είναι που αφορούν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ασφάλεια. Αυτά περιέγραψα. Δημιουργούνται ερωτηματικά και προβλήματα. Κάποιοι έχουν αντίρρηση όσον αφορά την πολιτική μα για πραγματική ταυτότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντική για να παρεμποδίσουμε διάφορε βλάβε ε, που θα προξενούνται διαφορετικά. Υπάρχουν συνεχίε για την αυτόματη διαδικασία και επεξεργασία ε, των στοιχείων για να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο που δεν έπρεπε να εμφανίζεται. Λοιπόν, κάπου στο Βερολίνο κάποιο πολιτικό μα είπε πώ να τα καταφέρουμε τόσο ώστε αυτοί που κάνουν τον έλεγχο να μην πρέπει να βλέπουμε περιεχόμενο φρικτό όπω είναι κατά, ε, ε, τρομοκρατικό περιεχόμενο ή θέματα κακοποίησης παιδιών κλπ. Λοιπόν και το θέμα των διαφημίσεων ε, ε, ήταν αυτό που συζητήσαμε και θέλουμε να είναι φτηνέ οι διαφημίσεις κυρίως για τις νόμες επιχειρήσεις. Είναι ευρύ το θέμα αυτό, είναι ευρύτατα τα διάφορα θέματα. Θα συζητήσουμε εκτενάστερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, περνάμε στις ερωτήσεις. Ξέρετε τους κανόνες. Ένα λεπτό υπάρχει τώρα διαθέσιμο για κάθε ερώτηση. Δύο λεπτά για τις απαντήσεις. Για κάθε απάντηση την ερώτηση θα πρέπει να την απευθύνετε προς ένα άτομο Οι ερωτήσεις ε, θα γίνονται βάσει του συστήματος ΔΕΟΝΤΟ. 14 μέλη έχουν ζητήσει, οπότε ακολουθώντας τον κανόνα όπως έχουμε συμφωνήσει θα, θα δώσω το λόγο στους ομιλητές ε, διαδοχικά. Ο κύριος Ράντεφ από το ΕΛΚ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι για τον Λορδό Άλλα. Να υποθέσουμε ότι το Facebook χρησιμοποιεί κανόνες που διασφαλίζουν την προστασία των χρηστών του, δηλαδή κατά των κυβερνοεπιθέσεων. Ως αποτέλεσμα, ωστόσο, το Facebook δεν ελέγχει τα δεδομένα των χρηστών του και τα προωθεί σε προγραμματιστές και σε τρίτα μέρη και δεν ξέρει ε, πώς προστατεύονται αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο και πώς το Facebook ε, ε, ελέγχει τους προγραμματιστές εταιρείε που λαμβάνουν δεδομένα από χρήστες του Facebook να προστατεύουν τα δεδομένα αυτά από κυβερνού υποθέσεις, ειδικότερα δεδομένων των αρχών 1 και 3 από τη τεχνολογική συμφωνία που η υπέγραψαν πάνω από 40 εταιρείε συμπεριλαμβανομένου του Facebook τον Απριλίο φέτο. και κάτι άλλο το Facebook ε, τι κάνει με αυτούς που δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τα δεδομένα των χρηστών του ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. Very much for that um, Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Να απαντήσω σε δύο τμήματα. Μια, ένα πρώτο κομμάτι πιο ευρέως ως τομέας. Αισθανόμαστε την ευθύνη αλληλοβοήθειας. Σε κάποιους τομείς που περιέγραψα, η δυναμική που επιδιώκουμε είναι οι μεγάλες εταιρείες όπως το Facebook, το Google και οι λοιποί να προσπαθήσουμε να βρούμε μεθόδους ε, να χρησιμοποιούμε από κοινού πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με τις άλλες εταιρείε. Η κυβερνοασφάλεια δεν πρέπει να είναι ένας τομέας ανταγωνιστικός ούτε τομέας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Προσπαθούμε μάλλον να θα πρέπει να προσπαθούμε να προστατεύσουμε ολόκληρο το οικοσύστημα με εργαλεία όπως ανταλλαγές απειλών, threat exchange κτλ. Χρησιμοποιώντα από κοινού, ανταλλάσσοντα πληροφορίε για να είμαστε όλοι ασφαλεί. Και θέλω να είμαι σαφή. Όταν μια εταιρεία έχει μια δυναμία, δηλαδή αν κάποιοι κακόβουλοι αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα σύστημα και χρησιμοποιήσουν ε, τα δεδομένα αυτά για να μπορούν να περάσουν σε άλλα συστήματα, γι' αυτό μα συμφέρει όλου να είμαστε ασφαλεί. Το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης αφορά έναν πολύ ενδιαφέροντα τομέα. Την ευθύνη μεταξύ ενός πρώτου μέρους και ενός τρίτου μέρους όπου πηγαίνουν τα δεδομένα. Σαφώς το Facebook μετά από την κατάσταση με την Cambridge Analytica το εξετάζει όλα αυτά σε βάθος. Ορισμένα μέτρα που έχουμε λάβει ήταν μειωμένη πρόσβαση ε, και έλεγχος αυτό που αναμένει ο κόσμος από εμά. Αλλά ξέρετε, όλοι μας έχουμε ένα τηλέφωνο στο χέρι μας, όλοι εφαρμο... Ε, καθιστάμε εφαρμογές καθημερινά και κατά την εγκατάσταση εφαρμογών πάντα μεταβάζονται δεδομένα. Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση που κάνετε. Δεν μπορώ να σας δώσω μια απάντηση ε, για το πόσο δύσκολη πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία, ε, πόσα εμπόδια πρέπει να βάλουμε στην πλατφόρμα, στο χρήστη και στο τρίτο μέρος θα πρέπει να γίνει ένας ανοιχτός διάλογος για όλα αυτά ε, ε, και να πούμε όλα θα τα κάνει το πρώτο μέρος, τότε θα πρέπει να κλείσουμε την πλατφόρμα γιατί δεν θα είναι ανταγωνιστική και σταματάμε την καινοτομία. Αν δεν αναλάβει καμία ευθύνη όμως το πρώτο μέρος, τότε ο κόσμος ενοχλείται. Οπότε πρέπει να γίνει ένας διάλογος. Πρέπει να δούμε πώς θέλουμε να επιμεριστεί η ευθύνη ώστε να υπάρχει προστασία των δεδομένων χωρίς ε, υπερβολικά εμπόδια σε όσους προσπαθούν να κινηθούν online νόμιμα. Η Birgit Zippel από τους σοσιαλιστές έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα μπω σε άλλη διαμάχη με υπάλληλο του Facebook, αλλά κατάλαβα ότι το να φτιάχνει μια εφαρμογή σου δίνει ήδη αρκετά μεγάλη και ευρεία πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Κάτι που είναι απαράδεκτο αν δείτε τι έχουν, έχει γίνει σε άλλου τομεί. Θέλω όμω να απευθύνω ένα ερώτημα στην κυρία Πάχαλ. Γιατί πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τι ψηφιακέ υπηρεσίε χωρί να γνωρίζουν ακριβώ τι ακριβώ συμβαίνει και πώ ακριβώ ε, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του, πώ ε, δημιουργούνται προφίλ για αυτού. Δεν το γνωρίζουν αφού δεν είναι και δυνατόν. Επίσης, να ξέρουν ε, τι είναι ένας ψεύτικος λογαριασμός και πώς ακριβώς δημιουργείται. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς λοιπόν, προκειμένου να εφαρμόσουμε τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ε, θεωρείτε ότι χρειαζόμαστε και την ιδιωτική ασφάλεια και ιδιωτικότητα, την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα, χρειάζεται οι οργανώσεις νεολαίας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ασχοληθούν με τον αλφαβητισμό στην ψηφιακή εποχή. υπάρχει, εξ όσων γνωρίζετε, κάποια συνεργασία με τους υπεύθυνου ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων ε, των εταιριών και ποια μορφή έχει, αν όντως υπάρχει ήδη κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ζίπελ. Προφανώς μας απασχολούν όλα αυτά. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, ας το ξεκαθαρίσουμε. Ο GDPR έχει εξορισμού ε, και βάση σχεδιασμού αυτή την ε, έννοια της ιδιωτικότητας. Και αυτό ακριβώς είναι και το σημαντικότερο. Να γνωρίζουν οι χρήστες ε, ότι καταρχήν οι υπηρεσίες που χρησιμοποιώ προστατεύουν την ιδιωτικότητά μου και ε, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μου δίνονται εχέγγυα για την προστασία της ιδιωτικότητάς μου, της ιδιωτικής μου ζωής. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο ε, οι πλατφόρμες θα παρουσιάζουν τις διάφορες επιλογές στους χρήστες τους είναι πολύ σημαντικός. Η ηλεκτρονική ιδιωτικότητα θα είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο, γιατί ο GDPR δεν επαρκεί όσον αφορά τη στόχευση χρηστών και τη διαφήμιση. Χρειαζόμαστε λοιπόν και την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα, τη σχετική οδηγία ε, και ελπίζουμε στο Κοινοβούλιο να κάνει ό,τι μπορεί. Ο αλφαβοτισμός στα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικός, η ευαισθητοποίηση Επίσης και εμείς οι ίδιοι χρησιμοποιούμε εφαρμογές προκειμένου να ενημερώνουμε τους χρήστες, τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους και τους τρόπους που έχουν για να υποβάλουν καταγγελίες. Ε, επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο του GDPR είναι ότι οι αρχές ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων έχουν πλέον νομική υποχρέωση να απαντούν σε καταγγελίες που δέχονται και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό δίνει και περισσότερο κίνητρο στους χρήστες να κάνουν τέτοιες καταγγελίες αυτά η γενική ευαισθητοποίηση του κοινού είναι σημαντική, αλλά δεν χρειάζεται και να πλημμυρίσουμε τους ε, χρήστες και τους καταναλωτές με υπερβολικές πληροφορίες. Πρέπει κατά βάση οι ίδιες εταιρείε να αλλάξουν νοοτροπία όσον αφορά τον ε, χειρισμό και την επεξεργασία στο προσωπικό δεδομένο. Γιατί ε, ξέρετε ότι και στη Γερμανία αυτή τη στιγμή ε, το Facebook έχει γίνει αντικείμενο ελέγχου των αρχών τήρησης και προστασίας του ανταγωνισμού. Γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Κύριε Ντεμόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είχα μια ερώτηση να αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών των χρηστών ε, που αφορά διάφορα θέματα. Το πρώτο θέμα, το ερώτημα για τον Λόρντο Άρλαν. Ερώτηση. Όσον αφορά τα ψευδείς ειδήσει και τα συστήματα των ψεύτικων λογαριασμών, γιατί περιοριστούμε σε αυτή την εγγραφή που είναι τόσο κοινότοπη. Μήπως θα ήταν καλύτερο να έχουμε ένα σύστημα ε, εξακρίβωσης με κώδικες που αποστέλλονται στον αριθμό του κινητού του κατόχου και μετά συνεχίζω. Άλλη ερώτηση. Με το 2011. Το 2011 όταν μαθεύτηκε ότι υπάρχει αυτή η διάδοση στοιχείων που δεν ήταν ε, νόμιμη, ποια ήταν η αντίδραση εντός των κύκλων του Facebook, πώς συμπεριφερθήκατε, πώς κινηθήκατε, τι είδου μέτρα υιοθετήσατε και αν οι Ιρλανδικές αρχές ε, διέκοψαν αυτή τη διαβίβαση των στοιχείων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει. Καταρχάς, όσον αφορά την εξεκρίβωση, την επαλήθευση των λογαριασμών, χρησιμοποιούμε κώδικες που στέλνουμε στα κινητά ε, τηλέφωνα για, σαν ένα συμπληρωματικό στοιχείο για να μπορεί κανείς να εισέλθει στους λογαριασμούς. Δεν ζητούμε επί του παρόντος για την εγγραφή ε, πραγματικά ονόματα και άλλες πληροφορίες ταυτότητα, εκτό από αυτό που εξήγησε ο ο συνάδελφο, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο λογαριασμό. Αν μα έχει καταγγελθεί ότι ενδεχομένω μπορεί να είναι ψεύτικο αυτό ο λογαριασμό, εκεί μπορούμε να ζητήσουμε κάποιες πληροφορίες, μας στείλουν περισσότερε πληροφορίε για το πώ λειτουργούν τα διάφορα συστήματα και που χρησιμοποιούμε κωδικού μέσω SMS είναι αν κάποιο προσπαθεί να μπει στο λογαριασμό σα από περίεργη τοποθεσία για να εμποδίσουμε αυτού του είδου την πρόσβαση ε, στο λογαριασμό παρά για εξακρίβωση ταυτότητα. Είμαστε πολύ ανοιχτοί όσον αφορά αυτό το θέμα, το συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι κάποιοι από την άλλη πλευρά του επιχειρήματο θα πούν ότι δεν ενδείκνεται να συλλέγουμε ίσω τι πληροφορίε να ζητούμε αριθμού τηλεφώνων. Ε, ζητούμε αριθμού τηλεφώνων και προβληματίζονται κάποιοι. Όσον αφορά τη διαδικασία μετά το 2011, υπήρχαν δύο προσεγγίσει για τι ρυθμιστικέ αρχέ όσον αφορά ένα φορέα όπω είμαστε εμεί που είμαστε ρυθμιστικό. Πρώτα απ' όλα περιμένει κανεί μέχρι να υπάρξει ένα πρόβλημα και μετά να γίνει δίωξη και αυτό είναι ένα λογικό, λογική προσέγγιση. Το άλλο είναι διαδραστική προσέγγιση. Λέμε στου άλλου να πώ μπορείτε να βελτιωθείτε, τι βελτιώσει περιμένουμε και ερχόμαστε και κάνουμε μια επαναξελόγηση. Και με την Επιτροπή Προστασία Δεδομένων τη Ιρλανδία. Αυτό ακολουθήσαμε. Ήρθαν στα γραφεία μα, συζητήσαμε τι καταγγελίε του Μαξ ε, ένα ένας ταπεινός φοιτητής της νομικής από την Αυστρία που έκανε καταγγελίες ε, και η Επιτροπή λοιπόν ε, εξόδευσε πολύ χρόνο. Βάλαμε εκατοντάδε ανθρώπου να εξεργαστούν τα θέματα, πρότειναν κάποιε αλλαγέ. Αν δεν αρκούσαν, ζητήσαν ναι και άλλε. Αυτή ήταν μια αμφίδρομη διαδικασία που επανατροφοδοτεί το. Αγγέλικα Μίρνερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σαν να έχουμε Αυστριακή Προεδρία όλο το απόγευμα. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση. Ήθελα σε σχέση με το όσο είπε ο Μαρκ Σρέμς ε, είναι διαμετρικά αντίθετα αυτά που είπατε με όσα ακούσαμε, ακούγαμε όλο το απόγευμα ότι ουσιαστικά καθόλου ευρωπαϊκά δεδομένα δεν χρησιμοποιήθηκαν στην υπόθεση Cambridge Analytica και εσείς κύριε Σρέμς είπατε κάτι άλλο το οποίο καθιστά προφανές ότι δεν μπορούν να ισχυριστούν κάτι τέτοιο. Αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω προς εσάς λοιπόν, ε, Λόρδε Ρίτσαρντ Άλαν. Πώς απαντάτε σε αυτό, γιατί ήσασταν εδώ ολόκληρο το απόγευμα και η επίσημη εκδοχή του Facebook είναι ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκά δεδομένα. Και άλλη μια ερώτηση, πολύ συγκεκριμένη, είμαι φιλελεύθερη, στο κόμμα μου το GDPR και η προστασία των δεδομένων ε, είναι σοβαρά θέματα και εμείς ε, βρήκαμε ότι σύμφωνα με του εμπειρογνώμονε, του ειδικού τη προστασία των δεδομένων, εγώ ω πολιτικό δεν μπορώ πια να χρησιμοποιήσω το WhatsApp λόγω του mining όλων των δεδομένων που έχω στο τηλέφωνό μου. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, συμβαίνει αυτό ή όχι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ συγκεκριμένα τώρα για την κατάσταση της Cambridge Analytica που θέλω να την εξηγήσω. Υπάρχουν ευρύτερα ζητήματα για το κατά πόσο συγκεκριμένες εφαρμογές ε, ε, χρησιμοποιούν δεδομένα με τρόπους αθέμητους. Και εμείς προσπαθούμε να ε, καταπολεμήσουμε αυτή την κατάχρηση. Η Cambridge Analytica είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είχε ένα συμβόλαιο με την GSR του Alexander Kogan και εκεί είπαν συλλέξτε δεδομένα των Αμερικανών για να χρησιμοποιηθούν σε αμερικανικές πολιτικές εκστρατείες, προεκλογικές εκστρατείες και το 97% των ανθρώπων ε, που εγκατέστησαν τις εφαρμογές του Κόγκαν ήταν Αμερικανοί και εκεί πήρε τα δεδομένα ο Κόγκαν μαζί με κάποια ευρωπαϊκά δεδομένα αλλά τα δεδομένα που έδωσε στην Cambridge Analytica ήταν αμερικανικά γιατί αυτά ήθελαν. Αυτό προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε. Αν λοιπόν εσεί θέλετε να επενδύετε ότι η Cambridge Analytica έχει στα χέρια τη ε, διάφορα ευρωπαϊκά δεδομένα για να τα χρησιμοποιήσει για εκστρατείε προεκλογικέ στην Ευρώπη, αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχουμε τίποτα που να το αποδεικνύει αυτό. Ωστόσο, θα κάνουμε τον έλεγχο πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο για να το επικυρώσουμε. Αλλά η αλυσίδα των γεγονότων μα λέει ότι ουσιαστικά ω επιτοπλίστων συνέλεξαν αμερικανικά δεδομένα και αυτό λέει ότι έδωσε αμερικανικά δεδομένα. Αλλά απομένει να επιβεβαιωθεί. Θέλουμε να είμαστε απόλυτα διαφανεί με αυτό. Για το άλλο ερώτημα, μου κάνει έκπληξη. Όπω το έχουμε καταλάβει εμεί, ε, το WhatsApp έχει μια από τις καλύτερες πολιτικές προστασίας. Ε, το ξέρει ο κόσμος. Έχει κρυπτογράφηση για όλους τους χρήστες. Ε, κανείς στο Facebook ή στο WhatsApp δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας λόγω του τύπου κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν αυτές οι εφαρμογές. Υπάρχει υπερβολικά μεγάλη προστασία κάποια ερωτηματικά όσον αφορά τι λίστε επαφών και όλα αυτά. Μπορούμε να τι συζητήσουμε, αλλά για τα βασικά δεδομένα, τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται με πολύ ισχυρή κρυπτογράφηση. My question goes to Max uh, ε, ξέρω δύο μοντέλα. Ή, ή θα βγάλεις λεφτά στο δίκτυο με τη διαφήμιση ή με τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτά τα δύο συστήματα υπάρχουν. Και αυτά άλλωστε είναι εκείνα που κατέστησαν και δυνατή τη χρήση του διαδικτύου. Αυτό άλλωστε ε, προκάλεσε και την εκτόξευση της χρήσης των κοινωνικών ε, δικτύων. Αφενό λοιπόν υπάρχει η διαφήμιση, από την άλλη μεριά υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα, που σημαίνει ότι πρέπει οι δημοσιογράφοι, οι δημιουργοί περιεχομένου να αμείβονται. Και αυτό δυστυχώς είναι ένα στοιχείο που πολλές πλατφόρμες ηλεκτρονικές αρνούνται στους ε, ε, δημιουργούς. Πώς λοιπόν μπορούμε να συμβιβάσουμε αυτέ τι δύο πλευράς. Δεν ξέρω αν είμαι ο καταλληλότερος για να απαντήσω, αλλά μπορώ να σας ε, δώσω κάποια στοιχεία που ενδεχομένως απαντούν στο ερώτημά σας. Πρώτον, πρέπει να επανεξετάσουμε. Και αν κρατήσετε ένα πράγμα από την σημερινή ακρόαση, κρατήστε το εξή. Η online διαφήμιση δεν καθοδηγείται μόνο και αυτόματα από τα προσωπικά δεδομένα. Δεν χρειάζεται. Αν δηλαδή ε, κάτι στο πλαίσιο μιας διαφήμιση. Για παράδειγμα, μια διαφήμιση αυτοκινήτου σε μια σελίδα που, για τα αυτοκίνητα. Αυτό δεν χρειάζεται βεβαίως προσωπικά δεδομένα. Ο κλάδος απλά προσπαθεί να συμβιβάσει και να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και στην τηλεόραση, που δεν υπάρχει καθόλου στόχευση ως προς τις διαφημίσεις, στόχευση των χρηστών εννοώ. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Στην online διαφήμιση λοιπόν, χωρίς να έχω και εγώ τις τελικές απαντήσεις που μπορώ να σας δώσω, πρέπει να δούμε ποιος βγάζει ποια χρήματα και πόσα. Ε, μιλούσα πρόσφατα με έναν ε, εκδότη από την Αυστρία και ε, μου ανέφερε ότι στην στοχευμένη διαφήμιση λιγότερα χρήματα βγάζουν από ότι στη μη στοχευμένη, διότι το YouTube και το Facebook παρακρατούν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαφημιστικής διαπάνησης υπέρ του εαυτού τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας πρέπει να μπούμε πολύ πιο βαθιά. Ε, δεν αρκεί να πούμε όχι πλέον cookies. Είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένο και πολύ περίπλοκο το πρόβλημα. Και επειδή έχω λίγα μόνο δευτερόλεπτα στη διάθεσή μου και επειδή ο Ρίτσαρντ είπε ότι χρειάζεται να συζητήσουμε την ευθύνη των τρίτων, τότε δεν χρειάζεται, ε, εγώ θα έλεγα, δεν χρειάζεται καθόλου να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Υπάρχει πλέον στο άρθρο 26 και 27 του GDPR και υπήρχε και στην προηγούμενη, στην παλαιότερη οδηγία. Άρα καθόλου ανάγκη συζήτηση δεν υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα, διότι τα θέματα αυτά ήδη ρυθμίζονται από την νομοθεσία. Ευχαριστώ. Η Μίρια Μνταλή, επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτησή μου απευθύνεται στον κ. Σάλμστιτ. Λοιπόν, έχετε βρει κάποιες ερμηνείες νομοθετικές, λαμβάνοντας υπόψη τα προσωπικά δεδομένα στην Ευρώπη. Και ε, οι αποφάσεις των δικαστηρίων επηρέασαν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ανώσης και την εφαρμογή. Μας ενδιαφέρει πολύ τι θα γίνει με τη μελλοντική νομοθεσία. Κάπου κάνατε μια ερώτηση. Είπατε. Θα αλλάξει με το GDPR το θέμα. Με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Θα σταματήσει το GDPR την εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων. Εσείς που ενεργοποιείς τον τομέα τη μεταρρύθμιση τη ηλεκτρονική ιδιωτικότητα που έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο, πόσο σημαντική τη θεωρείτε και το μελλοντικό νομικό πλαίσιο θα μπορεί να αποτελέσει λύση, να καλύψει κενά. Και ποιες προτεραιότητες πρέπει να τεθούν. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Για, την, για το e-privacy βγήκα εκτός συζητήσεων. Βαρέθηκα τις βρυξές μετά από χρόνια συζητήσεων για το GDPR. Πρέπει όμως να ευθυγραμμιστεί τελικά το σύστημα με το GDPR. Δεν θα πρέπει ε, να θεωρείτε ότι ε, σαν δεδομένο ότι σαν αρχική προϋπόθεση θα διαβιβάζω τα δεδομένα και θα αντιβαίνει το GDPR. Για το GDPR θα είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ποια είναι η πολιτική ιδιωτικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων και εξεπλάγει από το πόσο αγνόησαν πολλά που θέματα που συζητήσαμε. Οι πρώτες καταγγελίες ήταν για καταναγκαστική σύμφωνη ε, Τώρα το προϊόν συνδέεται με την ε, συνένεση. Το αγνοούσαν οι επιχειρήσει. Το Facebook έλεγε πρέπει να συμφωνήσετε αλλιώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία. Ποια είναι η θεωρία πίσω από αυτή τη θέση. Νομίζω δικαστικά θα, θα καταπέσει, θα κοστίσει μέχρι το 4% του ΑΕΠ. Δεν ξέρω αν θα το προσεγγίσουν ή θα συνεχίσουν θα επιμείνουν. Αλλά αγνοείται το GDPR, θα συνεχιστεί αυτό. Έχω την εντύπωση ότι αντιδρούν οι επιχειρήσεις να μην μας ελέγχουν οι Ευρωπαίοι. Αν μας ελέγξουν οι Ευρωπαίοι λένε μεγάλες επιχειρήσεις, ο υπόλοιπος κόσμος θα μας πίεσει. Πρόκειται περί αγνίας, περί μη συμμόρφωσης, διαφορετικές ερμηνείες. Αλλά νομίζω ότι αγνόησαν την νομοθεσία μεγάλες επιχειρήσεις. Ελπίζουμε τελικά το 4% ότι θα λειτουργήσει. Φοβούνται τα, τα αντίμετρα της κυρώσεις οι μικρές επιχειρήσεις. Γι' αυτό προσφεύγουμε στα δικαστήρια για να υποχρεωθούν οι αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο και να μπορούν να υπάρχουν προσφυγές. Πιστεύω ότι θα υπάρχει διαφορά στις αντιδράσεις των διαφόρων κρατών μελών ανάλογα με την νομοθεσία τους. Ο κ. Μπουτικόφερ έχει το λόγο. Λόρδε Άλλαν, με ενοχλείτε με τον γοητευτικό σας κινησμό όταν λέτε ότι οι γνώμες δίστανται συχνά σε θέματα όπως ενημερωμένη συνένεση, συνένεση βάση γνώσης. Αυτός μεταφράζεται στο εξή. Παρότι ξέρουμε ότι παραβιάσαμε τον νόμο, δεν μπορούμε να πληρώνουμε ακριβώ δικηγόρου. Αυτό λέτε. Οπότε δεν θα κάνω ερώτηση σε εσά. Θα ρωτήσω την κυρία Πάκλ. Μπορείτε να εμβαθύνετε λίγο στα ζητήματα που θίξατε όσον αφορά τη συλλογική αποζημίωση, όσον αφορά τη λογοδοσία των πλατφορμών και τα λοιπά μέτρα. Θέματα όπως αλγοριθμική παρακολούθηση ή αλγοριθμική ηθική είναι θέματα για τα οποία θα μας συμβουλεύατε να εστιαστούμε ή πού θέτετε εσείς προτεραιότητα. Λοιπόν, να τα διαχωρίσουμε λίγο. Η συλλογική ε, προσφυγή θέλω να είμαστε σαφείς ο GDPR δεν προβλέπει συλλογική προσφυγή είναι μύθος αυτό το ακούμε δεξιά και αριστερά δεν συμπεριλαμβάνεται στο GDPR στο GDPR απλά το κράτος μέλος έχει την επιλογή να ε, εξουσιοδοτήσει οργανισμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων να προχωρήσουν σε συλλογικές δράσεις, να ε, ε, σταματήσουν παράνομες συμπεριφορές, αλλά μόνο αν αυτοί οι οργανισμοί έχουν λάβει εντολή από καταναλωτές ή από ενός καταναλωτών. Εκεί μπορούν να ζητήσουν να κάνουν προσφυγή. Το GDPR δεν, δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, αλλά η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Απριλίου για την προστασία των καταναλωτών περιλαμβάνει συλλογική προσφυγή για παραβιάσεις ε, της προστασίας των δεδομένων. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή το μέσο συλλογική προσφυγής να υιοθετηθεί το συντομότερο δυνατόν από τους νομοθέτες ώστε να έχουμε σίγουρα κάτι απτό στα χέρια μας το οποίο, στο οποίο μπορούμε να προσφύγουμε σε περίπτωση παραβίαση ε, ε, μαζικής κλίμακας τέτοιων δεδομένων γιατί αυτή τη στιγμή μόνο τέσσερα κράτη-μέλη προβλέπουν τέτοια προστασία για τους οργανισμούς καταναλωτών και στην περίπτωση του Facebook έχουν προσφύγει στα δικαστήρια ή θα το κάνουν με τι επόμενε ημέρε. Αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη δεν διαθέτει τέτοια μέσα. Οπότε μιλάμε για συλλογικέ προσφυγέ. Τώρα, όσον αφορά του αλγόριθμου, είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα αυτό, πιστεύω. Και αφορά ιδιαίτερα τον GDPR, ειδικότερα δεδομένη τη αυξημένη χρήση των αλγορίθμων για αυτόματη λήψη αποφάσεων ε, και για την τεχνητή νοημοσύνη. Και ένα από τα ζητήματα κλειδί είναι ότι θα πρέπει να διερευνήσουμε ε, στα θέματα τη εφαρμογή και τη ερμηνεία τη νομοθεσία τι δικαιώματα έχουν οι πολίτες όταν λαμβάνετε μια αυτοματοποιημένη απόφαση ότι θα έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα πράγματα βάσει των προσωπικών σας δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για να ληφθεί η απόφαση του κατά πόσο θα σας αποκλειστείτε από κάτι ή όχι και ο GDPR λέει ότι έχετε το δικαίωμα να λάβετε εξηγήσει. ότι έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε την απόφαση αυτή αλλά υπάρχει και κάποια βεβαιότητα. Οπότε ε, σίγουρα αυτό είναι κάτι για το οποίο θέλουμε μια σαφέστερη ερμηνεία από τα δικαστήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Τελβό, Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ στην κυρία Πάχλ θα κάνω μια ερώτηση. Εγώ συμμετείχα και στις ε, δύο ε, διοργανώσεις αυτής της ακρόασης και είχα θέσει το ερώτημα τι νόημα έχει να θέτουμε ε, ερωτήματα όταν η απάντηση που παίρνουμε είναι τα πάντα είναι μια χαρά. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση ότι καθόλου καθόλου καλά δεν μας τα λέτε. Ευτυχώς έχουμε αυτή τη νέα νομοθεσία και ευτυχώς οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων μας θα έχουν πλέον την εξουσία να την επιβάλλουν την νομοθεσία αυτή. Είναι μια πρόκληση βεβαίως Ιδίω ε, όσον αφορά την εναρμόνιση και την εναρμόνιση προσέγγιση που θα πρέπει να επικρατήσει στα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό το 4, η απειλή του 4% μπορεί και να αποδειχθεί ε, επαρκής. Άλλο μέσο που έχουν στη διάθεση πλέον οι καταναλωτέ είναι και αυτή η συλλογική προσφυγή. Πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε την ηθική βλάβη που μπορεί κανείς να υποστεί μέσω παραβίασης των προσωπικών του στοιχείων. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό νομίζω ότι είναι από τα βασικά βασικά ζητήματα του, που μας απασχολούν. Δεν έχω έτοιμη απάντηση, αλλά μπορώ να κρατήσω ότι ο GDPR ε, αναγνωρίζει ότι υπάρχει υλική και μη υλική ζημία, βλάβη που μπορεί να προκαλέσει μια παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Άρα αυτό αναγνωρίζεται πλέον σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει βλάβη. Δεύτερο στοιχείο, η αξία των ε, δεδομένων είναι κάτι που δεν έχει τυποποιηθεί, δεν έχει μετρηθεί ούτε ποσοτικοποιηθεί ακόμα, δεν υπάρχει ακόμα επαρκής νομολογία. Ο Μαξ μπορεί ενδεχομένω να δώσει περισσότερα στοιχεία ως προς αυτό και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει, πώς θα αποφανθεί το δικαστήριο όταν οι οργανώσεις μας προσφύγουν. Ζήτησαν 200 ευρώ ανά υποκείμενο δεδομένων στην υπόθεση Cambridge Analytica ε, επί όλους τους χρήστες που τα δεδομένα τους παραβιάστηκαν. Σας το λέω αυτό ενδεικτικά. Πάντως η βλάβη, η ζημία δεν είναι μόνο οικονομική που είναι και δύσκολο να αποδειχθεί και να θεμελιωθεί. Ε, πρέπει να υπάρχει αποζημίωση και για την μη οικονομική ζημία που έχει προκληθεί από παραβίαση. Αυστριακό δικαστήριο ε, επιδίκασε 750 ευρώ αναπερίπτωση και μάλιστα στον Καναδά ε, αντίστοιχες υποθέσεις δικαστήρια κατέληξαν έως και 25.000 ευρώ καναδικά δολάρια αποζημίωση για, για περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Τα 200 ε, ευρώ λοιπόν θα έλεγα ότι είναι το απόλυτα κατώτατο όριο που μπορούμε να προβλέψουμε αυτή τη στιγμή. Η κυρία Κορνέλια Έρνστ. Ευχαριστώ πολύ. Για τον Μαξ έχω ένα ερώτημα. Έχουν υπάρξει πολλές καταγγελίες, παράπονα, ε, προσφυγές από τη δική σας πλευρά που στέφθηκαν και με επιτυχία μάλιστα και μπράβο σας φυσικά. Το ερώτημα λοιπόν είναι ε, οδή προσφυγής, ε, αρχές κτλ. Το ερώτημα μου είναι το εξή. Τι πρέπει να κάνει η Facebook για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του Max Rems. Και δεν είναι ασήμαντο αυτό, γιατί υπάρχουν προσφυγέ και εναντίον άλλων εταιριών όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Δεύτερο ερώτημα. Τι συμβαίνει με τις εποπτικέ αρχές και σε ποιο βαθμό πράγματι είναι ικανές οι αρχές αυτές να διενεργούν τους ελέγχους που προβλέπονται. Και τρίτο ερώτημα, πολύ σύντομο. Θέλω να συμφωνήσω με την ε, συνάδελφο από τους ε, φιλελεύθερους για το WhatsApp θα ήθελα να μας πείτε και εγώ να μας πείτε περισσότερα στοιχεία. Να ξεκινήσω για το WhatsApp, λοιπόν. Λοιπόν, καλύτερα στοιχεία ε, δίδονται, καλύτερα στοιχεία διαβάζονται από ό,τι στο Facebook. Δεν μπορώ να σα δώσω περισσότερες πληροφορίες. Θα ήταν όμως χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την επισήμανση για τις αρχές. Με το GDPR έχουν τα εργαλεία και τις δυνατότητες έρευνας οι αρχές να επιβάλλουν κυρώσεις. Το θέμα δεν είναι νομοθεσία, αλλά η νοοτροπία όσον αφορά την ιδιωτικότητα. Εγώ, σαν απλός δικηγόρο, μπήκα στον τομέα της ιδιωτικότητα. Λοιπόν, περιμένει κανείς αν κάνει κάτι λάθο, παράβαση, θα πληρώσει το τίμημα, μία κύρωση. Με την ιδιωτικότητα, αν παραβιάσει την ιδιωτικότητα, κανείς δεν την πληρώνει. Ξεκινήσαμε παλιά με, ένα, με ήπια νομοθεσία ότι χρειάζεται συμμόρφωση κλπ. Τι πρέπει να δούμε τα δύο-τρία χρόνια τα επόμενα. Αν πρέπει να επικρατήσει μια νοοτροπία συμμόρφωσης μέσω επιβολής κυρώσεων στην Ευρώπη. Αν θα αλλάξει αυτό ή όχι. Θα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στις διάφορες χώρες και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει. Τι να κάνει το Facebook για να συμμορφωθεί. 90 με 95% της διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων είναι κάτι ορθό και νόμιμο. Ταιριάζει στο προϊόν που παρέχουν. Και, και ακόμα και στα πλαίσια καταγγελία μπορούν να συμμορφωθούν εύκολα. Υπάρχει θέμα ανοτροπίας. Άλλη προσέγγιση των ΗΠΑ, σύμφωνα με την νομοθεσία τη Καλιφόρνια, κινούνται στην Αμερική και η ευρωπαϊκή προσέγγιση έχει διαφορετικές δομέ. Θέλουν ένα γενικό σύστημα στην Ευρώπη. Γι' αυτό υπάρχει το πρόβλημα. Και στις διαφημίσεις. Θα μπορούσαν να λυθούν τα προβλήματα. Θα έβγαζε λιγότερα λεφτά βέβαια το Facebook, θα λυνόταν πολλά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Άλλο. Το ερώτημά μου απευθύνεται στον, Λόρτ Άλλαν. Με ενδιαφέρει Πώς λειτουργεί αυτή η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και πώς αξιολογείται την έως σήμερα δραστηριότητα της Ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θεωρείτε ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Κοιτάξτε, είχαμε θετικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια και μήνες. Γιατί θέλαμε να συμμορφωθούμε το GDPR. Ήρθαμε σε επαφή με πολλούς φορείς προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη. Στο παρελθόν φαινόταν ότι συνεργαζόμαστε κυρίως με τους Ιρλανδούς στα πλαίσια του οδηγίας. Τώρα, όλο και πιο συχνά, συνομιλούμε με πολύ περισσότερους αρμόδιους φορείς χωρών μελών της Ένωσης. Συνομιλήσαμε συνεργαστή με τον Στίβεν Τέντμαντ που πριν έρθει στο Facebook είχε ασχοληθεί σε αυτό το τομέα ε, στα πλαίσια του GDPR έχει σοβαρά καθήκοντα και κυρίως να έχετε σε επαφή με τις αρχές προστασίας των δεδομένων. Δεν θέλω να φανεί ότι προστατεύω όλα όσα κάναμε κατά το παρελθόν. Κάναμε λάθη. Επικριθήκαμε. Με κάποιες επικρίσεις συμφωνούμε. Με κάποιες επικρίσεις διαφωνούμε. Ίσως οφείλονται όλα αυτά και σε κάποιες ε, ε, ερμηνείες του νόμου. Κάποιες υποθέσεις κερδίσαμε, σε άλλες τις, άλλες χάσαμε, κάπου είχαμε δίκιο, κάπου είχαμε λάθος. Θέλουμε να συμμορφωθούμε το GDPR. θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές προστασίας δεδομένων. Θα ήθελα να κλείσουμε το MyCrump το, το κενό του 5 μέχρι 10%. Θα μας διευκόλυνε αν ικανοποιηθεί και νομίζω ότι είναι ένας στόχος που μπορούμε όλοι να θέσουμε για τον εαυτό μας. Η Ιζαμπέλα έχει το λόγο. Λόρδε Άλεν δεν με πείσατε πριν. Αν πραγματικά πρέπει να πολεμήσετε, θέλετε να πολεμήσετε τα fake accounts, πρέπει να έχετε ένα σοβαρό σύστημα. Τη στιγμή τη εγγραφή στέλνετε έναν κώδικα ασφαλεία, εξακρίβωση σε ένα κινητό τηλέφωνο και αυτό πιστεύετε ότι θα λύσει πολλά προβλήματα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι διαφορετικά αυτή η ανακοίνωση ότι θέλετε να επιλύσετε τα προβλήματα αυτών των fake accounts ε, μας κορυδεύει. Όσον αφορά την νομοθεσία ή την ιδιωτικότητα για το privacy. Σύμφωνα με την, με την παλιά νομοθεσία και τη βάση δεδομένη ήταν η καθημερινή ε, privacy policy όσον αφορά την προστασία των νόμιμων συμφερόντων, ποιο είναι το νόμιμο συμφέρον, να χρησιμοποιηθεί το δεδομένο για, να, για, για κερδοφορία. Τι σημασία έχει αυτή, αυτή η διατύπωση, ποια είναι η έννοια όσον αφορά τους fake accounts. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι πραγματικά χωράει πολλή συζήτηση εδώ πέρα δεν έχουμε πειθεί μέχρι στιγμής ε, ότι η συλλογή παραπάνω ευαίσθητων πληροφοριών είναι απαραίτητη για την επαλήθευση κάποια ταυτότητα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε σε πολλά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, το ζήτημα αυτό ε, υπάρχει περιθώριο να συζητηθεί. Εμεί, όπω το έχουμε καταλάβει προ το παρόν, είναι ότι όταν έχουμε σοβαρέ αμφιβολίε για την ταυτότητα κάποιου, και πιστεύουμε ότι μπορεί να πρόκειται για ψεύτικο λογαριασμό. Εκεί αιτιολογείται να ζητήσουμε παραπάνω πληροφορίε. Αλλά το να ζητάμε παραπάνω πληροφορίε από όλου του χρήστε του Facebook δεν συνιστάται. Τώρα η πολιτική του Facebook μπορεί να αλλάξει με τον καιρό, μπορεί οι χώρε να νομοθετήσουν διαφορετικά ε, σε χώρε όπω η Εστονία όπου υπάρχει ψηφιακή ταυτότητα, ναι, μπορεί να θελήσουν να νομοθετήσουν Οπότε δεν θέλω να σας πω ότι δεν μας ανησυχεί το πρόβλημα, απλά πρέπει να ζυγίσουμε κάπως τα ασφάλεια και ε, τη συλλογή των δεδομένων, να μην συλλέγουμε παραπάνω πληροφορίες από ό,τι είναι απαραίτητο. Το νομό μας συμφέρον ε, είναι αυτά πρέπει να κάνουμε για να παρέχουμε την ε, υπηρεσία στους χρήστες. Κομμάτι αυτών είναι η δραστηριότητα που υποχρεούμαστε εμείς να διαθέτουμε, να διασφαλίζουμε ότι είναι διαθέσιμη υπηρεσία. Ε, ναι, εντάξει, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά τα δεδομένα που παίρνουν τρίτα μέρη, αλλά πιστεύουμε και βάσει το δράσμα του Μαξ και άλλων αυτό θα δοκιμαστεί, πιστεύουμε από τώρα ότι πρέπει και συμφωνεί με το GDPR να βάλουμε μαζί τις ε, λειτουργίες ε, του κοινωνικού δικτύου, και τη δυνατότητα να παρέχονται, να διατίθεται αυτό το ε, ε μέσο κοινωνική δικτύωση σε ανθρώπου. Τελειώνει σιγά σιγά αυτό το απόγευμα στο οποίο κάναμε εκτενεί συζητήσει. Ε, θέλω να σα ευχαριστήσω όλου που ακολουθήσατε του κανόνε, που ήσασταν τόσο πειθαρχημένοι. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω και του δερμηνεί και να σα διαβεβαιώσω ότι πραγματικά εκτιμάμε τη δουλειά σας και είμαστε με το πλευρό σας. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο στις 2 Ιουλίου. Κύριος Κίνγκ, κυρία Γιώροβα, κύριος και Άντσιπ και ο κύριος Τίμερμανς και Φερστάγκερ Φεστάγκερ ακόμα περιμένουμε την απάντηση αλλά Ξέρουμε ότι θα έρθουν γιατί ε, είναι σημαντικό θέμα η στήριξη της νομοθεσίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και επίσης περιμένω και κάποιους άλλους ε, προσκεκλημένους ε, που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιώσει. αλλά είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους στην Επιτροπή μας. Επόμενη λοιπόν ακρόαση 2 Ιουλίου στο Στρασβούργο για τα μέλη της ΛΥΜΠΕ. Θα έχουμε και 28 Ιουνίου μια συνεδρίαση, δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Και μετά θα έχουμε 2, 9 και 10 Ιουλίου τις προγραμματισμένες μας συνεδριάσεις Στρασβούργο και Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα στις συνεδρίασεις. Καλό σας βράδυ.